So can the political advisor me tell if the members will come? It is now three minutes after half. Λοιπόν, καλησπέρα. Βλέπω λίγα μέλη, πολύ λίγα. Ένα εδώ, ένα εκεί. Τι συμβαίνει, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, κανονικά εγώ δεν πρέπει να περιμένω. Ίσως να, να περιμένουμε δύο λεπτά. Λοιπόν, υποσχέθηκα ότι θα αρχίσουμε και πέντε πέρα στο πεντάλεπτο και αρχίζουμε με, από το θέμα 20 της ημερήσιας διάταξης ανταλλαγή απόψεων για την εφαρμογή του Συμφώνου για συνεχείς βελτιώσεις με το Μπαγκλαντές. Ε, λοιπόν, αυτό αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας Γενικευμένων Προτιμήσεων και αφορά ειδικά την περίπτωση του Μπαγκλατές που είναι ε, μεγάλος ε, ε, αποδέκτης των γενικευμένων προτιμήσεων, το 66% των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή, εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 49 λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες που έρχονται από τον Μπαγκλατές. Άρα το Μπαγκλατές πραγματικά χρησιμοποιεί αυτό το πλεονέκτημα. Παρά τα αυτά, είχαμε και την ε, περίπτωση του Αναπλάζα το 2013 του Αναπλάζα και κοιτάξαμε το κείμενο πάρα πολύ προσεκτικά ε, βαθμολογήσαμε το σύμφωνο συνεχούς βελτίωσης ε, μελετώντας την υλοποίηση των υποχρεώσεων των γενικευμένων προτιμήσεων στο μπανγκλα ε, παρακολουθούμε από εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία. Κάναμε διάφορες συζητήσεις στην Επιτροπή, αλλά και στην ε, ομάδα παρακολούθησης ε, ε, Νότιας Ασίας και στείλαμε αντιπροσωπεία στο Μπαγκλατές το Νοέμβρη του 16 αν δεν κάνω λάθος. Οπότε ήρθε η στιγμή να γίνει συζήτηση. Ήθελα να πω, λέει το μέλος, ότι έχουμε διακεκριμένους εκπροσώπους του Μπαγκλαντές στην αίθουσα. Λόγω του ότι δεν είναι και τόσοι πολλοί οι συνάδελφοι, να τους δώσουμε λίγο χρόνο ή λίγο περισσότερο χρόνο από ότι τους είχε αρχικά δοθεί για να σχολιάσουν όχι είναι η απάντηση, διότι η εμπειρία από την μακρά συμμετοχή στο Κοινοβούλιο είναι ότι αν ξεκινήσουμε μια τέτοια διαδικασία χορηγώντας περισσότερο χρόνο ευθύς εξ αρχής τότε ο χρόνος δεν θα είναι η έναρξη και μισή, θα είναι παρα 25, θα είναι παρατέταρτο, ίσως και τρεις. Άρα θα ακολουθήσουμε την διαδικασία ανάλογα με τις εμφανίσεις στην Επιτροπή. Έτσι λοιπόν, παρότι είμαι ανοιχτό στις προτάσεις σας, στην περίπτωση αυτή δυστυχώς όχι. Οπότε, είναι κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς έχουν τα πράγματα δεδομένου ότι η ανανέωση του Ακόρτ ε, ως μια συνολική προσπάθεια έχει τεθεί στην ημερήσια διάταξη και η ειδική, η έκθεση των ειδικών του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας έχει ήδη φτάσει. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε τις μελλοντικές εξελίξεις και προοπτικές και όπως ε, ακούσατε και από τον συνάδελφο, έχουμε διακεκριμένους προσκεκλημένου, Είναι ο πρέσβης του Μπαγκλατές. Καλώς ορίσατε. Η κυρία Κάρεν Κέρτις, αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Προτύπων, Norms Department του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Η κυρία Τζένι Χολτκρόφτ, βοηθός Γενική Γραμματέας ε, του ε, Σωματείου των Industry All και ο δόκτωρ Πιέρ Γκρόνικ, ε, διευθυντής ε, του ΑΜΦΟΡΗ, που στο παρελθόν ήταν ε, η Ένωση Εξωτερικού Εμπορίου. Καλώς ορίσατε όλοι. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας για πέντε λεπτά για να μας παρουσιάσει την κατάσταση επιτόπου στο Μπαγκλαντές. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι τιμή που για το Διεθνέ Γραφείο Εργασία που βρίσκεται σήμερα εδώ να πάρει τον λόγο. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Το Διεθνέ Γραφείο Εργασία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν εταίροι στην στήριξη του συμφώνου αυτό, συνεχού βελτίωση και ε, βοηθήσαμε την κυβέρνηση του Μαγκλατέ σε διάφορου τομεί, συμπεριλαμβανομένων και των θέμων τη ε, επιθεώρηση εργασίας, τη βελτίωση συνθήκων ασφάλειας και υγείας και την προστασία των δικαιωμάτων. Η δέσμευση του Διεθνού Γραφείου Εργασίας με την κυβέρνηση του Μπαγκλαντέ ήταν σημαντική εκεί επί τόπου. Υπήρξε ένα σημαντικό πρόγραμμα τεχνικής συνεργασίας και ένα τακτικό σύστημα παρακολούθησης που πραγματοποιείται μέσω ειδικών μηχανισμών και που διευκολύνθηκε από την κύρωση από πλευρά του Μπαγκλαντές από τις 7 των συμβάσεις του ΑΚΟΡΤ και την ε, Συμβάση Εργασίας. Ήθελα να μας ενημερώσω όλους ε, για τις εξελίξεις του στο τελευταίο έτος όσον αφορά τα σχόλια των ε, οργάνων ε, παρακολούθησης. Ξέρουμε ότι το Μπαγκλαντές έχει εμφανιστεί στην ε, αρμόδια επιτροπή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για την εφαρμογή των ε, προτύπων επανειλημμένος τα τελευταία χρόνια και σε σχέση με την εφαρμογή της αρχής του συνέρχεστε και συνεταιρίζεστε και με, τα θέματα, εργασιακά θέματα. Στα τελευταία συμπεράσματα της Επιτροπής Εφαρμογής των Προτύπων έγιναν κάποιες συστάσεις και τέθηκαν κάποια θέματα προς την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές. Η Επιτροπή σημείωσε τη μακρά, ε, τη μακρά διάρκεια των θεμάτων που πρέπει να επιληθούν στο Μπαγκλαντές, κυρίως σε σχέση με τη σύμβαση του συνέρχεστε και Συνεθερίζεστε και τις προηγούμενες συζητήσεις που είχαν γίνει στην Επιτροπή. Και το γεγονός ότι δεν ήταν επαρκής η πρόοδο και βεβαίως έπρεπε να γίνουν περισσότερα άμεσα. Πιο συγκεκριμένα η εφαρμογή ε, των προτύπων ασχολήθηκε με την ανάγκη της, του νομοθετικής, εφαρμογής της νομοθετικής πράξης και νόμων για τις, ε, στις ζώνες επεξεργασίας ε, εξαγωγών σε σχέση με την ευθερία του συνέρχεστε και συντηρίζεστε και την αντιμετώπιση των διακρίσεων για να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση ανθρώπων που είχαν ε, ε, ε, απολυθεί παράνομα και την επιβολή προστήμων. Τελικά η Επιτροπή ζήτησε από την κυβέρνηση να εξασφαλίσει ότι οι αιτήσει εγγραφής θα διεκπεραιώνονται γρήγορα. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που συνεδρίασε πέρυσι, τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη, επανεξέτασε όχι μόνο τα θέματα αυτά, αλλά και άλλα θέματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης για την Επιθεώρηση Εργασίας. Και πιο συγκεκριμένα η έκθεση που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο εδώ και δύο εβδομάδες εκεί η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων σε σχέση με την ευκαιρία συνέρχεση και συνεταιρίζεστε χαιρετίζει κάποιες προτάσεις της κυβέρνησης για τροποποίηση του εργατικού νόμου του Μπαγκλατές και την εισαγωγή τυποποιημένων διαδικασιών ε, που θεσπίστηκαν σε σχέση με την εγγραφή στα εργατικά σωματεία που έχουν κάπως περιορίσει το χρόνο που αναμένεται για την εγγραφή αυτή όπως επίσης και τις αθέμητες εργασιακές πρακτικές όπω όπως επίσης και τις ιστοσελίδες που εισήχθησαν στο, ε, στο, ε, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας. Επίσης ε, σημείωσαν την ύπαρξη τριμερούς επιτροπής διαβούλευσης Παρά τα αυτά, σημείωσαν με ανησυχία ότι γίνονται νέα παράπονα για την ε, παρακράτηση, ε, σύλληψη και βία κατά των εργαζομένων και υπήρχαν πολλές εγγραφές ε, της εγγραφής που είχαν απορριφθεί. Αν δει κανεί την ιστοσελίδα του, του Υπουργείου Εργασίας, πολλές απορρίφθηκαν γιατί ε, τα σωματεία δεν είχαν καταφέρει να ε, συγκεντρώσουν το 30% συμμετοχής που απαιτείται για την εγγραφή. Και αυτό ενδεχομένως να εξηγεί το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν απάντησε εξίσου ενθουσιοδός στην πρόταση της κυβέρνησης να μειωθεί σταδιακά το απαραίτητο ποσοστό για την εγγραφή ε, των σωματείων στα διάφορα επίπεδα ανάλογα με τις επιχειρήσεις. Το 30% εξακολουθεί να παραμένει η απέτηση μέχρι 2.000 ε, εργαζομένους ενώ μέχρι πρόσφατα η έκθεση του ILO έλεγε ότι το 69% των επιχειρήσεων απασχολούν κάτω από 1.000 εργαζόμενους. Άρα οι εμπειρογνώμονες ανησυχούν ότι η προτινόμενη ε, μείωση ε, ελάχιστα θα επηρεάσει ε, την πλειοψηφία των επιχειρήσεων και άρα δεν θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην δημιουργία ελευθερίας, στην πρόθεση ελευθερίας που συνέρχεστε. Τώρα, όσον αφορά τις, τις ειδικές ζώνες επεξεργασίας, η Επιτροπή χαιρετίζει την προσπάθεια των αρχών να ευθυγραμμιστεί ο νόμος περισσότερο με τη σύμβαση αλλά υπογραμμίζει ότι πολλά θέματα εξακολουθούν να πρέπει να λυθούν και υπογραμμίζει την ανάγκη ότι οι ενώσεις μπορούν να βρουν μέλη εκτός των ζωνών αυτών και να συνεργαστούν με παράγοντες εκτός. Αυτά όσον αφορά τη, τη, Σύμβαση 87, την ελευθερία Συνέρχηση και συνεταιρίζεστε, αναμένεται ότι η οι αρχές εξακολουθεί να, ε, ε, εκεί εξακολουθεί να ισχύει η, δικαιοδοσία που προβλέπεται στο Μπαγκλαντές. Κατόπιν αυτού, ολοκλήρωσα τα πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ και είμαι ανοιχτή να απαντήσω σε ερωτήσεις. Πάρα... Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επισκόπηση από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο των συνδικάτων, από το Συνδικάτο Industry All, μέλος και της EG Metal. Σας καλωσορίζουμε κυρία Χολτκρόφτ και σας δίνουμε το λόγο. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω στην Επιτροπή. Είμαι βοηθός Γενικός Γραμματέας του All και επίσης μέλος της ε, Διευθύνουσα Επιτροπή για το ΑΚΟΡ, τη συμφωνία αυτή του Μπαγκλαντές. Έχουμε 20 συνδεδεμένα συνδικάτα στο ε, Μπαγκλαντές, μέλη και 15 από αυτά εργοποιούνται στον τομέα τη ένδυση. Θα σας ενημερώσω για το πώς έχουν τα πράγματα επιτόπου και ποια είναι η καθημερινή ε, εμπειρία των συνδικάτων. Όντως, ε, δεν έχει αλλάξει το κλίμα ως προς τον εκφοβισμό, την απειλή, τη βία κατά των συνδικαλιστών. Είχαμε πρόσφατο επεισόδιο στις 14 Φεβρουαρίου όταν τρεις οργανωτές από το SGSF ε, μέλος μας ε, μιλούσαν με εργαζόμενους στο εργοστάσιο όταν ο προϊστάμενος βγήκε προσπάθησε να τους βγάλει έξω από τα γραφεία και όταν αρνήθηκαν να πάνε μαζί τους οι εργοδότες, τους ξυλοφόρτω, οι οργανωτές συγγνώμη, τους ξυλοφόρτωσαν. Αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεν έχει αλλάξει τίποτα και οι μηνύσεις ε, χρησιμοποιούνται ως μέσο εκφοβισμού κατά των συνδικαλιστών. Θα θυμάστε ότι κάποιες μηνύσεις που έγιναν με κατηγορίες σε κάποια επεισόδια στην Ασούλια πριν από 12 περίπου μήνες. Πολλέ τέτοιες ε, ε, μηνύσει δεν έχουν ακόμη αποσυρθεί, εκκρεμωδικούν ε, οι υποθέσεις και υπάρχουν κάποιες παλιότερες υποθέσεις πριν από μία διετία όπου συνελήφθησαν εργαζόμενοι με αφίβολες κατηγορίες και παρά την ε, μη ε, διεξαγωγή δίκης ε, παρέμειναν σε προσωρινή κράτηση και μάλιστα όταν κλειδεύονται από το δικαστήριο χάνουν το ημερομίσθιό τους. Οπότε δεν είχαμε μεγάλη βελτίωση. Πάντως είχαμε ένα συνδικάτο στην Καζαπούρ που έκλεισε χθες από τις αρμόδιες αρχές μετά τις αναταραχές που έγιναν και τα επεισόδια για τους ε, χαμηλούς μισθούς και ακόμη δεν έχει επιτραπεί η επαναλειτουργία του από την τοπική αρχή και την αστυνομία. Σε ό,τι αφορά την εγγραφή των συνδικάτων, παρά την εισαγωγή των πρότυπων επιχειρησιακών διαδικασιών και πάλι είναι ιδιαίτερα επαχθής η διαδικασία για την εγγραφή των συνδικάτων στα εργοστάσια. Το βάρος απόδειξης που φέρουν τα συνδικάτα, κυρίως γύρω από τον κατάλογο των εργαζομένων, ονοματεπώνυμα, ταυτότητες, οικογενειακές σχέσεις, αυτή η κατάλογη και η σύνταξή τους είναι υπερβολικά επαχθής και είναι δύσκολο να διορθωθούν κάποιε ανακρίβειε στον κατάλογο. Ακόμη και αν ένα συνδικάτο καταφέρει τελικά να συγκεντρώσει τι υπογραφέ και τι πληροφορίε που χρειάζεται για να αποδείξει ότι 30% των εργαζομένων σε ένα εργοστάσιο θέλουν να προσχωρήσουν στο συνδικάτο, που και αυτό είναι πολύ δύσκολο, πολλέ φορέ τα εργοστάσια δίνουν διαφορετικού καταλόγου με εργαζομένου, πολύ πιο διευρυμένου στις αρχές καταχώρησης, οπότε η αρχή καταχώρησης απορρίπτει την αίτηση εγγραφή στο συνδικάτο γιατί δεν υπάρχει αντιστοιχεία των καταλόγων και αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο. Γενικώ πιστεύουμε ότι το κλίμα στο οποίο λειτουργούν τα συνδικάτα στον Παγκλαντέ δεν έχει δυστυχώς αλλάξει και τα εμπόδια στην ελευθερία του συνεταιρίζεστε εξακολουθούν να ισχύουν δυστυχώ. Ένα άλλο θέμα στο οποίο θα ήθελα πιστήσω την προσοχή σα είναι η έλλειψη πρόοδου σε ό,τι αφορά του ε, μισθού των υπαλλήλων σε εργοστάσια τη ε, ένδυση και το θέμα τη προστασία. Είπαμε ότι θα συστηθεί ένα συμβούλιο για τους μισθούς, αλλά αυτό συνέρχεται μία φορά την πενταετία και έχουν τους χαμηλότερους μισθούς του κόσμου σχεδόν στον Μπαγκλαντές ε, οι εργαζόμενες εργοστάσια ένδυσης και ο ρυθμός ε, αναβάθμισής τους, αύξησής τους είναι απελπιστικός. Και μάλιστα παρόλο που υποτίθεται ότι οι εργαζόμενοι θα συμμετείχαν στο συμβουλευτικό αυτό όργανο, τα συνδικάτα δεν έχουν κληθεί να λάβουν μέρος ε, στο, στο Συμβούλιο για τους μισθούς. Πάντως, ε, ε, η αντίδραση της κυβέρνησης του Μπαγκλαντές για το ΑΚΟΡΤ και τη συμμετοχή κάποιων συνδικάτων είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα, γίνει, δεν θα συνεχιστεί το ΑΚΟΡΤ αυτή η συμφωνία. Τελικά, ε, αν δεν είναι έτοιμο το πρόγραμμα της κυβέρνησης για να συνεχίσει να διαδεχθεί το ΑΚΟΡΤ, τελικά θα γίνεται επιτήρηση παρακολούθηση του ΑΚΟΡΤ σε εξάμεινη βάση και ε, υπάρχουν αμφιβολίες ε, για το αν θα συμφωνήσουν τα συμβαλόμενα μέρη, δηλαδή εργοδότες ε, και συνδικάτα και επίσης δεν υπάρχει συμφωνία για το ποια θα είναι τα κριτήρια ή το κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις από το κυβερνητικό πρόγραμμα. Πάντως, από ό,τι μας λέει το, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, μέχρι στιγμής το κυβερνητικό πρόγραμμα δεν είναι έτοιμο για να διαδεχθεί πλήρως τη συμφωνία αυτή το ΑΚΟΡΤ και ελπίζουμε να συνεχιστεί τελικά μέχρι ότου είναι όριμο το κυβερνητικό πρόγραμμα για να αναλάβει τη διαδοχή. Επίση, θέλουμε να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα κριτήρια και σωστέ αξιολογήσει. Επίση μα προβληματίζει το πώ το κυβερνητικό πρόγραμμα θα ολοκληρώσει τι διαδικασίε διατησία σε εργοστάσια που δεν καλύπτονται από το ακόρντο ούτε από τη συμμαχία μετά από τις πιέσεις που ασκούνται από τα διεθνή εμπορικά σήματα, τις διεθνείς μάρκες Γι' αυτό για να σας εξηγήσω ότι εξακολουθούμε να έχουμε αμφιβολίες και σίγουρα δεν συντρέχουν ακόμη οι προϋποθέσεις του Συμφώνου Βιωσιμότητας που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον Μπαγκλαντές. Οπότε καλό θα ήταν στα πλαίσια του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων να γίνει μια έρευνα για μη συμμόρφωση εκ μέρους του Μπαγκλαντές. Σας ευχαριστούμε. Έχουμε Χολτ, ε, ένα νέο ε, ε, ακρονίμιο από το αμφόρι, αν δεν κάνω λάθος. Θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο. Το αμφόρι δεν είναι ακρονίμιο. Το αμφόρε... Α, είναι η αμφορά. Ο αμφορές μάλλον, αμφορές που χρειαζόταν και χρησιμοποιεί κατά το παρελθόν ε, για τη μεταφορά πραγμάτων. Εμείς ε, χρησιμοποίησαμε αυτή την ονομασία για τη δική μας την Ένωση που εκπροσωπεί περίπου 2.000 ε, εισαγωγείς με ετήσιο κύκλο εργασιών 1,7 δισεκατομμύρια. Και όπως είπατε και εσείς, αλλάξαμε την ονομασία μας από Foreign Trade Association σε BSI και BPI και αμφόρε. Το Μπαγκλαντές λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για τα μέλη της δικής μας της Ένωσης. Μετά την Κίνα και την Ινδία, το Μπαγκλαντές είναι η τρίτη χώρα από την οποία εισάγουμε προϊόντα. Περίπου 7% είναι ε, το εισαγωγές ε, του συνόλου όγκου των εισαγωγών μας από το Μπαγκλαντές. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τη χώρα αυτή. Τα τελευταία πέντε χρόνια μετά τα τραγικά γεγονότα στη Ράνα Πλάζα, ε, περίπου που 6.000 καταγγελίες κατέφτασαν σε εμά. Προσπαθήσαμε να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα. Όσον αφορά το ακόρ τη συμφωνία αυτή, επιτρέψτε μου να αναφέρω τρία πράγματα. Πρώτον, η συμφωνία αυτή του ΑΚΟΡ θεωρούμε ότι ήταν επιτυχία. Η ουσιαστική συμμετοχή επιχειρήσεων από την Ευρώπη, από κοινού μαζί με συνδικάτα, καταδεικνύει με απόλυτη σαφήνεια ότι οι εισαγωγεί ε, επιθυμούν να αναλάβουν τι ευθύνε του. Ε, περίπου το 45% των μελών του ΑΚΟΡ βρίσκονται αυτή τη στιγμή οργανωμένοι, είναι μέλη και τη ε, δική μα τη Ένωση. Τα διορθωτικά μέτρα εφαρμόζονται κατά πάνω από 80% ικανοποιητικό αυτό και αν έχει κανεί κατά νου το 90% που είναι ο στόχος, ε, μάλλον θα το πετύχουμε. Η χώρα έχει κάνει άλμα όσον αφορά την προστασία, πυροπροστασία κυρίω ε, των κτηρίων και νομίζω ότι έχουν μειωθεί κατά πολύ τα ατυχήματα, βεβαίω δεν αποκλείονται πλήρω. Και για τον λόγο αυτό οφείλουμε να αποτίσουμε φόρο τιμή στο θέμα αυτό στο Μπαγκλαντές. Ε, το ΑΚΟΡ, η συμφωνία μπορεί να επιβάλλει μέτρα μετά από αποφάσεις ε, διαιτητικού δικαστηρίου. Συνέβη αυτό συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο ε, και ο θυγόμενος είπε ότι θα καταβάλει το πρόστιμο. Άρα δηλαδή βλέπετε ότι το ακόρ μπορεί να είναι και ουσιαστικό. Κατά τα άλλα θέλω να σας πω ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες. Γι' αυτό λοιπόν περνάω στο δεύτερο θέμα, στη νέα συμφωνία με νέους φιλόδοξους στόχους, διευρυμένη μερίσια διάταξη. Πλήρης μεταφορά της ε, ευθύνη στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντές. Αυτό δεν θα ήταν σωστό γιατί δεν θα μπορούσε να εγγυάται συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τη διεύρυνση της εντολής τη θεωρούμε πολύ σημαντική γιατί ε, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα με την ελευθερία του συνεταιρίζεστε, με πολλές άλλες ελευθερίες. Αυτό το υπενήχθησαν και οι προλαλήσαντες. Τα μέλη της δικής μας της Ένωσης έχουν ε, αναφερθεί επανειλημμένα στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντές έτσι ώστε να μεταρρυθμιστεί το εργασιακό δίκαιο και να διασφαλίζονται κάποιες ελευθερίες. Ε, στο θέμα αυτό θα επιμείνουμε και μεταξύ άλλων προγραμματίζουμε για τον Απρίλιο μια νέα, ένα νέο γύρο συζητήσεων στην ίδια την ΤΑΚΑ. Ε, όσον αφορά τον αριθμό εκείνων που υπογράφουν το ΑΚΟΡ, έχει μειωθεί βέβαια ο αριθμός τους και αυτό δεν οφείλεται στο ότι δεν ενδιαφέρονται, αλλά οφείλεται στο ότι ε, για να υπογράψει κανείς σημαίνει ότι δέχεται και κάποιες νομικές λεπτομέρειες όπως και τον συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο θα γίνεται χρηματοδίτης κατά τη διάρκεια ανακαινήσεων που προβλέπονται στη συμφωνία στο ΑΚΟΡ. Όσον αφορά τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, αυτό είναι σημαντικό. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν αναλαμβάνουν επιχειρηματικό κίνδυνο, κυρίως για μονάδες παραγωγής, επί των οποίων δεν έχουν κανένα απολύτως έλεγχο. Οι επιχειρήσεις βέβαια αριθμός τους σίγουρα θα αυξηθεί ε, μέχρι το τέλος Μαΐου που θα υπογράψουν δηλαδή το ακόρ Μέχρι τώρα έχουμε άλλους 53 που έχουν υπογράψει που σημαίνει ότι έχουμε ξεπεράσει το στόχο μας ε, που είχαμε θέσει για το τρέχον ΑΚΟΡ, την τρέχουσα συμφωνία. Τρίτος βασικός μας ε, στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προποθέσει έτσι ώστε η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και οι επιχειρήσεις που έχουν υπογράψει το ΑΚΟΡ να μπορούν να επιδιώξουν τους στόχους με δική τους ευθύνη. Οι ε, κατά την άποψή μας ε, μπορούν να επιτευχθούν μόνο εφόσον στηρίζονται και από το εσωτερικό της χώρας. Η εξωτερική ανάθεση διοικητικών διαδικασιών σε ξένες επιχειρήσεις κατά την άποψή μου ε, αυτό δεν είναι αποτελεσματικός τρόπος, δεν είναι βιώσιμος. Ε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω και τελειώνω ότι εμείς δεν θα αποσυρθούμε από τον Μπαγκλαντές ακόμα και αν κάποια ε, στιγμή επιτευθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Εμείς θα συνεχίσουμε να επιμένουμε. Έχουμε κατά νου μία σειρά προγραμμάτων, παραδείγματος ένα πρόγραμμα το οποίο εκπνέει τον Απρίλιο, διήρκησε για τρία χρόνια και αυτό ήταν είναι πολύ σημαντικό για μας. Σε γενικές γραμμές θεωρούμε ότι το Μπαγκλαντές βρίσκεται σε σωστό δρόμο. Βεβαίως και υπολείπονται ακόμα πολλές βελτιώσεις. Ε, πρέπει να ληφθούν ακόμα συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε ευγνώμονες για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Κοινοβούλιο επιλαμβάνονται τις υπόθεσεις του Μπαγκλαντές και να ξέρετε ότι εμείς είμαστε ένας εταίρος σας και συνεργάτης στην προσπάθεια αυτή. Και τώρα για σύντομη παρέμβαση ο πρέσβης του Μπαγκλαντές, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εξοχότητες κυρίες και κύριοι. Σας είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνετε να έρθω και να σας παρουσιάσω τις απόψεις μας για την εφαρμογή του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπαγκλαντές. Και όταν μιλούμε για το Σύμφωνο Βιωσιμότητας δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι το Μπαγκλαντές ε, διανύει μια πολύ σοβαρή κρίση που μας κληροδότησε η γείτονα χώρα στέλνοντας μεγάλους αριθμούς πρόσφυγες ροχίνγκια και με τους ελάχιστους πόρους που έχουμε προσπαθούμε να δώσουμε καταφύγιο σε ένα περίπου εκατομμύριο ροχίνγκιας. Οπότε αυτό μην το ξεχνάτε όσο συζητάμε την κατάσταση εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας των Μπαγκλαντές. Το Μπαγκλαντές ε, είναι ευγνώμων και αναγνωρίζει την υποστήριξη ε, και αρρωγή των εταίρων ε, του Συμφώνου ώστε να γίνουν τα εργοστάσια των Μπαγκλαντές ασφαλέστερα. Τώρα, τα Εργοστάσια ένδυσης ε, με την έναρξη του Συμφώνου Βιωσιμότητας έχουν ε, περάσει από αυστηρούς ελέγχους και επιθεωρήσεις, έχουν γίνει πολλές επιδιορθώσεις ε, και ανακατασκευές και μάλιστα ως εργοστάσια δεν πληρούν τους όρους του συμφώνου απομακρύθηκαν, αφαιρέθηκαν από τον κατάλογο των δικαιούχων εξαγωγών. Οπότε δεν έχουμε πια μόνο ασφαλή εργοστάσια ενδυμάτων, αλλά έχουμε και το πιο εξυγχρονισμένο σύστημα και φιλοπαρε... φιλοπεριβαλλοντικό σύστημα εργοστασίων ένδυσης των Μπαγκλαντές. Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες που τις έχει αναγνωρίσει και η διεθνής κοινότητα και οι εταίροι μας ότι η ασφάλεια και προστασία στον τομέα ένδυσης έχει εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό. Και ένα μεγάλο τμήμα των κονδυλίων έχει επενδυθεί ακριβώς σε αυτό το θέμα. Οι προλαλήσαντες μίλησαν για την τριμερή συμβουλευτική επιτροπή και τα συναφή. Δεν θα επεκταθώ λοιπόν σε αυτό. Εγώ θα ήθελα α, κυρίως να κάνω το καθήκον μου και επιτρέψτε μου να μιλήσω λίγο περισσότερο από ό,τι δικαιούμαι, γιατί θα ήταν άδικο να περιοριστώ μόνο σε λίγα σημεία. Θα βάλω πάντως τα δυνατά μου να μην μακρηγορήσω. Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την Ακόρτ και τους φίλους μας από τα συνδικάτα και κυρίως από το συνδικάτο Uniglobal και το Industry All για την σχολαστική διενέργεια των επιθεωρήσεων ε, των εργοστασίων. Πραγματικά τους συγχαίρομαι για το έργο τους που είναι πολύ αξιόλογο. Και ε, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας επιτελεί ένα αξιέπαινο έργο στο Μπαγκλαντές. Και ε, η ύψη προτεραιότητα της κυβέρνησης του Μπαγκλαντές είναι η ευημερία των πολιτών της. Και γι' αυτό ε, αναμειγνύουμε και μπλέκουμε όλους τους κοινωνικούς εταίρους και τους ενδιαφερομένους στην προσπάθεια τροποποίησης του εργατικού νόμου του Μπαγκλαντές και τη σύσταση της Τριμερούς Επιτροπής, προκειμένου να λάβουμε υπόψη τις συστάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και να πραγματοποιήσουμε τις απαραίτητες αλλαγές στο εργατικό νόμο. Μάλιστα, ο εργατικός νόμος ε, προηγούμενος είχε πάλι τροποποιηθεί χάρη στι συστάσει και λαμβάνοντας υπόψη συστάσεις του ΔΟΕ με το νέο εργατικό νόμο ε, οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και εργαζομένων ε, εκπροσωπούνται ισότιμα με τους ε, κυβερνητικούς εκπροσώπους και κάθε μέλος της Τριμερούς Επιτροπής εκφράζει τις απόψεις του και κάνει συστάσεις. Κάτι τέτοιο θα αποβεί προ όφελο των εργαζομένων του Μπαγκλαντές, λαμβάνοντας υπόψη και την κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα της χώρας. Από την διαμόρφωση του Συμφώνου Βιωσιμότητας, η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και το Υπουργείο Εργασίας και Απασχόλησης έκαναν πολλά σημαντικά βήματα για την εφαρμογή του Συμφώνου Βιωσιμότητας και θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Οι πρόσφατες εξελίξεις των πρότυπων επιχειρησιακών διαδικασιών SOP που αναφέρουν και οι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεύτερον, η δημοσιότητα και πρόσβαση των επιγραμμικών βάσεων δεδομένων σε όλα τα συνδικάτα, προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερε εργασιακέ σχέσει. Τρίτον, αισθητή αύξηση του προπολογισμού και των ανθρώπινων πόρων, προκειμένου να γίνουν οι επιθεωρήσει των εργοστασίων με αυξημένο δυναμικό. Τέταρτον, ε, η το εργατικό νόμο και ο εργατικό νόμο για την ζώνη μεταποίηση προ εξαγωγή ακολουθούν τι συστάσει του ΔΟΕ και οι σχετικέ τροποποιήσει τη νομοθεσία θα εγκριθούν όσον όπα από το Κοινοβούλιο. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να υπάρχει διάσταση απόψεων για το ποιο θα πρέπει να είναι το κατόφλι για την σύσταση συνδικάτων στα εργοστάσια και ποιο θα έπρεπε είναι το ποστό συμμετοχή. Αλλά στη στενή συνεργασία με του φίλου και εταίρου ε, συνεχίζουμε τι συζητήσει και θα ήθελα εγκατακλείδη να πω ότι η, η συνεργασία που έχει ξεκινήσει μετά το Σύμφωνο Βιωσιμότητας έχει δημιουργήσει μια μεγάλη όθηση και δυναμικό. Θα το αξιοποιήσουμε για να έχουμε μεγαλύτερη επιτυχία. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω τώρα να ε, ε, καλωσορίσω μια ομάδα φοιτητών πολιτικών επιστημών από το Παρίσι, νομίζω. Ορίστε, καλώς ορίσατε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Κάρη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μόλις επέστρεψα από τον Μπαγκλατές, όπως γνωρίζετε, η περασμένη εβδομάδα ήταν πράσινη εβδομάδα και συνόδευσα την αντιπροσωπεία Νότιας Ασίας του Κοινοβουλίου στα πλαίσια ε, μιας υποεπιτροπής της Επιτροπής μας. Μου έδωσαν πολύ εκτεταμένες ε, σημειώσεις για την ομιλία μου. Δεν σκοπεύω να επαναλάβω όσα είπαν οι προλαλήσαντες και θέλω να βοηθήσω, να ευχαριστήσω πολύ κάποιους από τους προσκεκλημένους που είπαν όσα είπαν. Θέλω όμως να πω δύο λόγια για τις προηγούμενες συναντήσεις μου που είναι σχετικά πρόσφατες την περασμένη εβδομάδα και άρα ε, ε, θα μας ενημερώσουν αρκετά. Πολλές από τις προκλήσεις τέθηκαν κυρίως σε σχέση με τα συνδικάτα και τη διαδικασία εγγραφής, και πρέπει να συμφωνηθεί ε, ακόμα η δημιουργία των συνδικάτων στις ειδικές ζώνες της ε, EPZ, της, EPZ, τις ζώνες μεταποίησης ε, προς εξαγωγή και μοιάζει ότι όπως έχουν τώρα τα πράγματα δεν έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση παρά το ότι πέρασε χρόνος. Θυμάμαι πολλά από τα επιχειρήματα που εξακολούθησαν σήμερα στο Μπαγκλαντές να μου τα προβάλλουν και τα οποία τα είχα ξανακούσει πριν από δύο χρόνια επί της ουσίας δεν είχε σημειωθεί παραμικρή πρόοδος στο, στον αφορά, στο τομέα των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ τον πρέσβη για τα όσα μας είπε, όμως θυμάμαι ότι πριν δύο χρόνια μου είπαν ότι πρέπει να προσλάβουμε Περισσότερου επιθεωρητές για να γίνουν οι επιθεωρήσεις ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υλοποιηθούν οι νέε διατάξεις. Δύο χρόνια αργότερα εξακολουθώ να ακούω τα ίδια πράγματα. Άρα ε, ουσιαστικά υπάρχει ανάγκη όχι μόνο για δεσμεύσεις ότι θα γίνει πρόοδος, αλλά εν περιπτώσει να δούμε και την πρόοδο αυτή. Υπάρχουν όμως και τομείς στους οποίους σημειώθηκε πρόοδος και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε και όχι μόνο να το αναγνωρίσουμε αλλά και να δώσουμε περαιτέρω ενθάρρυνση. Πράγματι γνωρίζω τις πολύ πρόσφατες εξελίξεις που έχουν ε, βαρύνει ακόμα περισσότερο την κυβέρνηση αλλά και το λαό του Μπαγκλαντές, κυρίως μέσω της κρίσης των Ροχίντζα που έχει εξελιχθεί σε πολύ μεγάλες διαστάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα εμπορικό χώρο για το Μπαγκλατές αν είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε κάπως περισσότερο τη χώρα να αντιμετωπίσει με την άμεση αυτή εξέλιξη την κατάσταση που αντιμετωπίζει. Δεν ξέρω πώς θα το πετύχουμε, αλλά τόσοι έμπειροι συνάδελφοι στην αίθουσα θα έχουν προτάσεις. Έχω και εγώ κάποιες, μπορούμε όμως να το δούμε. Ένα από τα βασικά θέματα που προκύπτει ξανά και ξανά και εξανατέθηκε σήμερα προηγουμένως σε σχέση με τις γενικευμένες προτιμήσεις είναι και το θέμα του ότι και από πλευράς ε, των ε, εργοστασίων του Μπαγκλατές ε, οι οποίοι επιθυμούν να πετύχουν τα επιθυμητά τα πρότυπα, αλλά και αυτό είναι προϋπόθεση και για τη δική μας πλευρά. Υπάρχουν όμως πιέσεις όσον αφορά τις τιμές των παραγγελιών που δέχονται. Και εδώ υπάρχει ανισορροπία. Μου το έδειξαν απολύτως σαφές κατά την παραμονή μου εκεί. Πώς οι αγοραστές πηγαίνουν γνωρίζοντας ποια είναι η βασικότατη τιμή, η κατώτατη τιμή ε, για ένα προϊόν και προσπαθούν να ολοκληρώσουν, να πετύχουν μια ψηλότερη τιμή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχουν τα περιθώρια που να επιτρέπουν να εφαρμοστούν οι απαιτήσει που ισχύουν εδώ και που εμείς θέλουμε να ισχύουν. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανισορροπία η οποία πλέον έχει φτάσει στο σημείο που δεν είναι βιώσιμη η κατάσταση. Και αυτό θα δημιουργήσει πιέσεις, ιδίως σε θέματα εργασιακών δικαιωμάτων και αμοιβών. Κύριε Πρόεδρε, όμως και εμείς κάποια στιγμή πρέπει εμείς να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό απέναντι στους πολίτες μας. Γιατί οι πολίτες θέτουν πολύ σωστά τα θέματα αυτά, όχι μόνο για απέναντι στις εταιρείες από τις οποίες αγοράζουν, αλλά και στους εκλεγμένους εκπροσώπους τους. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει αποκλειστικά και μόνο η τιμή, αλλά πώς ε, παρήχθη, τι είδους αμοιβέ πληρώνονται γι' αυτό, ποιες είναι οι συνθήκες τις οποίες ζουν οι άνθρωποι αυτοί. Άρα πρέπει αυτό τον κύκλο να τον τετραγωνίσουμε κάποια στιγμή και, να, ε, ε, και ρωτάω την Επιτροπή κατευθείαν σήμερα. Τι είμαστε σε θέση, τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε για να ασχοληθούμε με το θέμα. Και το ερώτημα το απέφυγαν εντελώς. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Βλέπω ότι έχει το σφυρί, ξέρω τι θα κάνεις, δεν θέλω να σε έχω να αντιμετωπίσω με το ε, σφυρί και γι' αυτό θα σταματήσω και θα καθίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος, <laughs> πολύ καλά. Οπότε τώρα θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο, αλλά με ξεκάθαρο στους συναδέλφους. Πολύ συγκεκριμένα όμως ερωτήσεις προς τους ειδικού και την Επιτροπή. Και με συγκεκριμένο στόχο. Πείτε μας σε ποιον απευθύνεται η ερώτηση. Αγνές, είσαι πρώτη. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και εγώ βέβαια έχω σημειώσει πάρα πολλά όπως και ο συνάδελφός μου. Ε, πιστεύω ότι η κατάσταση είναι αρκετά σαφής πλέον μετά από αυτά που ακούσαμε. Ως εκ τούτου ε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφερθώ στο ιστορικό σε άλλα θέματα. Βέβαια είναι σαφές ότι η διεθνής κοινότητα έχει ζητήσει από την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές να εφαρμόσει ε, μια σαφή ε, υποχρέωση όσον αφορά θέματα υγείας και ασφάλειας ε, και πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί βεβαίως και χάρη της πίεσης που ασκήθηκε από τα συνδικάτα και από τους ε, παραγωγούς. Βεβαίως υπάρχει και μία σαφής σειρά δεσμεύσεων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τους ε, κανονισμούς ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Ε, η έκθεσή σας στην Επιτροπή νομίζω είναι σαφές ότι όσον αφορά τις τέσσερις υποχρώσεις, δεσμεύσεις δηλαδή μεταρρύθμιση του εργασιακού δικαίου, ε, των ε, ζώνων μεταποίησης προς εξαγωγή, τα συνδικάτα, ε, την κατάργηση των διακριτικών μεταχειρήσεων εις βάρος των συνδικάτων. Όσον αφορά αυτά τα θέματα δεν σημειώνεται καμία πρόοδος. Παρότι βέβαια το ερώτημα κατά πόσον αρκούν τα χρήματα για αξιοπρεπή ε, διαβίωση. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Εγώ θέλω να απευθυνθώ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι προηγουμένως ε, ακούσαμε δύο διαφορετικές ε, ημερομηνίες καταληκτικές ημερομηνίες. Κάποιοι είπαν ότι η μεταρρύθμιση του εργασιακού δικαίου θα πρέπει να γίνει πριν από τον Μάιο του 2017, μετά πήγε Αύγουστος του 2017 και Τώρα πλέον μιλάμε για το Φεβρουάριο και έχουμε αυτή την έκθεση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που η έκθεση αυτή για μας είναι σημαντική. Ε, ερωτώ λοιπόν, ή... θέλω να πω το εξής πριν παρέλθει κάποια συγκεκριμένη ε, καταληκτική ημερομηνία, νομίζω και εμείς θα πρέπει να είμαστε σοβαροί και να ξεκινήσουμε μία επίσημη έρευνα για το ερώτημα κατά πόσον η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές ε, εξακολ... της αξίζει να εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η γενικευμένη προτίμηση που υπάρχει προς την ίδια. Όχι ότι θέλουμε να άρουμε αυτή την προτίμηση, αλλά διότι να καταλάβουν όλοι ότι είμαστε σοβαροί και στις υποχρεώσεις μας και όσον αφορά στις καταληκτικές ημερομηνίες. Πολύ ωραία. Η Λούλα. Ευχαριστώ μετά την ανάγνωση της έκθεσης εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας ε, του Μπαγκλαντές και μετά από ανάγνωση εκθέσεων μη κυβερνητικών οργανώσεων ή συνδικάτων αλλά και μετά από τους καλεσμένους μας ε, θεωρούμε ότι ε, ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί οι στόχοι του Συμφώνου Βιωσιμότητας. Έχουμε το θέμα των συνδικάτων, των εργασιακών επιθεωρήσεων και την λήψη υπόψη των συστάσεων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Έγιναν πολλέ προσπάθειε στους πυλώνες που αφορούν τα εργασιακά δικαιώματα και την ασφάλεια των κτίριων και των εργοστασίων, αλλά ακόμη ε, παρασάγκα απέχουμε από, τα, ε, από την τήρηση των συμφωνιών, των συμβάσεων του διεθνού Γραφείου Εργασίας. Ε, θα πρέπει να ενταθούν εκεί οι προσπάθειε. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την υπεύθυνη στάση των επιχειρήσεων δεν θα πρέπει να υπάρχουν σχετικές συστάσεις και όχι μόνο για τη βελτίωση της στάσης αλλά και την υπευθυνότητα, την υπεύθυνη συμπεριφορά που θα πρέπει να, γίνουν, να, να δείχνουν οι επιχειρήσεις. Και οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα αξίας που περνάει και από τον Μπαγκλαντές θα πρέπει να είναι οι πρώτε ενδιαφερόμενε για την τήρηση των εργασιακών προτύπων και προδιαγραφών και τη βελτίωση τη κατάσταση. Γιατί δυστυχώ ε, η πείρα μα ε, δημιουργεί υπόνοιε για το κατά πόσο είναι ειλικρινεί οι επιχειρήσει. Ε, Επίση, οι επιχειρήσει που μεταθέτουν την παραγωγή τους στο Μπαγκλαντές θα πρέπει να λάβουν ξεκαθαρή θέση και να είμαστε κι εμείς κατηγορηματικοί ότι αν δεν τηρούνται οι οι προδιαγραφέ θα επιβάλλονται κυρώσει. Η συμφωνία και η συμμαχία, η Accord και η Alliance δηλαδή, ε, έχουν αρκετές ε, ελλείψεις στην εφαρμογή. Και μάλιστα υπάρχει κίνδυνος να έχουμε όλο και λιγότερα αποτελέσματα ή να έχουμε αποτελέσματα μόνο σε ορισμένους τομείς όπως είναι η ασφάλεια των κτίριων που το επισημάνουμε και το αναγνωρίσαμε αλλά ταυτόχρονα να μην έχουμε αξιοπρεπή εργασία και σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων στα εργοστάσια ενδυμάτων, γιατί αυτό είναι και θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων. Επίσης, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένω απευθύνε εκκλήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίω στην έκθεση ό,τι φορά την εμβληματική πρωτοβουλία για το ε, τομέα των κλωστιφαντουργίων, που ήδη έχει συμπληρώσει και ένα χρόνο ζωή. Νομίζω ότι θα πρέπει επιτέλου να δούμε αποτελέσματα αυτών των εκκλήσεων. Η Καρολίν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε ότι ε, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, αλλά εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει είναι ότι αν δεν τηρούνται διατάξεις, ε, τότε πώς λειτουργεί όλη η διαδικασία. Ο κύριος Πρέσβης είπε ότι αυτές οι επιχειρήσεις διαγράφονται από τον κατάλογο των εξαγωγιών ε, Ποιε είναι οι παραβάσεις που οδηγούν στο να αφαιρεθεί κανείς από τον κατάλογο και τι γίνεται μετά, ποια είναι η διαδικασία. Να υπογραμμίσω αυτά που είπε η Άγνες ε, και η Κομισιόν το είπε αυτό πέρυσι ότι θέλει να εξετάσει το θέμα να δει ε, κατά πόσον ε, το Μπαγκλαντές θα πρέπει να εξακολουθήσει να έχει τις γενικευμένες αυτές προτιμήσεις. Γνωρίζουμε ότι τα πράγματα υπολείπονται στην πρακτική εφαρμογή. Συγκεκριμένα η Κομισιόν τι προτίθεται να κάνει. Ευχαριστώ. Καταρχήν, να μην ξεχνάμε και το συνολικό πλαίσιο. Το Μπαγκλαντές ε, δεν είναι μια εύπορη χώρα ή μια χώρα με μεγάλο φυσικό πλούτο ή πολλού φυσικού πόρου και φαντάζομαι ο πρέσβη θα συμφωνεί. Οπότε αυτήν την άποψη ε, τα εργοστάσια ένδυση, η μια χωρα με μεγαλο φυσικο πλουτο η πολλους φυσικους πορους και φανταζομαι ο πρεσβης θα συμφωνει οποτε αυτην την αποψη τα εργοστασια ενδυσης η κροστιφαντουργια του μπαγκλαντες ήταν μια ε, μεγάλη επιτυχία για τη χώρα αυτή για παράδειγμα, δίνει άμεση απασχόληση σε 4 εκατομμύρια ανθρώπους ο τομέας ένδυσης. Ε, και 55% αυτών είναι γυναίκες, ε, έτσι λέει εδώ. Δεν το λέω εγώ, εδώ το λέει η έκθεση που έχω. Οπότε ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία για τη χώρα αυτή η άνθηση του τομέα ένδυση. Τώρα έχουμε δύο εκπροσώπου των συνδικάτων που έλαβαν το λόγο και του δώσαμε και αρκετό χρόνο να μιλήσουν. Είχαμε όμω και πολυάριθμου εκπροσώπου των κεντροαριστερών κομμάτων που ζήτησαν το λόγο και τον έλαβαν. Ε, και μην ξεχνάτε ότι στην Γερμανία μόνο το 18% του εργατικού δυναμικού συμμετέχει, είναι οργανωμένο σε συνδικάτα. Και νομίζω ότι πρόσωπο τη Διεθνού Οργάνωση Εργασία είχε μια αμερικανική προφορά. Στι Ηνωμένε Πολιτείε, λιγότερο από το 8% του εργατικού δυναμικού είναι οργανωμένο σε συνδικάτα στον ιδιωτικό τομέα. Οπότε ανακύπτει η ερώτηση, ή μάλλον όχι ερώτηση, αλλά μια σκέψη που θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σα. Κοιτάξτε, το Μπαγκλαντέ είναι μια χώρα που έχει πολλά εγγενή προβλήματα και ε, λόγω κλίματος και ε, λόγω άλλων αιτιών. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι μια εύπορη χώρα, δεν έχει φυσικό πλούτο. Και παρόλα αυτά η βιομηχανία της κατάφερε να ανθίσει τα τελευταία χρόνια. Έχει ενισχύσει και έχει χειραφετήσει ε, πάρα πολύ κόσμο και 55% του μεγάλου αριθμού απασχολουμένων είναι γυναίκες. Οπότε θέλουμε να επιβάλλουμε στη χώρα αυτή ε, όλα αυτά τα αρνητικά και συμπαραμαρτούνται τη υπερβολική νομοθεσία και γραφειοκρατία. Όχι. Κρίμα θα ήταν. Ναι, πολύ θα ήθελα να μάθω τι μορφή θα έχουν οι εμπορικέ συμφωνίε Ηνωμένου Βασιλείου και Μπαγκλαντέ στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να απευθυνθώ στους στον προλαλήσαντε και να το πω καλύτερα ε, να κάνουμε εδώ μία συζήτηση. Είναι σωστό να υπάρξει η συζήτηση. Μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μήπως ε, μπορείτε να τοποθετηθείτε στην ετήσια έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, γιατί θα ήθελα να έχω μία διεξοδική έκθεση ε, επί του θέματος. Αναφέρεται ότι το Μπαγκλαντές δεν έχει σημειώσει καμία απολύτως ε, ε, πρόοδο όσον αφορά τη βία κατά των συνδικάτων. Εξακολουθεί να υπάρχει εκφοβισμός εργαζομένων, βία κατά των εργαζομένων και ο εργασιακός νόμος εξακολουθεί να υπολείπεται κατά πολύ του αναμενόμενου. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να διεξάγουμε μια έρευνα επί του θέματος. Πρόεδρος, νομίζω ότι όλες οι ερωτήσεις ε, αφορούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε δύο εκπροσώπους από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, την Αλίνα Μπόιτσουκ, η οποία είναι ε, αναπληρώτρια διευθύντρια της μονάδας. Ε, δεν ξέρω ποιος θέλει να ξεκινήσει. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μας ε, δίνετε το λόγο. Μάλιστα, είναι αλήθεια πράγματι, τα περισσότερα ερωτήματα αφορούν την Κομισιόν. Όπως ξέρετε, ασχολούμεθα με τον Μπαγκλαντές εδώ και κάποια χρόνια και έχουμε ασκήσει πίεση στις αρχές του Μπαγκλαντές να ε, παρουσιάσουν συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα στη χώρα. Ε, συνεργαζόμαστε λοιπόν ε, στο πλαίσιο μιας εταιρικής σχέσης, όχι με την ανετής επιβολής ε, κυρώσεων. Γιατί, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι συνεργαζόμαστε με μια χώρα η οποία ε, κατατάσσεται στις χώρες με τις ε, ελάχιστα ανεπτυγμένες οικονομίες. Ε, πρέπει να τις στηρίξουμε. Οι οικονομίες αυτών των χωρών είναι ιδιαίτερα ευάλωτες και αυτό για μας είναι το σημείο εκκίνησης. Δηλαδή εταιρική σχέση και αυτή η μορφή συνεργασίας έναντι μιας πολύ ευάλωτης χώρας. Η συμφωνία ήταν να υπάρξει μια συμμαχία και με άλλες χώρες ε, που πρεσβεύουν το ίδιο και με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Διότι ε, το δεύτερο στοιχείο της συνεργασίας μας ε, είναι να στηρίζουμε και να σεβόμαστε τα εργασιακά δικαιώματα και αυτά που προβλέπει το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Εμείς σεβόμαστε το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, του υποβάλλουμε κάθε φορά τις απόψεις μας και τις πληροφορίες πληροφορίες μας σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα. Όμως πρέπει να σας πω ότι ανησυχούμε, ανησυχούμε βαθύτατα και εδώ συμφωνώ με τον κύριο Καρίμ ότι πράγματι πολύ συχνά ακούμε τα ίδια και τα ίδια από τις αρχές του Μπαγκλαντές και κατ' ουσίαν ε, τα τελευταία χρόνια οι απαντήσεις δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Ξακολουθούμε λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι. Πιστεύουμε όμως ότι τελικά έχει ξεκινήσει διάλογος και εμεί θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτή την οδό, την οδό του διαλόγου διότι το περάσουμε σε μια άλλη προσέγγιση, μια προσέγγιση επιβολής κυρώσεων, θα πρέπει τότε, αν το κάνουμε αυτό, να σκεφτούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος ηττημένος. Ε, παρόλα αυτά υπάρχουν όλα τα εργαλεία, είναι ανοιχτά. Ε, γνωρίζετε ότι όσοι είναι οι ε, αποδέκτες τέτοιων ε, δυνατοτήτων που προσφέρουμε ε, πρέπει να τηρεί συγκεκριμένα εργασιακά δικαιώματα. Άρα δηλαδή όσον αφορά τη βεντάλια ε, μέτρων που έχουμε στη διάθεσή μας πράγματι υπάρχει και αυτό αλλά θα είναι το τελευταίο το έσχατο που θα χρησιμοποιήσουμε αν δεν λειτουργήσει κανένα άλλο μέτρο. Ε, αν διαβάσει κανείς τις εκθέσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ε, και αν έχοντας ακούσει και την εκπρόσωπο του Διεθνούς Γραφείου, την κυρία Κιόρτης, θα κατάλαβε ότι η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων έχει καταγράψει ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Άρα δηλαδή η εικόνα ε, είναι μεικτή, έχει πάρα πολλά στοιχεία και ως εκ τούτου δεν πρέπει να τιμωρήσουμε τη χώρα. Ε, το μήνυμα που έχουμε λάβει είναι ότι πρέπει να δώσουμε κάποιο χώρο στο Μπαγκλαντές να μπορεί να αναπνεύσει για να μπορεί να συνεχίσει ε, τις μεταρρυθμίσεις που έχει ήδη δρομολογήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Α, συγγνώμη. Και το τελευταίο σχόλιο πριν βάλουμε τελεία. Τι με λιγενέστε. Στα μέσα Μαρτίου, σε λίγες εβδομάδες, θα συνεδριώσουμε στην ΤΑΚΑ. Πρόκειται για τη συνεδρίαση 3 5 προκειμένου να δούμε τις τελευταίες συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και αργότερα μέσα στο 2018 σε συνεργασία με τον ΟΣΑ θα διευκολύνουμε τον διάλογο για τις πρακτικές ανεφοδιασμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους, τα μεταποιητικά εργοστάσια στον τομέα της ένδυσης. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους της ΕΕΔ θα ήθελα να εκφράσω την απόλυτη συμφωνία μου με τα λεγόμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά το διάλογο και την προσέγγιση που εθετούμε απέναντι στον Μπαγκλαντές. Έχουμε συνεχή διάλογο και τακτικά διαμηνύουμε την ανάγκη εφαρμογής των υποχρεώσεων για να προχωρήσουμε. Και όπως είπε και κάποιος καλεσμένος σας, βρισκόμαστε σε ένα ιδιαίτερο πλαίσιο που ισχύει αυτή τη στιγμή στον Μπαγκλαντές λόγω της πρωτοφανούς άφηξης προσφύγων Ροχίνγκια με την κρίση που δημιουργήθηκε στην Βυρμανία. Αυτή η κατάσταση ήταν άνευ προηγουμένου και θα πρέπει να το λαμβάνουμε και αυτό υπόψη όταν συζητούμε για τη χώρα. Ε, πάντως ε, υποστηρίζουμε και πολιτικά και οικονομικά την ε, χώρα αυτή, τον Παγκλαντές, που με πολύ γενοδορία υποδέχεται τους πρόσφυγες από το Μιανμάρ. Και μάλιστα στην τελευταία διάσκεψη των δωρητών ε, έγιναν πολλές υποσχέσεις και επιδιώκουμε τη συνέχιση της οικονομικής αρρωγής. Επίσης, παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς και τις επερχόμενες εκλογές ενώ έχουμε ταυτόχρονα και τακτικό διάλογο στις κοινέ Επιτροπές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Χριστής Διακυβέρνησης. Και μάλιστα θα έχουμε και στην ΤΑΚΑ την, την άνοιξη την ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε και εκεί συχνά επισημαίνουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, την, ε, το κράτος δικαίου και τις ε, προσδοκίες μας σε ό,τι αφορά τις εκθέσεις, την τήρηση των συστάσεων των εκθέσεων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας και της εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας. Τώρα, ως προς την, τις αποστολές παρακολούθησης σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία EBA όλα πλήν των όπλων και θα παρακολουθούμε και το θέμα αυτό φυσικά προσεκτικά. Ε, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Μπαγκλαντές για το 2021 επιδιώκει το καθεστώς ε, της χώρας που δικαιούται ενισχυμένο σύστημα προτιμήσεων, GSP-SYN. Και θα πρέπει στο μεταξύ να έχουν ε, εγκριθεί, κυρωθεί και εφαρμοστεί οι σχετικές συμφωνίες. Θεωρείται ρεαλιστική αυτή την προοπτική ώστε να ολοκληρωθούν όλα αυτά μέχρι το 2021 για να λάβει το καθεστώ των ενισχυμένων δασμολογικών προτιμήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, το εξετάσαμε και κρίνουμε ότι παρά είναι αισιόδοξο το χρονοδιάγραμμα του 2021 καταρχήν. Ε, τα Ηνωμένα Έθνη είναι το όργανο λήψη αποφάσεων. Εκεί αποφασίζει τα, Ηνωμένα Έθνη αποφασίζουν αν μια χώρα πρέπει να χαρακτηρίζονται λιγότερο ανεπτυγμένε ή όχι. Και πρέπει να περάσουν 9 χρόνια συνήθω μεταξύ της ε, ε, τήρησης των ε, κριτηρίων και της σταδιακής ε, από, απομάκρυσης από τον κατάλογο των λιγότερων αναπτυγμένων χωρών, των LDCs. Μέχρι στιγμής δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Αλλά αν από του χρόνου δεν πληρεί πια τον Παγκλαντές τα κριτήρια για να είναι οικονομικά και κοινωνικά λιγότερο αναπτυγμένη χώρα, θα πρέπει να περάσουν 9 χρόνια μέχρι να ε, εφαρμοστεί εμπράκτος αυτή η διαδικασία. Γιατί θα πρέπει να προηγηθούν συζητήσεις, ε, αποδοχή, θα πρέπει το Μπαγκλαντές ε, να δεχτεί αυτό τον αποχαρακτηρισμό τις λιγότερο αναπτυγμένε χώρες. Υπάρχει και μια περίοδο χάριτος όπου η χώρα θα πρέπει να αποδεχθεί και να προσαρμοστεί στις αλλαγές. Δεν πρόκειται να γίνει λοιπόν αυτό πολύ γρήγορα. Αλλά ανάλογα με το πώς θα συμβεί και το τι μορφή θα έχει ο νέος κανονισμός ε, για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και ανάλογα με τα κατα... σίγουρα εκεί ο σεβασμός ε, της σύμβασης ε, θα είναι προαπαιτούμενο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υποβάλω και ερώτηση δεν υπάρχουν μάλλον άλλες ερωτήσεις προς τους εμπειρογνωμόνες μας, στους καλεσμένους. δεν ξέρω αν κανείς επήγεται να δευτερολογήσει. Αν όχι, να σας ευχαριστήσω θερμά και να ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον μόνιμο εισηγητή, τον κύριο Καρίμ, για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καθώς κλείνω θα αρχίσω από εκεί που ξεκίνησα και πριν. Ευχαριστώντας όλους τους προσκεκλημένους που ήρθαν εδώ να συμμετέχουν. Είναι πολύ σημαντικό για μας το ότι βρήκατε το χρόνο να μας δώσετε τα στοιχεία σας. Δεν θα ήθελα κανείς να φύγει από το κτίριο και ε, αισθανόμενος ότι δεν εκτιμήθηκε ο χρόνος του και η συμμετοχή του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Το καλύτερο θα ήταν να κλείσω ακριβώς επί του θέματος που μόλις ανέφερε η Κομισιόν. Είναι ένα εξαιρετικά λεπτό ζήτημα αυτό. Το 2021 είναι κάτι παραπάνω από υπερφιλόδοξο για το να αποκτήσει το καθεστώς ε, που θα το βγάλει από τις LDC, τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια κατάσταση όπου η κυβέρνηση έχει στριμωχτεί σε μια αγωνία όσον αφορά τις φιλοδοξίες που έχει δηλώσει σε σχέση με τι είναι εφικτό. Η Κομισιόν έχει δίκιο. Αυτό που χρειάζεται εδώ είναι να δημιουργηθεί ένα κοινό πρόγραμμα εργασίας μεταξύ του Μπαγκλαντές και των Ηνωμένων Εθνών. Ενδεχομένως το 2021 τα Ηνωμένα Έθνη διαπιστώσουν ότι μπορούν να κάνουν ανακοινώσεις. Όμως αυτό δεν θα είναι το τέλος. θα υπάρξει ανάγκη συνεργασίας με τον Μπαγκλαντές επί Έξι, 6-7 χρόνια, πριν καταλήξουμε σε κάποια τέλος. Και πολλά, πάρα πολλά διακυβεύονται σχετικά με το αν θα κρατήσει την προσβασιμότητα του το Μπαγκλαντές στα πλαίσια των προγραμμάτων γενικευμένων προτιμήσεων. Πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους σε μια μεταβατική φάση, όπως καθώς εκείνοι συνεργάζονται με τα Ηνωμένα Έθνη για την αποφύτισή τους, για την εξέλιξή τους. Αυτό είναι εφικτό Μπορούμε να το κάνουμε. Νομίζω όμως ότι η κοινή γνώμη της χώρας είναι απολύτως ενήμερη για το τι ακριβώς θα γίνει, πώς θα γίνει, ποια θα είναι η φάση μετα... μεταβατική φάση και η φάση αποφύτησης. Είναι δύσκολη κατάσταση, δεν μπορεί κανείς να την αποφύγει και βεβαίως έχουμε και εμείς τις δικές μας δυναμικές εκλογές του 19 υπάρχει εδώ αυτό το θέμα. Το Ηνωμένα Έθνη είπαν ότι τελικά το Μπαγκλαντές δεν θα περάσει πριν από το 2024 στη, στη, στην ομάδα των χωρών μεσαίου εισοδήματος. Θα υπάρχει νέα κομισιόν, νέο κοινοβούλιο το 2024, άρα η δυναμική είναι πάρα πολύ σημαντική για την μετατόπιση των στόχων, καταστόχων, των στόχων κινούμενη άμμος και άρα είναι ακόμα πιο σοβαρό πριν από τις εκλογές του 2019 να έχει δημιουργηθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας με τον Μπαγκλαντές με συμφωνημένες προτεραιότητες και ένα μια συμφωνημένη διαδρομή για τη σχέση μας. Βλέπω όμως ότι υπάρχουν πολλές, πολλοί κίνδυνοι και παγίδες ε, πριν φτάσουμε στο σημείο αυτό. Αυτά έχω να πω, δεν ακούγονται πολύ αισιόδοξα, αλλά είναι η καλύτερη ε, πορεία που μπορώ να χαράξω. Δε, υπάρχει ανάγκη σοβαρότατου διαλόγου μεταξύ ημών και του Μπαγκλαντές, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πράγματι, κύριε Κάριμ, πρέπει να ακολουθήσουμε την οδό αυτή και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια ξεκάθαρη προοπτική πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Χάρη λοιπόν στους εμπειρογνώμονες είμαι πεπισμένος ότι θα εξακολουθήσουμε να είμαστε σε επαφή επί του θέματος. Μην διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας αν το θεωρήσετε απαραίτητο. Ευχαριστούμε και πάλι. Λοιπόν, ε, πάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 21. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ σημαντικό θέμα. Συγητήσω ο κύριος Βίνκλε. Πρόκειται για, την, ε, για τις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, σημαντικά προβλήματα με την Κίνα. Έχουμε την πολιτική, την εμπορική του 2025, ε, τις 10 προτεραιότητες, πώς θα ε, εντοπιστούν και χαρακτηριστικούν αυτές οι προτεραιότητες, οι στρατηγικές επενδύσεις της Κίνας ε, στην Ευρώπη, κάποιες περιπτώσεις, dumping, πολλά φλέγοντα θέματα. Το Κοινοβούλιο Um, Το Κοινοβούλιο λοιπόν ε, τοποθετείται γενικά στη σχέση με την Κίνα ως εκ τούτου τα πολιτικά κόμματα το πολιτικό θέμα το εξετάζει η ΑΦΕΤ και εμείς εξετάζουμε την εμπορική διάσταση των ε, θεμάτων. Ο εισηγητής μας για όλα αυτά είναι ο κύριος Βίνκλα και θα ήθελα να τόσο το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πίσω από τις Ηνωμένε Πολιτείες, ε, ε, η Κίνα είναι και ο ε, μεγαλύτερος εξαγωγέας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή συνολικά μιλάμε για περίπου ένα δισεκατομμύριο ε, την ημέρα εμπορικό αντικείμενο στη σχέση μας με την Κίνα. Ξέρω ότι τα γνωρίζετε όλα αυτά, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου όλα αυτά τα στοιχεία οποτεδήποτε μιλάμε για τις εμπορικέ σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα. Ο πρόεδρος Σιντσιμπίν ε, στις ε, το 19ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος παρουσίασε την έκθεσή του. Εκεί ε, μίλησε για μια νέα περίοδος που θα ξεκινήσει στην Κίνα. Αυτή ήταν μια ομιλία η οποία απευθύνεται στο εσωτερικό της Κίνας αλλά περιλάμβανε σαφή μηνύματα και για ε, αλλοδαπούς ε, είπε ο πρόεδρος ότι η Κίνα θα ε, επεκτείνει τις εμπορικές της συναλλαγές και την αλυσίδα αξίας είπε ότι θέλει να προσφέρει απελευθέρωση και μεγαλύτερη πρόσβαση στην ιστορική αγορά. Θα ανοίξει την υπηρεσία των υπηρεσιών, ε, θα καλύψει τα συμφέροντα και θα προστατεύσει τα συμφέροντα των εξωτερικών επενδυτών. Δυσμεύτηκε επίσης ότι η Κίνα ε, θα συνεχίσει να προσπαθεί να μην έχει υπερπροσφορά, να έχει μια ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση. Είπε επίσης ότι στηρίζει το πολυμερές εμπορικό σύστημα, την παγκόσμια οικονομία και είπε ότι η Κίνα θα σταθεί θετικά απέναντι στο περιβάλλον, θα συνεργαστεί για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τώρα, αν τα δούμε όλα αυτά ρεαλιστικά, άραγε υπάρχει κάτι το σημαντικό και το ρεαλιστικό σε αυτά που παρουσίασε ο Πρόεδρος. Εμείς ε, θεωρούμε ότι η Κίνα είναι μια νέα Κίνα, ε, διαφορετικές οι εξωτερικές εμπορικές της σχέσεις Υπάρχει κάθε λόγος να πιστεύουμε ότι το εμπόριο θα είναι ε, μια κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της Κίνας ε, στο μέλλον. Ακούσαμε και κατά το παρελθόν πολλές υποσχέσεις ότι θα ανοίξει η αγορά της Κίνας, αλλά δυστυχώς οι επιχειρήσεις μας μας λένε ακριβώς το αντίθετο. Η Κίνα υποσχέθηκε κατά το παρελθόν να περιορίσει την υπερπαραγωγή της, αλλά πολλά προϊόντα της εξακολουθούν να κατακλείζουν τις αγορές μας και να ρίχνουν τις τιμές. Τέλος, δυστυχώς υπάρχει ε, στασιμότητα, διέξοδο και στις σχέσεις με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Η Κίνα δεν σέβεται τους κανόνες, άρα δηλαδή απομένει να δούμε τι θα γίνει τελικά, τι θα κάνει η Κίνα στις καλές εμπορικές σχέσεις. Η Κίνα ε, παλαιότερα ήταν για μας πολύ σημαντική αναπτυσσόμενη αγορά. Τώρα όμως τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγές μας προς την Κίνα δεν έχουν αυξηθεί σημαντικά παρότι έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι εισαγωγές μας κυρίως κατά την προηγούμενη χρονιά. Υπάρχει λοιπόν εμπορικό έλλειμμα προς όφελος της ε, Κίνας Έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση για μάσα, αλλά μόνο κατά τη. Οι άμεσες επενδύσεις ε, προς την Κίνα έχουν μειωθεί, απ' την άλλη οι επενδύσεις της Κίνας προς την Ευρώπη έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η ροή επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Κίνα έχει ξεπεράσει τις επενδύσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προς την Κίνα. Αυτό που δεν υπάρχει ακόμα είναι ένα σαφές νομικό πλαίσιο. Ε, το 2013 ξεκίνησαν οι επενδυτικές διαπραγματεύσεις, αλλά σήμερα έχουμε επιτύχει μόνο με τριοπαθή πρόοδο. Υπάρχει πρόοδο σε κάποιε διαπραγματεύσει με την Κίνα για τι γεωγραφικέ ενδείξει. Υπάρχουν κοινέ πρωτοβουλίε όπω η πλατφόρμα ε, συνδεσιμότητα. Επίση, εργαζόμεθα ε, και καταβάλουμε προσπάθειες να αυξήσουμε τις επενδύσεις μας μέσα από το ΕΦΣΥ και να έχουμε και μια άλλη κοινή πρωτοβουλία με την Κίνα ε, σχετικά με τη ζώνη παριθμών 1. Τέλος πάντων, αυτό που βλέπουμε ότι τα τελευταία προγράμματα δυστυχώς ε, δεν έχουν την απαραίτητη διαφάνεια και δεν καλύπτουν τα πρότυπα της βιωσιμότητας. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να καθορίσουμε το μελλοντικό μας όραμα για τη σχέση σχέσει ανάμεσα στην Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεργαζόμαστε με την ΑΦΕΤ ε, στο πλαίσιο του κανόνα υπαριθμών 54 που σημαίνει τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, τις απόψεις τους ε, για, για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής θα τις εντάξει σε ένα και μόνο ψήφισμα. Όπως είπε και ο Πρόεδρός μας, η Κίνα είναι ένας πολύ σημαντικός εμπορικός εταίρος και αυτό το ψήφισμα προφανώς και είναι δική μας απόλυτη αρμοδιότητα. Να πω και κάποια άλλα θέματα για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Είμαι πεπισμένος ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει μια σταθερή σχέση, ε, να υπάρχει ουσιαστική αμοιβαιότητα στις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις μας με την Κίνα. Είναι επίσης απαραίτητο να ε, συντονίσουμε τις προσπάθειες ε, των επιχειρησιών μας. Η συνεργασία πρέπει να υπερισχύει κυρίως στη σημερινή εποχή όπου βλέπουμε ότι αυξάνεται όλο και περισσότερο ο προστατευτισμός, δηλαδή από τους εταίρους μας πάνε περισσότερο σε γραμμή σύγκρουσης. Ε, εγώ πιστεύω όμως ότι δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να υπάρχει περισσότερη συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκείνη που θα πρέπει να στηρίζει τη συνεργασία. Και αυτό, επαναλαμβάνω, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τα οικονομικά συμφέροντα, τις αξίες και τα συμφέροντα των κρατών μελών και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει, όπως σας είπα, ο κανονισμός υπαρθμών 54. Με βάση αυτόν ε, λειτουργούμε εδώ στην Επιτροπή μας. Ε, έχουμε συζητήσει τις περίπλωσες εμπορικές σχέσεις ε, με τους βασικούς μας εμπορικούς εταίρους και γνωρίζουμε ότι όλα αυτά σημαίνουν ότι δεν υπάρχουν μόνο εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις. Είναι απόλυτα σαφές οι διαπραγματευτέ μας, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης, οι διπλωμάτες μας, τα κρατη όλοι να στέλνουν συντονισμένα μηνύματα στους Κινέζους εταίρους μας. Και μεταξύ άλλων μπορούμε να κάνουμε και αναφορά στις συζητήσεις που έχουν γίνει ότι είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το θέμα του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα θα τηρούμε πλήρως τις υποχρώσεις μας. Να αναφέρω συγκεκριμένο παράδειγμα. Συζητάμε για το νέο μηχανισμό επενδύσεων, το screening των επενδύσεων, συζητάμε ε, οι θεσμοί και τα κράτη-μέλη. Κατά την άποψή μου, αυτή είναι μια αντίδραση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ε, αυτή η στρατηγική ε, είναι απόλυτη απόλυτα ουδέτερη. Ολοκληρώνοντας αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ έχω δεσμευτεί να συνεχίσω τη δουλειά μου ε, με τους συναδέλφους από την ΑΦΕΤ. Όλοι μας θα πρέπει να ακούσουμε την άποψη των ε, εμπειρογνωμόνων όταν θα προετοιμάσουμε τη γνωμοδότησή μας. Οφείλουμε να κατανοήσουμε καλύτερα, να δώσουμε έτσι μια φρέσκια ματιά στις ανάγκες των Κινέζων εταίρων μας. Ε, θεωρώ ότι συμβανέβαλε κατά πολύ και θα συμβάλλει επίσης περισσότερο ότι θα πάμε στην Κίνα το Μάιο. Χαίρομαι ε, για τις απόψεις που θα ακουστούν, για να με βοηθήσουν να συντάξω εγώ την έκθεσή μου και όπως το έχω κάνει και κατά παρελθόν θα συνεχίσω να κάνω ό,τι μπορώ έτσι ώστε να προκύψει ένα ισόρροπο αποτέλεσμα από τη γνωμοδότησή μας. Μια γνωμοδότηση που αφορά έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους μας, ένα εταίρος ο οποίος ε, κατ' ουσίαν καθορίζει ακόμα και την ευημερία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιούλιο Βίνκλερ. Ε, περνάμε στους κοιόδης ηγητές. Κυρία Μακλάρκιν. Yeah, no here, so Α, συγγνώμη, δεν το είχα σημειώσει. Συγγνώμη, εγώ αντικαθιστώ την Αλέσια. Θα μιλήσω εκ μέρους της Αλέσια Μόσκα. Ε, σίγουρα η... είχαμε 170 δισεκατομμύρια το εμπορικό μας έλλειμμα το 2016 και επίση ε, η Κίνα έγινε καθαρό επενδυτή στην Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκέ εξωτερικέ ε, επενδύσει άμεσα στην Κίνα αυξάνονται, ενώ οι ροέ από την ε, Κίνα ακολουθούν αντίστροφη πορεία. Και μάλιστα οι διαπραγματεύσει για επενδυτική συμφωνία έχουν ξεκινήσει από το 2013, αλλά δεν προχωρούν αρκετά. Βέβαια, σίγουρα ε, η Κίνα υπονομεύει το, την Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου μια και θετεί τι υποχρεώσεις να ανοίξει την ε, ενιαία αγορά, την εσωτερική της αγορά ή να ε, υπονομεύει τις πολυμερείς σχέσεις παρόλο που δημοσίως ισχυρίζεται το αντίθετο. Σίγουρα η Κίνα αυξάνει την επιρροή της και στις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στις γειτονικές χώρες. Οι γεωπολιτικά προσανατολισμένες επενδύσεις της ε, υπονομεύουν την ενότητα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα ε, είδαμε την αλλαγή της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην Κίνα μετά την αγορά βασικών υποδομών της Ελλάδας από Κινέους επενδυτές όπως το λιμάνι του Πειραιά ή ε, ηλεκτρικό δίκτυο. Η Κίνα ασκεί τεράστιες, τεράστια επιρροή στην Ελλάδα και θυμάμαι μάλιστα όταν η κινα ασκει τεραστια μπλόκαρε ε, μία δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη ε, προκειμένου να μην καταδικάσουμε τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το πώς εφαρμόζει τα ανθρώπινα δικαιώματα η Κίνα είναι κατά και του μηχανισμού ελέγχου των επενδύσεων η Ελλάδα λόγω των στενών σχέσεων που έχει με την Κίνα. Θα πρέπει λοιπόν να, να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένους αριθμούς και στοιχεία. Εγώ περιλαμβα... προτείνω τη συμπερίληψη των ακόλουθων σημείων. Άμεση εφαρμογή της πρότασης για την θέσπιση μηχανισμού ελέγχου των ξένων επενδύσεων από τους συνομοθέτες. Δεύτερον, θα πρέπει να αναζωογονήσουμε τις συζητήσεις για τις διεθνείς ε, ε, δημόσιες συμβάσεις και να λάβουμε υπόψη τα συμπεράσματα του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση. Τρίτον, είναι σημαντικό να ολοκληρωθούν οι επενδυτικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα πριν ε, ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Ταϊβάν και το Χονγκ Κόνγκ ε, να δούμε πώς θα αποκαταστήσουμε συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού για τους Ευρωπαίους επενδυτές και να ξεκινήσουμε άμεσες διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις και του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν. Η Αλέσα Μόσκα προσβλέπει σε αγαστή συνεργασία με τον εισηγητή προκειμένου να καταλήξουμε σε ισχυρή κοινή θέση της Επιτροπής. Και τώρα η ΕΜΑ. Η σχέ... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η εμπορική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας είναι από τις ε, σημαντικότερες στον κόσμο και γι' αυτό όπως είπε ο εισηγητής, ε, έχουμε φτάσει τα 515 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο το 2016. Ε, άρα είναι απολύτως σαφές ότι ο όγκος του εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Κίνας, ακόμα και χωρίς συμφωνία, είναι τεράστιος και αυτός δείχνει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη εμπορική συμφωνία κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά σε τώρα στις υποεξέλιξη διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας και την συμφωνία για τις επενδύσεις επενδύσεις που μπορεί να θεωρηθεί ως πλατφόρμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι επενδυτές στην Κίνα. Τα συσσωρευτικά στοιχεία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνα είναι χαμηλότερα από αυτά με τις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα και πρέπει να βρούμε τρόπους να προχωρήσουμε. Ε, σε αυτή, μέσα σε αυτή τη συμφωνία επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών. Και άρα μέσω αυτή τη συμφωνία ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να δώσουμε κίνητρα για την αγορά αντιμετωπίζοντα θέματα όπως το κανονιστικό περιβάλλον, η έλλειψη διακρίσεων, όπως επίσης και οι εγγυήσει ε, της μεταχείρισης των Ευρωπαίων επενδυτών και αντιστρόφως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή προσπαθεί να δημιουργήσει νέα κανονιστικά μέσα όπως το Διεθνές Μέσο Προμηθειών και το ε, Μέσο Επενδύσεων για να δημιουργήσει συνθήκες ισότητας και στην κινέζικη αγορά. Άρα θεωρούμε ότι αυτό θα επιτευχθεί καλύτερα στο πλαίσιο αυτής της διμερούς διαπραγμάτευσης. Επίσης θα έπρεπε να δούμε ότι πρέπει να επιδιώξουμε καλύτερη συνεργασία στον τομέα της τεχνολογίας και κοινοτομίας. Πολλά μπορούμε να κάνουμε από κοινού. Όμως για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις μας να κοινοτομήσουν και να αναπτύξουν ε, προϊόντα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η πνευματική ιδιοκτησία θα προστατεύεται πλήρως και να συνεχίσει η λειτουργία του μηχανισμού προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Πρέπει όλα αυτά από κοινού να μας οδηγήσουν δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου προστασία τη διανοητική ιδιοκτησία και της πρόθεσης του δίκαιου ανταγωνισμού και της κοινοτομία στο μέλλον. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την δουλειά που συνεχίζει να κάνει στο θέμα αυτό και προσβλέπω στη συνεργασία μας στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριο Χέλμουντ Σόλτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αναμφίβολα λοιπόν πρόκειται για ένα ιδιαίτερα περίπλοκο θέμα αυτό με το οποίο ασχολούμαστε τώρα και γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολο να διαχωρίσει κανείς που θα ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει τα πολιτικά, θα ξεκινήσει τα οικονομικά, σε θέματα ανάπτυξης που τελικά είναι προϋπόθεση για την Κίνα έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι οι οποίοι αναφέρθηκαν στο τελευταίο συνέδριο του κόμματος. Εγώ συμφωνώ με τον εισηγητή ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιλέξουμε ορισμένα θέματα και να επισημάνουμε ε, το πού και σε ποιους τομείς πρέπει να συνεργαστούμε. Κυρίως ε, όσον αφορά την επενδυτική συμφωνία, η οποία ε, κατά την άποψή μου πρέπει να προσπαθήσουμε να την επιταχύνουμε. Να επιταχύνουμε δηλαδή τη σύναψή της. Κατά τα άλλα, δυστυχώς τώρα η σκιώδη συζυγήτρια του ε, των σοσιαλιστών, των σοσιαλδημοκρατών έφυγε και δεν θα τα ακούσει, αλλά εγώ θα το πω δεν χρειάζεται να φοβόμαστε την Κίνα. 1,3 δις άνθρωποι αν αυτοί θελήσουν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους, να υιοθετήσουν το δικό μας τον τρόπο ζωής, προφανώς και θα καταναλώνουν πόρους. Και προφανώς θα πρέπει να ενισχυθεί η δική τους η βιομηχανία, η γεωργική τους παραγωγή και αυτά, κατά την άποψή μου, πρέπει να τα αντιμετωπίσει κανείς με απόλυτη ειλικρίνεια. Όσον αφορά δε τη διμερή σχέση, είναι σαφές ότι θα πρέπει να εκφράζονται τα συμφέροντα των δύο πλευρών. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε συμφέροντα και όσον αφορά το σύνολο των συμφερόντων μας, έχουμε και επιμέρους συμφέροντα. Συμφέροντα κρατών και πιο κάτω επιμέρους, επιμέρους ομάδων, πληθυσμιακών, ε, μειονοτήτων, οτιδήποτε Μιλάμε δηλαδή για μια περίπλοκη παγκόσμια οικονομία. Ε, εκείνο το οποίο διακυβεύεται αυτή τη στιγμή είναι πώς θα μπορέσουμε κι εμείς ε, να επηρεάσουμε την παγκόσμια οικονομία. Εάν όμως φοβόμαστε την Κίνα, τις επενδύσεις τους για τον τύπο, ε, διαβάζουμε συνεχώς κίτρινος κίνδυνος και ούτω καθεξής. Στοιχεία στην Γερμανία το 2017, το 2017 μειώθηκε η εξαγορά επιχειρήσεων από την Κίνα σε σχέση με το 2016. Συγκεκριμένα, το 2016 Είχαμε 68 γερμανικές επιχειρήσεις σε κινέζικα χέρια, μειώθηκαν σε 45. Το 2017 βέβαια οι κινέζοι επενδυτές ε, επένδυσαν μόνο 12,6 δις δολάρια. Στη Γερμανία αυτή τη στιγμή έχουμε 54 συναλλαγές, ε, επενδυτικές συναλλαγές με την Κίνα, άρα δηλαδή είναι ο πρώτος επενδυτής στη Γερμανία, μετά ακολουθούν οι Βρετανοί και μετά οι Ιταλοί. Παράλληλα, να σας πω και το εξής, ότι στη Γερμανία το ίδιο χρονικό διάστημα είχαμε 155 εξαγορές από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ακολουθούν οι Ελβετοί και μετά οι Βρετανοί που αγόρασαν πάνω από 80 γερμανικές επιχειρήσεις. Με άλλα λόγια, έχουμε στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά για την οικονομία της αγοράς. Τίθεται λοιπόν το εξής ερώτημα. Τα ε, κριτήρια δημόσιων διαγωνισμών και οι προϋποθέσεις γενικότερα, πώς θα πρέπει να διαμορφωθούν. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να το εξετάσουμε αυτό στη δική μας την Επιτροπή. Να δούμε ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να ισχύουν για την επενδυτική δραστηριότητα. Τι πρέπει να γίνεται όταν κάνουμε το screening των επενδυτών. Πώς διασφαλίζονται οι θέσεις απασχόλησης. Πόσο μακροπρόθεσμα θα είναι τα χορηγούμενα δάνεια. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να συμβάλλουμε έτσι ώστε να βελτιωθούν περαιτέρω οι ε, εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις μας με την Κίνα. Πραγματικά περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον τη συνεργασία με τον εισηγητή. Είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριο Ντάρτμαουθ. Ευχαριστώ. Μπορεί να σας σοκάρει. Τέσσερις προτάσεις ε, θα διατυπώσω μόνο. Η κυρία Μακλάρκιν πολύ ε, εύστοχα μίλησε για την αξία και τον όγκο εμπορίου που γίνεται μεταξύ των 28 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας. Επίσης, επισήμανε βλωτά ε, ότι χωρίς ε, εμπορική συμφωνία και αυτό επιβεβαιώνει δεν χρειάζεται κανείς εμπορική συμφωνία για να έχετε τεράστιο τεράστιο όγκο εμπορικών συναλλαγών. Επίση, έχω μια απλούστατη ερώτηση προ τον εισηγητή και δεν είναι καθόλου εύκολο να απαντηθεί, παρόλο που είναι απλή ερώτηση. Αναφέρεται συνήθω ότι όταν μιλούμε για την Κίνα και το εμπόριο, πολύ συχνά αναφέρεται ότι η Κίνα δεν ακολουθεί τους κανόνες, δεν σέβεται τους κανόνες του παιχνιδιού, όπως κάνουν άλλοι εταίροι. Δεν θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση τον εισηγητή μας, ούτε να το στριμώξω. Απλώς το ρωτάω να μου πει αν γνωρίζει. Θεωρεί ότι ισχύει αυτό το σχόλιο ε, είναι ακριβές, ανακριβές, ε, είναι μισή... Υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό το σχόλιο ή όχι. Ισχύει ότι η Κίνα δεν σέβεται τους κανόνες του εμπορικού παιχνιδιού και παίζει βρώμικο παιχνίδι κατά κάποιο τρόπο. Γιατί αυτό ακούγεται πολλές φορές όταν γίνεται συζήτηση για την Κίνα και το εμπόριο. Ο εισηγητής που γνωρίζει αυτά τα πράγματα, τι γνώμη έχει. Ε, κύριε Ντάρθμουθ, θεωρείτε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε παίζουν με τους κανόνες του παιχνιδιού, σέβονται τους κανόνες του παιχνιδιού. Φαντάζομαι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Παρατήρηση πρώτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τη μόχλευση που έχει και τους μηχανισμούς μόχλευσης. Ε, και ε, αυτό να φανεί στη νέα μεθολογία και την, ε, η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διαρευνητικό έλεγχο των άμεσων ξένων παιδίσεων είναι καλή πρόταση. Δείχνει έτσι ότι είμαστε ενωμένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Κινέζικη τακτική του Διέρη και Βασίλευε. Ε, κατά τη γνώμη μα, κατά τη γνώμη των πρασίνων, το screening των άμεσων ξένων επενδύσεων είναι σημαντικό μηχανισμό των εξωτερικών σχέσεων και τρόπο διαφύλαξη του δημοκρατικού μα ε, μοντέλου. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει για την επενδυτική συμφωνία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ουδέποτε δεν πρόκειται να δεχθεί μια συμφωνία που έχει αμφίβολης αξίας ε, προτάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει να προσπίσουμε το με μοντέλο μας για βιώσιμο εμπόριο, ιδιαίτερα στη σχέση μας με την Κίνα. Και τέλος, δεδομένων των νέων προκλήσεων που ε, ανέκυψαν την τελευταία πενταετία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς ε, σκοπεύει να προσαρμόσει την ε, Ευρωπαϊκή Στρατηγική απέναντι στην Κίνα σε ό,τι αφορά το εμπόριο και τις επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να διαχωρίσει το εμπόριο από τις επενδύσεις. Δεν θα πρέπει, που δεν είναι να επιδιώξει μόνο άνοιγμα της αγοράς, αλλά θα πρέπει να υιοθετήσει μια πιο στρατηγική προσέγγιση του συνόλου των σχέσεων μας με την Κίνα. Ευχαριστώ και τώρα η Κομισιόν. Ποιος θέλει να πάρει τον λόγο. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο για τα πολύ εύστοχα σχόλιά του. Όλοι θυμόμαστε βασικά στοιχεία και νούμερα για την κατάσταση με την Κίνα. Δεν θα τα επαναλάβω. Όμως είναι διαμφισβήτητο ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Κίνα είναι ε, βασικός εμπορικός εταίρος για την Ένωση και άρα είναι σημαντικός εταίρος για τις επιχειρήσεις μας και ότι πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξαρτώνται από την κινέζικη αγορά ενώ πολλές εταιρείες της Ένωσης ε, έχουν πολλά κέρδη, μεγάλο μέρος των κερδών τους στην Κίνα. Άρα η πρόσβαση στην Κίνα είναι ζωτική σημασία για την παγκόσμια στρατηγική τους. Κατόπιν αυτών όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την πραγματικότητα κάποιων δυσκολιών που προκύπτουν με την Κίνα. Αυτό αναφέρθηκε και από κάποιους από τους ομιλητές. Μπορούμε να πούμε <clears throat> ότι η διμερής εμπορική σχέση με την Κίνα είναι από τις πιο σύνθετες από αυτές που έχουμε όλους τους εμπορικού εταίρους. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε θέματα κρίσιμης σημασίας και εσείς Πρόεδρε αναφερθήκατε σε κάποια από αυτά όπως έλλειψη αμοιβαιότητας, πρόβλημα ισότητας αντιμετώπισης, υπερπαραγωγικότητα, το θέμα της πρόσβασης της αγοράς ε, κάποιων στην αγορά της Κίνας. Αυτά είναι πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επιχειρήσεις μας και πρέπει να προσπαθήσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώς, όταν βλέπουμε τι γίνεται στην Κίνα και ο κύριος Βίνκλερ αναφέρθηκε κάπως και σε αυτό, <clears throat> είναι σαφές ότι η μεταρρυθμισή δεν έχει οδηγήσει σε χειροπιαστή τα ανοίγματα στην αγορά των επιχειρήσεών μας και όχι μόνο των δικών μας και των Αμερικανικών και των Ιαπωνικών και γενικά όλων των ξένων επιχειρήσεων. Και υπάρχουν και ενδείξεις ότι η κινέζικη αγορά κλείνει λόγω κανονισμών που κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση. Θέματα ασφάλειας, οι κανονιστικές απαιτήσεις ή πραγματικά διακρίσεις, καθαρές διακρίσεις κατά των ξένων επιχειρήσεων, απλά και μόνο επειδή δεν είναι κινέζικες. Αυτό που είδαμε από το, την συνέλευση του κόμματος ε, πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ενισχυμένος έλεγχος από το κόμμα στις κρατικές επιχειρήσεις της Κίνας και όπως ακούσαμε μια πιο πιεστική Κίνα σε διεθνές επίπεδο. Αυτό είναι προβληματικό. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς τώρα θέματα επιδοτήσεων, ε, απαιτήσεων για τοπικό περιεχόμενο και κάποια άλλα αμφιλεγόμενα θέματα, το σύστημα των ε, κοινωνικών πιστώσεων, που από ό,τι δείχνουν, ε, από ό,τι φαίνεται δείχνουν ότι η Κίνα δεν παίζει με τους ίδιους κανόνες ε, απέναντι στις εταιρείε μας. Ε, βλέπουμε μια εξαιρετικά φιλόδοξη Κίνα, η οποία θα συνεχίσει και το λέει ξεκάθαρα, με τα σχέδιά της, θα συνεχίσει να ενισχύει την εσωτερική της βιομηχανία κυρίως με βάση τη στρατηγική Made in China 2025 βλέπουμε ότι η Κίνα πηγαίνει, βγαίνει στον κόσμο κυρίως με την πρωτοβουλία της One Belt One Road και έχει γίνει περιορισμένη πρόοδο σε θέματα ε, διαφάνειας και βιώσιμης ανάπτυξης Τώρα πάλι βλέπουμε ότι η Κίνα προσπαθεί να υπονομεύσει τους πολυτερούς, πολυμερείς οργανισμούς και το ρόλο τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε αντιμετωπίσει μια σοβαρή πρόκληση. Το ερώτημα είναι πώς θα βρεθεί η σωστή ισορροπία που θα εγγυάται ότι μπορούμε να αναπτύξουμε μια σωστή εμπορική σχέση με την Κίνα που όπως είπα αρχικά είναι σημαντικός εταίρος. Έχουμε τις διαπραγματεύσεις για τις επενδύσεις που αναφέρατε. Θα εξακολουθήσουμε να πιέζουμε ως σύνολο αλλά και ως κράτη-μέλη για μια αμοιβαιότητα στη σχέση, μεγαλύτερη ισότητα για να αντιμετωπιστούν σοβαρά τα θέματα της υπερβολικής δυναμικότητας, της... αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες. Όταν δείχνουμε ενότητα, όταν δείχνουμε το τη δύναμή μας μπορούμε να προχωρήσουμε. Ας πούμε, καταφέραμε πέρυσι να καθυστερήσουμε την υλοποίηση, των, την εφαρμογή των νέων προτύπων των νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την Κίνα που δημιουργούσε προβλήματα στη βιομηχανία μας. Πείσαμε τους Κινέζους να σταματήσουν τον νέο κανονισμό για τις ε, πιστοποιητικά εισαγωγή τροφίμων που θα έκλεινε εντελώ την ε, η κινέζικη αγορά σε εξαγωγή τροφίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ήταν σοβαρό θέμα για τις επιχειρήσεις μας. Ε, γίνονται η διαπραγματεύση για τις επενδύσεις παρότι πράγματι η πρόοδος είναι αργή, πορούν επειδή οι αρχικές θέσεις είναι πολύ διαφορετικές και υπάρχουν θεμελιώδη ζητήματα. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση για τις γεωγραφικές ενδείξεις η οποία συνεχίζεται και είναι και σε καλό δρόμο. Και σε πολυμερές επίπεδο θα διαπιστώσατε ότι καταφέραμε στη δημιουργία του Παγκοσμίου Φόρουμ G20 για την ε, παραγωγικότητα του Χάλιβα και αναγκάσαμε την Κίνα να, να μας δώσει στοιχεία για τη ε, βιομηχανική παραγωγή. Αυτές είναι κάποιες θετικές εξελίξεις, αλλά πρόκειται για σοβαρή προσπάθεια που απαιτεί ε, δέσμευση από μας. Έχουμε την ε, υποστήριξη με την έγκριση της νέας μεθοδολογίας anti-dumping. Θα είδατε και τα θέματα των στρεβλώσεων με την Κίνα. Έχουμε τον ε, εξυγχρονισμό των ε, μέσων εμπορικής άμυνας και το, διεθνές, το εργαλείο για τις διεθνείς δημόσιες συμβάσεις. Όλα αυτά μας δίνουν τα μέσα να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που έχουμε με την Κίνα. Και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινάμε με άλλες χώρες που συμφωνούν μαζί μας όπως οι Ηνωμένες και η Ιαπωνία. Σωστά επισημάνατε την υπουργική δήλωση που έγινε στο περιθώριο της διάσκεψης του Buenos που αφορά ε, μια σειρά από πρακτικές πολιτικές και την αντιμετώπιση τους, που ε, κάποιες έχουν σχέση και με την Κίνα. Εν κατακλείδη λοιπόν και για να είμαι ειλικρινής εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές δυσκολίες για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών με την Κίνα κυρίως στο τομέα του εμπορίου γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ ανοιχτή απέναντι στην Κίνα και στις επενδύσεις και στην εμπορία προϊόντων και άρα ε, ε, δεν μπορούμε να επιφέρουμε τόσο μεγάλη ισορροπία όταν ήδη είμαστε πολύ ανοιχτοί στις κινέζικες επιχειρήσεις. Αν όμως καταφέρουμε να μοχλέψουμε λίγο τις δραστηριότητες της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών και όλων των θεσμικών οργάνων με τρόπο συνεκτικό ε, για να και συντονιστούμε με τους βιομηχανικούς κλάδους θα μπορέσουμε να κινηθούμε και να ασκήσουμε πίεση προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει λοιπόν να υπενθυμίσουμε την κατάσταση και με πολύ μεγάλη χαρά θα σας στηρίξουμε στην προσπάθεια αυτή. Αν η Επιτροπή σας επισκέψει την Κίνα, όπως είπατε, με τα μεγάλης χαράς θα θέλαμε να σας υποστηρίξουμε ε, με συγκεκριμένες ενημερώσεις, έγγραφα και όλα επί όλων των σχετικών εμπορικών θεμάτων που σήμερα αναφέρθηκαν. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Thanks ευχαριστούμε. Όντως, ε, μεγάλη ευκαιρία να επιλύσουμε τις εκκρεμότητες. Αλλά ε, τις μικρότερες προκλήσεις μπορούν να τις ε, αντιμετωπίσουν και άλλα ίσονα σημασίας ε, όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τις μείζονες προκλήσεις καλύτερα να τις αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι και σημαντικότατο όργανο. Τώρα ε, θα δώσω το λόγο σε κάποιον από τη Βόρεια Ευρώπη που μπορεί να μην ο πλέον έμπειρος ε, της ομάδας αλλά εργάζεται σκληρά για την Επιτροπή και εδώ και πολύ καιρό και σήμερα είναι η τελευταία του συνεδρίαση στην ε, Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου γιατί θα φύγει. Ευχαριστούμε για το έργο σου στην Επιτροπή για την εμπιστοσύνη σου και καλή επιτυχία στο μέλλον. Σε ευχόμαστε. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τι να πω. Ήταν ε, πραγματικά τιμή μου και μεγάλο προνόμιο που εργάστηκα στην Επιτροπή σας και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ε, χαρακτηριστική λιτή φιλανδική απάντηση. Σας ευχαριστούμε. Γιούλιου Βίνκλερ, έχετε το λόγο. Ε, θα ήθελα και εγώ, πριν περάσω στο τελευταίο σκέλος της ε, παρέμβασής μου, να συγχαρώ και να αποχαιρετήσω το γραμματέα μας, τον κύριο Χάιντι, Χάικη Σότη, να τον ευχαριστήσω θερμά για την ανεκτήμητη ε, βοήθειά του και σίγουρα η λακωνική αποχαιρετιστήρια ομιλία του είναι ενδεικτική τη μεγάλη αξία του ούκα το εφα. Ευχαριστώ του συναδέλφου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχόλιά του και είμαι βέβαιο ότι βρισκόμαστε στην αρχή αυτών των συζητήσεων. Θα πρέπει να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να εντάξουμε τα πιο σημαντικά σημεία στην έκθεση αυτή. Φυσικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε επί παντός επιστητού, γιατί είναι πολλά τα σημαντικά θέματα, δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα, αλλά θέλουμε μια έκθεση που πραγματικά να αντικατοπτρίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επειδή με προκάλεσε ο παλιός μας συνάδελφος ο κύριος Ντάρτμοντ ε, για την, ε, και την ε, δημοσκόπηση που έκανε ή την έρευνα που έκανε η απάντησή μου είναι όχι, ότι δεν ισχύουν συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού με την Κίνα ή τουλάχιστον δεν είναι αρκετά ισότιμος ανταγωνισμός με την Κίνα και πιστεύω ότι με την έκθεσή μας θα συμβάλλουμε στο να αποκατασταθεί θεμετώ ή πιο θεμητό ή πιο ισότιμο ανταγωνισμό. Η δεύτερη ερώτηση ήταν πιο ε, πονηρή. Με ρωτήσατε αν ε, παίζει καθαρό παιχνίδι ή όχι η Κίνα ή αν παιζει καθαρο παιχνιδι οχι η κινα η αν ειναι εν μέρει αληθή αυτή η διαπίστωση ή όχι. Μπορώ να σας ε, απαντήσω ότι η διαπίστωση αυτή είναι ταυτόχρονα και αληθής και εσφαλμένη όχι μόνο βλέπουμε και το βεβαιώνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Εμπορικό μας Επιμελητήριο στην Κίνα δείχνουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι Κινέζοι πραγματικά παρακάπτουν τους κανόνες και έχουμε τέτοια παραδείγματα παραβίασης των κανόνων, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και μία συνεχή συζήτηση για τις ευρωπαϊκές μας αξίες, γιατί αυτό που θέλουμε είναι να ε, στηριχθούμε στις αξίες μας, οπότε με αυτές ε, πηγαίνουμε στην Κίνα. Και διαπιστώνουμε ότι και οι Κινέζοι έχουν αξίες και καλό είναι να τις αξιοποιήσουμε και αυτές. Αν λοιπόν αξιοποιήσουμε τις αξίες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτους δικαίου, δημοκρατίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι εταίροι Κινέζοι μας ε, εδράζονται σε κάτι που αποκαλούν κινέζικες αξίες. Και οι αξίες στο ΜΕΝ και το δεν μπορεί να μην συμπίπτουν 100% συνεχώς, αλλά υπάρχουν κάποια κοινά σημεία. Ε, εν κατακλείδη, ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και αν κάποιος ε, δεν έχει επισκεφθεί την Κίνα τα τελευταία 3-4 χρόνια, ε, να, να πάτε οπωσδήποτε, γιατί αυτά που ξέρατε μέχρι τώρα δεν ισχύουν πια. Οπότε είναι σαν να μην έχετε πάει ποτέ. Σας συνιστώ να ξαναπάτε. Καλώ, θα το κάνουμε τόσο άλλο σε λίγες εβδομάδες. Επόμενο θέμα, επόμενο βήμα μάλλον της διαδικασίας είναι η συζήτηση της έκθεσής σου τον Απρίλιο και μετά θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Ε, είμαστε μέσα στο χρόνο για το επόμενο θέμα ε, που είναι η έκθεση του Δανιέλ Κάσπαρη. Έχετε το λόγο κύριε Κάσπαρη. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Μάρτιο του 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο κανονισμού επί του θέματος του πώς ακριβώς θα κατορθώσουμε να ανοίξουμε την αγορά των δημοσίων συμβάσεων. Στο Κοινοβούλιο ε, σκεφτήκαμε το θέμα για δύο περίπου χρόνια και κατόπιν τον Ιανουάριο του 2014 καταθέσαμε και ψηφίσαμε 85 τροπολογίες επί του θέματος στην Ολομέλεια. Για να παραμείνει το θέμα ανοιχτό, ε, δεν κλείσαμε όμως το όλο θέμα στην πρώτη ανάγνωση. Αυτό που ήταν εκνευριστικό ήταν ότι στο Συμβούλιο μετά δεν έγινε τίποτα. Το Νοέμβριο του 2014 υπήρξε μια συζήτηση προσανατολισμού στο Κοινοβούλιο και ε, αργότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τις εκλογές αποφάσισε τον Ιανουάριο του 2016 να καταθέσει στο Κοινοβούλιο πολύ τροποποιημένη πρόταση κανονισμού. Περίεργα όλα αυτά, διότι δεν έλαβε χώρα και τριμερή διάλογος. Ούτε καν υπήρξαν άτυπες συζητήσεις μεταξύ Κοινοβουλίου, Κομισιών και ε, Συμβουλίου και εγώ εξ γνωρίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρέπει και επιθυμεί να έχει τριμερή διάλογο ή να καταθέτει κάποιες δικές προτάσεις. Δεν έγιναν όλα αυτά. Τώρα έχουμε τροποποιημένο κανονισμό χωρίς, επαναλαμβάνω, να υπήρξαν έστω και άτυπες συζητήσεις ανάμεσα στους θεσμούς. Υπάρχει λοιπόν το εξής. Τι θα κάνουμε αφενός υπάρχουν κάποια σημεία όπου η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υιοθετεί τις προτάσεις του Κοινοβουλίου. Παραδείγματος χάρη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προβλέπονται διευκολύνσεις έχουμε το, την απομάκρυνση του περίφημου decentralized pillar, όπου η ιδέα είναι ότι οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες θα μπορούν να αποφασίζουν αν θέλουν να αποκλείσουν κάποιον αλλοδαπό επενδυτή ή όχι. Αυτό είναι ένα καλό βήμα. Κατόπιν υπάρχει το εξή. Η τροποποιημένη πρόταση υπαρχει το εξης ικανοποιεί κάποια αιτήματά μας και άλλα όμως τα αγνοεί πλήρως αυτά που είχαμε εκφράσει στην πρώτη ανάγνωση. Εμείς είχαμε μιλήσει για το περιβάλλον, για κοινωνικά θέματα που θα θέλαμε να εξεταστούν. Επίσης είχαμε εκφράσει την επιθυμία πέντε χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού να υπάρξει αναθεώρηση. Δυστυχώς τίποτα από αυτά και ε, επιτάχυνση της διαδικασίας που ζητήσαμε κατά την πρώτη ανάγνωση ούτε αυτή θα λάβει χώρα. Ποιον εδώ έκανε ένα μικρό τρίκ, δηλαδή είπε ότι τους εννέα μήνες τους κατεβάζει στους οκτώ μήνες ε, αντί να παρατείνει από τους 3 στους 4 μήνες. Συνολικά λοιπόν μιλάμε για 12 μήνες, ε, συμπαθητικό αυτό που προτείνει η Κομισιόν, αλλά μη μας θεωρείτε και χαζούς, το καταλάβαμε. Το τρίτο, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, προβλέπει επιπρόσθετα στοιχεία όπου πρέπει να σας πω ότι δεν ε, χάρηκα ιδιαίτερα. Το ένα είναι μηχανισμός προσαρμογής τιμών. Αυτό μου θυμίζει πολύ τα ε, εργαλεία του dumping, όπου το θέμα είναι να υπάρχει μια ε, αγορά, η αγορά καταστρέφεται, αλλά σε αυτό τον κανονισμό το θέμα δεν είναι να παραγωνιστούν στρεβλώσεις αγοράς, αλλά ο στόχος είναι να ανοίξουν άλλες χώρες τις αγορές τους δημοσίων συμβάσεων. Το θέμα δεν είναι να ε, δοθεί το μήνυμα ότι θέλουμε να αυξηθούν κάποιες τιμές, αλλά θέλουμε να πούμε σε άλλες χώρες, εμείς επιθυμούμε ανοιχτές αγορές, ανοιχτές αγορές για κρατικές προμήθειες, αν όμως μία χώρα χώρα, με συγχωρείτε, μετά από πολλές διαπραγματεύσεις δεν θέλει να ανοίξει την αγορά του, τότε ως έσχατο εργαλείο θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να κλείσουμε πλήρως την αγορά μας για ε, ενδιαφερόμενους από αυτό το κράτος. Εμείς όμως δεν το θέλουμε αυτό, θέλουμε οι αγορές μας να παραμείνουμε ανοιχτές. Αυτός όμως ο μηχανισμός προσαρμογής τιμών δεν έχει καμία απολύτω σχέση με τις δικές μας τις επιθυμίες. Θα κάνουμε λοιπόν το εξή ε, και έτσι πρέπει να καταλάβετε και να ερμηνεύσετε τις ε, τροπολογίες μας θέλουμε να πάμε πίσω ακριβώς σε αυτά που είχαμε αποφασίσει στην πρώτη ανάγνωση όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγνόησε παντελώς τις προτάσεις μας. Δεύτερον, ε, στα σημεία όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, καταθέτει νέες προτάσεις περί προσαρμογής τιμών, γι' αυτό το θέμα έχω προετοιμάσει κάποιες ε, τροπολογίες για να έχουμε ξεκάθαρη θέση. Θα ήθελα λοιπόν να ε, καλέσω όλους να ασχοληθούν με το θέμα. Γνωρίζουμε ότι βεβαίως και μεσολάβησαν οι ευρωεκλογές, γι' αυτό χρειαστήκαμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά τώρα πια νομίζω ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε να κλείσει το θέμα σε αυτή την θητεία του Κοινοβουλίου και γιατί όχι να ψηφιστεί το θέμα και μέχρι το τέλος του έτους στην Ολομέλεια. Λοιπόν, λοιπόν η καταληκτική ημερομηνία κατάθεση τροπολογιών είναι 21 Μαρτίου. Το Μάιο μπορούμε μάλιστα να ψηφίσουμε. Και επαναλαμβάνω, η δική μου η κατευθυντήρια γραμμή είναι πάμε πίσω, πίσω σε αυτά που είχαμε αποφασίσει κατά το παρελθόν. Και θα ήμουν ευγνώμων εάν οι συνάδελφοι μπορούσαν να δεχθούν τις τροπολογίες τις οποίες έχω καταθέσει. Χαίρομαι που θα ακολουθήσει η συζήτηση. Ευχαριστούμε και εμείς, λέει ο Πρόεδρος. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία όσον αφορά τις δυνατότητες που έχουμε για το αν θα ψηφίσουμε κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας ή όχι. Ο κύριος Σούστερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ αντικαθιστώ ε, τη συνάδελφα μου Ροτρίγκη Πινέντες και γι' αυτό θα διαβάσω την ομιλία στα αγγλικά. Η συμφωνία GPA έχει υπογραφεί μόνο από λίγα μέλη του ΠΟΕ. Το πεδίο εφαρμογή είναι περιορισμένο και οι περισσότερε αναδυόμενε οικονομίε δεν θέλουν να ενταχθούν. Η ευρωπαϊκή αγορά είναι ανοιχτή στο διεθνή ανταγωνισμό, αλλά πολλοί από του εταίρου μα διστάζουν να ανοίξουν τι δικέ του αγορέ. Επιπλέον, τα προστατευτικά μέτρα αυξάνουν σε πολλέ από τι αγορέ αυτέ. Για να αντισταθμιστεί αυτό το γεγονό, η ομάδα μου θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξασφαλίσει ε, μια ισοτιμία και ευκαιρίες αγοράς για τις εταιρείε μας. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι πρέπει να, υπά, στηριχθεί το μέσο που προτείνει η Κομισιόν γιατί αυτό μπορεί να ενισχύσει τη θέση μας στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και να ε, βελτιώσει τις συνθήκες πρόσβασης των, αγορών μας, ε, των εταιριών μας στις δημόσιες αγορές των χωρών αυτών. Δεν είναι εργαλείο προστατευτισμού αλλά είναι μια, ένας τρόπος να εξασφαλιστεί καλύτερη Παρ' όλα αυτά το IPI πρέπει να αποτελέσει εργαλείο αναλογικό, ε, αποτελεσματικό και κυρίως ρεαλιστικό σχετικά με το τι είναι εφικτό ε, στα πλαίσια της νομοθετικής διαδικασίας. Η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι ο κανονισμός να εγκριθεί και να τεθεί ενισχύει γρήγορα. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα κάποια στοιχεία των, της νέας πρότασης όπως η διαγραφή τον αποκεντρωμένου πυλώνα, την εφαρμογή το μέσο τη μείωση του γραφειοκρατικού άχθους και την αυξημένη διαφάνεια όσον αφορά τις έρευνες της Κομισιόν και τα ευρήματά τους. Το IPI είναι πρόταση του 2012 που προκάλεσε μικτές αντιδράσεις στο Συμβούλιο. Μια ομάδα κρατών μελών τότε θεώρησε τον κανονισμό προστατευτικό. Ε, αυτό οδήγησε σε αδιέξοδο επί χρόνια. Χαιρόμαστε που η νέα πρόταση της Επιτροπής προσπαθεί να περάσει, να σπάσει αυτό το αδιέξοδο. Γι' αυτό η ομάδα μας πιστεύει πιστεύει ότι πρέπει να λειτουργήσουμε επικοδομητικά και να προσπαθήσουμε να διευκολυνθεί η συμφωνία με το Συμβούλιο. Δεν θεωρούμε ότι αν επιστρέψουμε στη θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο το 2014 θα μας βοηθήσει να απελευθερώσουμε τα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε με βάση τη νέα πρόταση που έχει υποβάλει η Κομισιόν. Και υπό την έννοια αυτή θεωρούμε η επιστροφή στο κλείσιμο της αγοράς που προτείνει ο εισηγητής θα μας οδηγήσει σε νέο αδιέξοδο πλέον. Ε, σε έναν αυξανό όλο και περισσότερο προστατευτικό κόσμο θεωρούμε ότι το κλείσιμο αγοράς των δημοσίων αγορών μας δεν θα είναι καλή ένδειξη. Ε, το όσον αφορά το, το, μέτρο προσαρμογής της τιμής ε, ε, εντάσσεται εκεί. Τώρα είναι ευπρόσδεκτη πρώτα στο μιλητή να ληφθούν υπόψη τα περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων. Συμφωνούμε επίσης με τον εισηγητή για τον περαιτέρω μείωση του διοικητικού άχθους και να ενταχθούν όλο και περισσότερο περισσότερο ε, ε, τοπικές οντότητες στις διατάξεις του κανονισμού. Πρέπει να υπάρξει περισσότερη ευελιξία στο μέσο αυτών και να ε, θεσπιστούν διαφορετικά κατόφλια για τα δημόσια έργα και τις υπηρεσίες. 5 εκατομμύρια ως όριο δημοσίων έργων είναι πολύ, είναι πολύ ψηλό, ενώ για τα δημόσια έργα μπορεί να είναι πολύ χαμηλό. Τέλος, πρέπει να συμπεριληφθεί η δυνατότητα να μην εφαρμοστεί το μέσον αν θα οδηγούσε σε μονοπωλιακή θέση εντός του κλάδου. Η ομάδα μου έχει υποβάλει σχετικές τροπολογίες και είμαστε έτοιμοι, ε, ε, ε, ανοιχτοί απέναντι στον οσηγητή και τις άλλες ομάδες για να έχουμε μια επικοδομητική προσέγγιση ώστε να εγκριθεί ο κανονισμός. Ευχαριστώ. Καταπληκτικά. Η αίμα. Thank you. Um... Ευχαριστώ. Πριν κάνω τα σχόλιά μου για την ενημερωμένη αυτή επικαιροποιημένη πρόταση, ήθελα να, συνεχί... να συγχαρώ τον Ντάνιελ για το αξιόλογο έργο του σε ένα δύσκολο ζήτημα. Εμείς είμαστε κατά της, ε, του διεθνούς ε, ε, μέσου για τις δημόσιες συμβάσεις ε, και γιατί πιστεύουμε ότι κάτι θα μειώσει ε, ή θα περικόψει την οικονομική ανάπτυξη τώρα που τη χρειαζόμαστε περισσότερο και θα οδηγήσει τις ΗΠΑ στην υιοθέτηση ε, μέσων μέτρων αντιπερισπασμού. Βέβαια κάποιες αλλαγές έγιναν θετικές στην αναθεωρημένη πρόταση και κυρίως το ότι αφαιρέθηκε το θέμα του κλεισίματος ε, της Ευρωπαϊκής Αγοράς Δημοσίων ε, Συμβάσεων και παρόλο που υπάρχουν κάποια μέτρα προσαρμογής των τιμών δεν είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσουν τρίτες χώρες να ανοίξουν τις δικές τους αγορές δημοσίων συμβάσεων και μάλιστα αν δημιουργήσουμε φραγμούς στην είσοδο άλλων χωρών θα είναι αναμενόμενο και από τις τρίτες χώρες να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Επίσης, η γραφειοκρατία που θα χρειαστεί και οι εξιολογήσεις για να πληρωθούν τα κριτήρια για την επίκληση ενό τέτοιου μηχανισμού προσαρμογή τιμών είναι τόσο χρονοβόρα διαδικασία και τόσο δαπανηρή, ώστε θα χάναμε το ενδιαφέρον τρίτων χωρών ή το ενδιαφέρον των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Τα νέα προτινόμενα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάπως καλύτερα και σίγουρα καλύτερα από το πλήρε κλείσιμο τη αγορά, αλλά δεν συμφωνώ με τον ασυγητή γιατί ο εισηγητή προτείνει επαναφορά του αρχικού μηχανισμού ε, που προβλέπει περιορισμό ε, τρίτων χωρών από την αγορά δημοσίων συμβάσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως είμαστε υπέρ των τροπολογιών που προβλέπει αποκλεισμό των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων λιγότερων αναπτυγμένων χωρών και αναπτυγμένων χωρών από το πεδίο εφαρμογή της πρότασης. Και η επικεντρωμένη διαδικασία όπου κάποιος θα μπορούσε ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκλείσει την προσφορά αλλοδαπού επενδυτή ε, δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Θεωρούμε ότι έτσι θα αυξήσουμε τα αποτελέσματα του μέσου αυτού στις τρίτες χώρες, αποκλείοντας τις αρχικές αρνητικές συνέπειες της αρχικής πρότασης. Δεν θεωρούμε ότι είναι σκόπιμο ένα τέτοιο μέσο. Παρ' όλα αυτά συμμετέχουμε στη συζήτηση και θα συνεργαστούμε με τον εισηγητή και τους σκιώδης εισηγητές ε, για το θέμα αυτό. Και με πολύ προσοχή και στενά θα παρακολουθούμε την πρόοδο στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Η Φρεντερίκ. Ο Αρνό απουσιάζει γιατί ετοιμάζει την ε, προσγείωσή του στο Λουξεμβούργο, όπως ξέρετε. Είναι πολύ άσχολος. Θα μεταφέρω εγώ τις παρατηρήσεις του προς τον εισηγητή και την Επιτροπή. Καταρχήν θέλει να ευχαριστήσει τον Ντανιέλ Κάσπαρη για το σχέδιο έκθεσης. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Προστασίας του Καταναλωτού ανέδειξε τα προβλήματα ε, που περιέχει πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, δημιουργεί σοβαρέ ανησυχίε για το πώ θα επηρεάσουν την διεθνή αγορά. Καταρχήν, το βασικό του ε, μέλημα και ο βασικό του προβληματισμός είναι ότι από τη στιγμή που θα δημιουργήσουμε την νομοθεσία θα δημιουργηθούν προβλήματα στι ευρωπαϊκέ ε, επιχειρήσει, με την αύξηση τη γραφειοκρατίας. Για παράδειγμα, η πρόταση ω έχει μπορεί να ακυρώσει κοινέ αγορές ή να τις καταστήσει εξαιρετικά δύσκολες. Επίσης, το πεδίο εφαρμογή των ένδικων μέσων ε, είναι ασαφές. Ο Χάνο Τάκουλα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει το παιδί εφαρμογή και να δώσει κάποιες εξηγήσεις για το πώς θα ισχύσει με τρόπο ώστε να προστατεύει τις ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις. Γιατί φαίνεται ότι η πρόταση αυτή ανοίγει ακόμη περισσότερο την αγορά ε, περιορίζοντας τη δυνατότητα μέσων προσφυγής. Ε, το τελευταίο σχόλιο του κ. Τάκουλα αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της πρότασης. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να τις διευκολύνουμε για να ακολουθήσουν τις διαδικασίες. Επίσης, ε, σημαντικό είναι όταν οι εταιρείε αυτές αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, αυτό να μην περιπλέξει περαιτέρω τη δομή των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων. Ο Χάνου Τάκουλα πιστεύει ότι ε, καλό θα ήταν να καταθέσει κάποιες τροπολογίες και προσβλέπει σε αγαστή συνεργασία με τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές. Ευχαριστώ. Δεν φαντάζομαι ο ίδιος να καταθέσει τροπολογίες, δεν θα καταθέσει πια τροπολογίες αφού έφυγε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή που με προσκάλεσε να συνεργαστούμε. Το βρίσκω πολύ καλό. Να, σε αυτό το θέμα μπορούμε να συνεργαστούμε. Βέβαια αυτό σπάνια συμβαίνει, το να συνεργαζόμαστε εμείς σε αυτή την Επιτροπή. Κατόπιν τούτου θεωρώ ότι μπορούμε πράγματι να συμφωνήσουμε επ' αυτής της ε, έκθεσης γιατί ο παλαιός ε, κανονισμός ε, είχε επιβληθεί από την, στο, πνεύμα του Global Europe και του De Kucht. Εν όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει και πρέπει να σκεφτούμε μα τι το χρειαζόμαστε αυτόν τον κανονισμό. Αν δούμε λιγάκι ε, τη σχέση ενός κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε, σε σχέση με τον ΠΟΕ θα διαπιστώσουμε ότι ένας από τους λόγους ε, για αυτά που αποφάσισε η Κομισιόν είναι ότι η Κίνα και η Ινδία είχαν παλαιότερα το καθεστώς του παρατηρητή. Όμως η Κίνα παρουσίασε συγκεκριμένες απόψεις οι οποίες παλαιότερα απορρίφθηκαν από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, κατόπιν τούτου αυτός ο κανονισμός εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μακροοικονομικό πλαίσιο. Ένα άλλο θέμα το οποίο θέλω να προβάλλω εκ μέρους της ΓΚΟΕ είναι το εξής. Όσο καλό και αν είναι να ανοίξουμε αυτές τις ε, αγορές των ε, δημοσίων συμβάσεων. Υπάρχουν κάποια αγαθά για τα οποία δεν πρέπει να ισχύει πλήρες ε, κατεστώς απελευθέρωσης. Αυτό θυμάμαι όταν συζητάγαμε για τη ΣΕΤΑ και για άλλες σημαντικές συμφωνίες. Αν τα πάρουμε όλα σημείο προς σημείο και τα δούμε προσεκτικά, θα διαπιστώσουμε ότι αυτό που σας είπα έχει κάποια βάση. Προσβλέπω στη συνεργασία και ελπίζω να τα καταφέρουμε μια χαρά. Όλοι χαίρονται, λέει ο πρόεδρος. Όλοι είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ο Κρίστοφ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τον Ντάνιλ για την παρουσίαση. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση γιατί πραγματικά είναι ανοίγει μια νέα εποχή, στη, ένα νέο αντικείμενο στην ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική. Αν τα εμπόδια είναι πάρα πολύ ψηλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευρά άλλων, για την Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευρά, α σηκώσουμε και τα δικά μα. Έχει ψηλού δασμού, διαπραγματευόμαστε ή κατεβάζει ε, του δικού σου και ίσω να κατεβάσουμε και του δικού μα. Και με αυτό το μαγικό τρόπο. Τι θα γίνει. Ας δούμε την κοινή λογική για να δούμε αν η πρόταση της Κομισιόν ε, περνάει από τον έλεγχο της κοινής λογικής, το Υπολογίσαμε, με βάση αυτή την κοινή λογική, υπολογίζουμε ότι ας πούμε θα έχουμε νέα πρόσβαση σε αγορές αξίας 4 δις. Μέσω κάποιας ασαφούς λογικής στη σοφία τους μπόρεσαν να μας πούν ποιος θα ανοίξει ποια αγορά κατόπιν των απειλών που θα κάνουμε εμείς για το κλείσιμο των αγορών μας θα ήθελα να σας προκαλέσω να επιστρέψετε με άλλες προτάσεις που αφορούν δασμούς. Αν αυτό είναι μια νέα ευφύς λογική την οποία εισάγεται, να το κάνουμε. Αυτό λέω ότι δεν ισχύει προφανώς. Απλώς τα τέσσερα δίστα φαντάστηκαν για να πουλήσουν την πρόταση. Όλοι το ξέρουμε αυτό, το και εμείς και εκείνοι. Αλλά δούμε το κόστος λένε τώρα θέλουμε να προσαρμοστούν οι τιμές προς τα πάνω αν κάποιος δεν έχει παρκώς ανοιχτή αγορά. Και αυτό σημαίνει ότι εάν πρόκειται να αγοράσω ένα μηχάνημα ακτίνων χ, δεν θα επιλέξω αυτό που πρέπει από την τάδε χώρα ή αν το επιλέξω θα πληρώσω πιο ακριβά, θα αγοράσω λίγο πιο, μια, πιο, ένα μηχάνημα λίγο πιο ακριβό από την Κίνα, αν ανταυτού θα αγοράσω ένα αμερικανικό ή γερμανικό. Εγώ ισχυρίζομαι ότι αυτό σημαίνει ότι αφού το μηχάνημα θα είναι πιο ακριβό, κάποιος θα πρέπει να πληρώσει κάτι παραπάνω, αν προσαρμόζουμε τις τιμές προς τα πάνω. Αυτό κάνουμε το, κάνω αυτόν τον έλεγχο γιατί αν έχετε τη μαγική ικανότητα να προβλέψετε το κόστος και τα ωφέλη πρέπει να μπορείτε να προβλέψετε πόσο πιο ακριβά συνολικά για την Ευρώπη θα είναι αυτό. Πόσο θα κοστίσει αυτό. Λέτε δεν υπάρχει κόστος. Είναι αμεληταίο. Εντάξει. Πολύ ενδιαφέρον. Μην, πιστέψετε, μην το πιστέψετε. Είναι ασαφής λογική αυτό. Το δεύτερο που λέτε ότι δεν έχει κόστος είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος αντιπίνων αν προχωρήσουμε έτσι. Θα ήθελα η Κομισιόν να μην μιλήσει για την, ε, τις την νομοθετή των Ηνωμένων Όταν ο πρόεδρος Τραμπ κάνει την νομοθετησία του, να μην πείτε τίποτα. όταν λέτε ότι αυτό θα οδηγήσει σε αντίπεινα από, από άλλους, μην το λέτε πια. Αυτές είναι μία από τις προτάσεις που έχω δει από την Κομισιόν. Ούτε καν δεν περνάει το τεστ της κοινή λογικής. Να επιστρέψετε όταν θα έχετε το κόστος της πρότασης και θα μπορείτε να απαντήσετε πιστικά επί των ωφελών. Μέχρι τότε, ωραία κοιμωμένη καλύτερα. I have feeling that... Έχω το αίσθημα ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις εντός του ΕΛΚ. Απίστευτο υπάρχουν οι ριζοσπάστες και οι μετριοπαθείς. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, επόμενος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Κασπάρη για την έκθεσή του, την οποία και χαιρετίζουμε. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά καρπός διεξοδικής ε, μελέτης και συμμεριζόμαστε πολλές από τις ιδέες και τις προτάσεις σας. Για να μην πω και όλες. Ίσως όχι 100% αλλά σίγουρα στερνιζόμαστε τις περισσότερες. Και ήδη έχουμε συμπεριλάβει στην αναθεωρημένη μας πρόταση πολλές ε, συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είμαστε έτοιμοι για συνεργασία μαζί σας προκειμένου να διερευνήσουμε και άλλες ε, ε, προτάσεις για τη μείωση του γραφειοκρατικού άχθους και να διασκεδάσουμε και άλλες ανησυχίες που έχει επιτροπήσει και το Κοινοβούλιο. Τώρα, ποιο είναι το κυρίως θέμα εδώ. Το θέμα είναι ότι η ευρωπαϊκή αγορά είναι τεράστια και ανοιχτή, ενώ άλλες χώρες ουσιαστικά κλείνουν τις δικές τους αγορές αντί να τις ανοίγουν περισσότερο αναφέρθηκε ο νόμος «Αγοράζω Αμερικανικά» στις Ηνωμένε Πολιτείες, το Buy American Act. Αλλά υπάρχουν και άλλες τάσεις και πρωτοβουλίες ε, σε άλλες χώρες που είναι είτε ανοιχτές είτε κρυφίες προκειμένου να κλείσουν, να περιορίσουν την αγορά τους σε ξένους ε, ε, παράγοντες. Η αγορά δημοσίων συμβάσεων είναι τεράστια και μεγάλη ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της καινοτομίας, της υψηλής ποιότητας και των υψηλών προδιαγραφών. Τώρα, έχουμε δει και έχω διαπιστώσει και εγώ προσωπικά πόσο δύσκολη είναι η διαπραγμάτευση με τους εμπορικούς μας εταίρους για εμπορικές ε, συμφωνίες που στόχο έχουν το άνοιγμα των αγορών τους για τις, δημοσιε, για δημόσιες συμβάσεις. Ενώ θεωρούν ως δεδομένη την ανοιχτή ε, ευρωπαϊκή αγορά δημοσίων συμβάσεων, ενώ ήδη είναι πρόθυμοι να ανοίξουν τις δικές τους αγορές δημοσίων συμβάσεων. Ενώ ε, τα πλεονεκτήματα είναι ήδη απτά και ορατά. Όταν διαπραγματευόμαστε με τον Καναδά και την Ιαπωνία, και μόνο η αμυδρή πιθανότητα της παρουσίασης της ε, πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ακόμη σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε ακόμη και μόνο η ύπαρξη της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει οδηγήσει ε, σε μία σημαντική συμφωνία με τον Καναδά και την Ιαπωνία σε ό,τι αφορά τους κανόνες αλλά και την πρόσβασή μας στις αγορές δημοσίων συμβασεών τους. Ήδη λοιπόν έχουμε συγκεκριμένα πτά παραδείγματα. Θετικά βέβαια αυτή η ε, λανθάνουσα απειλή δεν μπορεί να υπάρχει για πάντα και διαπιστώνουμε στις διαπραγματεύσεις μας ότι ότι οι εταίροι μας έχουν αμφιβολίες. Δεν ξέρω αν είναι σοβαρή η πρόταση, αν θα υλοποιηθεί ή όχι. Πιστεύουμε πάντως ότι η πρωτοβουλία αυτή και η συγκεκριμένη πρόταση πρέπει να υιοθετηθούν το συντομότερο δυνατόν, γιατί δεν είναι πρόταση ε, προστατευτική και αυτό είναι σημαντικό να το τονίσουμε. Ούτε λέμε ότι πρέπει σώνει και καλά να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέσο, να το χρησιμοποιούμε μάλλον συνεχώς. Απλώς αυτό, αυτό το μέσο είναι η ίστατη λύση, η έσχατη λύση. Θέλουμε προηγουμένως ε, να διαπραγματευτούμε με όλες τις ε, χώρες που κλείνουν τις αγορές τους και που δεν επιτρέπουν στις επιχειρήσεις μας να λάβουν μέρος στις, ε, στους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων και να αξιοποιήσουν τέτοιες δυνατότητες. Όπως είπα λοιπόν, Είμαστε έτοιμοι να διερευνήσουμε και άλλες προτάσεις. Και αυτό που βλέπουμε και συζητούμε είναι πώς θα εφαρμόσουμε εμπράκτος και ουσιαστικά την υπάρχουσα νομοθεσία μας. Γιατί τα περιβαλλοντικά, τα κοινωνικά και άλλα θέματα και άλλες πτυχές μπορούν ήδη να εφαρμοστούν ε, και υπάρχουν στο ισχύον μας νομικό πλαίσιο. Μάλιστα, από τη στιγμή που τα ευρωπαϊκά αγαθά, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πληρούν υψηλότερες προδιαγραφές ε, και προσφέρουν προϊόντα που πληρούν κοινωνικές, περιβαλλοντικές ε, και άλλες πτυχές, αυτό δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε επιχειρήσεις μας. Και δεν χρειαζόμαστε αυτό το μέσω διεθνών προμηθειών για αυτό το λόγο. Αυτό που Ο σκοπός για τον οποίο χρειαζόμαστε το IPI, αυτό το μέσο για τις διεθνεί προμήθειες, είναι για να δώσουμε κίνητρα στους εμπορικού μας εταίρου να καθίσουν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων μαζί μας και να διαπραγματευτούμε από κοινού κανόνες για την πρόσβαση στις αγορές δημοσίων συμβάσεων ε, με δίκαιη και ισότιμη βάση. Αυτά και είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία. Εννοείται. Ο κύριος Κάσπαρη. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι στη συζήτηση κατέστη σαφέ, ε, ποιε ε, είναι οι ευκαιρίε που μπορεί να προσφέρει αυτό το μέσο αλλά και ποιοι κίνδυνοι. Ε, όσον αφορά τους κινδύνους, ο Κρίστοφ ε, επισήμανε αυτούς τους κινδύνους. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο ε, είναι απόλυτα σαφές. Εμάς, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ε, άλλες χώρες να ανοίξουν τις αγορές τους για τις δημόσιες συμβάσεις και όχι να τις κλείσουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο αρχικό της σχέδιο είχε κάποιες ε, διατάξεις που όμως εμάς δεν μας ικανοποίησαν. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή αυτός ο κανονισμός, όλες οι εθνικές νομοθεσίες που δίνουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κλείσουν οι αγορές, όλες αυτές οι εθνικές νομοθεσίες καταπίπτουν. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν θέλουμε να αρθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση. Εμείς θέλουμε να ανοίξουν οι αγορές και θέλουμε με τη θέση σε εφαρμογή αυτού του μέσου να ανοίξουν περισσότερο οι αγορές στην Ευρώπη, όχι να κλείσουν. Σας είπα με το ότι θα αρθούν και θα πάψουν να ισχύουν οι εθνικές νομοθεσίες. Αλλά τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι σήμερα στις ε, διαπραγματεύσεις σε διεθνές επίπεδο το όλο θέμα δεν προχωράει. Εμάς, επαναλαμβάνω, δεν μας ενδιαφέρει να κλείσουμε αγορές αγορές, ε, μας ενδιαφέρει να ανοίξουμε αγορές. Και όποιος δεν συμφωνεί θα πρέπει τουλάχιστον να ξέρει ότι στο μέλλον ε, οι ευρωπαϊκές αγορές θα είναι πιο κλειστές για εκείνον. Ε, θέλω να δω τι θα γίνει με τις τροπολογίες και τι θα γίνει τελικά στην ψηφοφορία στην Ολομέλεια, καταληκτική μερομηνία τροπολογιών, λέει ο Πρόεδρο, 21η Μαρτίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε στο επόμενο θέμα, στο υπαριθμό 23. Είναι η... Είναι η ειναι εφαρμογη των εμπορικών, εμπορικών προτιμήσεων σε σχέση με την επισήμανση προϊόντων που προέρχονται από τους οικισμούς. Είναι ένα θέμα που συζητείται από καιρό. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα που αναφέρεται ότι προέρχονται από το Ισραήλ, προέρχονται όντως από το Ισραήλ και όχι από οικισμούς, παράνομους οικισμούς εκτός Ισραήλ. Και εδώ υπάρχει ένα σημείωμα από την Κομισιόν. Για κάποιους λόγους δεν λειτουργεί, δεν εφαρμόσεται και χρειάζονται διευκρινήσεις. Ο κύριος Φερνάντο Περό και Ντεπίνικ, ο οποίος ελπίζω να είναι εδώ, Και πριν του δώσω το λόγο, θα δώσω το λόγο στην Μαρία Ρενό, την εισηγητριά μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως συνήθως στην Επιτροπή αυτή παρακολουθούμε όλες τις εμπορικέ συμφωνίες. Δεν, θέσα, δεν ασχοληθήκαμε με την Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ εδώ και πολλά χρόνια, αλλά πρόσφατα ακούστηκαν πολλά σχετικά με το ότι δεν τηρείται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θεωρώ λοιπόν λογικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέσει στην Κομισιόν ερωτήματα, παρότι γνωρίζουμε ότι η υλοποίηση ε, συμφωνία Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ με όλα τα υποερωτήματα είναι οριζόντιο θέμα στην Κομισιόν και εμπλέκονται πολλές γενικές διευθύνσεις και άρα οι ε, απαντήσεις δεν είναι άνετο να δοθούν και δεν είναι ε, συγκεκριμένες ε, σε ερωτήματα που, δίνει, που θέτει συνήθως το Κοινοβούλιο. Η Συμφωνία Σύνδεσης κατά την άποψή μου συνολικά και έχει βαλάβει θέση και το Κοινοβούλιο πρέπει να αξιολογηθεί γιατί όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε ο, ο, μηχανισμός που τον αφορά και συγκεκριμένα οι εμπορικές προτιμήσεις που παραχωρούνται στα Ισραηλινά προϊόντα ε, έχουν, αφορούν μια νομοθεσία που δεν τηρείται. Το Σεπτέμβριο του 2017 ε, δημοσιεύτηκαν πολλά άρθρα που λένε ότι έμπαιναν σε στο ευρωπαϊκό έδαφος ε, υπό εμπορικές προτιμήσεις προϊόντα των επικισμών αυτών. Ε, αυτό έπρεπε να επαληθευτεί. Ε, μετά από λίγες εβδομάδες μέσω της αντιπροσωπείας της στο Τελαβίβι η Κομισιόν διαπίστωσε ότι ήταν τεχνικά αδύνατον να ελεγχθεί η προέλευση και να γίνει διαφοροποίηση από την, με την ε, θεσμοθέτηση του ταχυδρομικού κώδικα και έγινε μια προσπάθεια συνεργασίας με, εργασίας εναλλακτικές λύσεις αλλά οι Ισραηλινές αρχές ε, ήταν διστακτικές να τροποποιήσουν το σύστημα του ταχυδρομικού κώδικα. Ε, κατόπιν είχαμε το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών του Δεκεμβρίου που καλεί τα κράτη να ε, θεσπίσουν πολιτική διαφοροποίηση μεταξύ του Ισραήλ εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων του και των κατεχωμένων εδαφών από το 1967. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό και βάσει αυτών των διαπραγματεύσεων διαπιστώσεων είναι, ε, είναι, μοιάζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραβιάζει την ίδια της νομοθεσία όσον αφορά τη Συμφωνία Σύνδεσης. Έχω λοιπόν κάποιες ερωτήσεις. Πρώτον, ε, αναγνωρίζει σήμερα η Κομισιόν εδώ ότι τα προϊόντα των, των επίκων ε, μπαίνουν στην Ένωση με προτιμησιακό καθεστώς, με προτιμησιακούς δασμούς. Πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα είναι το άρθρο 79 της Συμφωνίας Σύνδεσης που επιτρέπει να ληφθούν μέτρα αν το ένα μέρος θεωρεί ότι το άλλο μέρος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του στα πλαίσια της συμφωνίας. Γιατί λοιπόν ε, ε, αυτή η κατάσταση διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια χωρίς κάποιο μέτρο, γιατί το Κοινοβούλιο δεν ενημερώθηκε για την κατάσταση αυτή, ενώ έγιναν τακτικά οι συνεδριάσεις παρακολούθησης. Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των προϊόντων αυτών που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι Όντω υπάρχουν τέτοια προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά. Τα προϊόντα που περνούν από τα τελωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωσης ή τα ποσά των δασμών που ε, έχουν έρθει για να δείξουμε ότι έχουν ε, επωφεληθεί από αυτό το καθεστώ ε, τα προϊόντα από αυτού του οικισμούς. Το Νοέμβριο του 2015 ε, ε, δημοσιεύτηκαν κάποια στοιχεία και ρώτησε προς την Κομισιόν. Μπορεί να ζητήσει, να απαιτήσει από τα κράτη-μέλη Κομισιόν μια αξιολόγηση της ε, ερμηνευτικής ανακοίνωσης για τα προϊόντα αυτά σε σχέση με το τι κάνουν τα κράτη-μέλη για να συμμορφωθούν με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πέμπτη ερώτηση. Κάποια από τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι αυτή η ερμηνευτική ανακοίνωση που αφορά τα προϊόντα δεν είναι δεσμευτική, ενώ πρόκειται για μια ερμηνεία του ευρωπαϊκού δικαίου απέναντι στους καταναλωτές. Ποια η ποια είναι η αντίδραση Κομισιόν από αυτού. Και τέλος, στη διάρκεια των διαφόρων συναντήσεών μου διαπίστωσα ότι υπάρχουν πολλές σκιές ζώνες ε, ε, μη ξεκάθαρες όσον αφορά την ερμηνεία. Δηλαδή η προέλευση αφορά και το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλαγή της προέλευσης από τον διανομέα αρκεί ή θα πρέπει αυτός να αναφέρει στον εξαγωγέα ε, την, διαφορά, την διαφορετική προέλευση. Επιπλέον υπάρχουν και ε, στοιχεία που πρέπει να δοθούν στα κράτη-μέλη για να βοηθηθούν στην συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εν κατακλεί το 2012 το ε, Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ε, εκτίμησε ότι οι εξαγωγέ των επικισμών αυτών είναι περίπου 230.000 ευρώ το μήνα. Επιπλέον, οι εξαγωγέ των Παλαιστινίων εκτιμώνται σε περίπου 17 εκατομμύρια το χρόνο. Συχνά λοιπόν μα λένε ότι οι εξαγωγέ από τι περιοχέ αυτέ που εποφελούνται από αυτέ τι περιοτιμησιακές συνθήκε, είναι πάρα πολύ λίγε. Αλλά 230.000 ε, σε σχέση με 17 εκατομμύρια το χρόνο από του Παλαιστινίου, πράγματι είναι πολύ πολλά προϊόντα τα οποία εξάγονται παράνομα επειδή αποφελούνται ε, από προτιμησιακού. δασμούς. Δεν θέλω να κάνω σύγκριση που να είναι αδικαιολόγητη, αλλά δουλεύουμε και για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καθόρισε κάποιους κανόνες λέγοντας είτε ότι τα προϊόντα αυτά από τις ψυχισμούς δεν μπορούν να μπουν με ε, προτιμησιακού δασμούς ή αν έρθουν θα πρέπει να ταυτοποιούνται και να μην υποφελούνται από αυτέ τι προτιμήσεις. Αλλά ε, εδώ δεν έχουμε την ίδια κατάσταση με, το, με αυτά που ισχύουν στο Μαρόκο και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι επίγον, επίγον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει τα ερωτήματα του Κοινοβουλίου επαρκώς ώστε να αποφύγουμε να έχουμε προβλήματα με το σύνολο της συμφωνίας με το Ισραήλ γιατί τότε θα ήταν σοβαρό και για τους Ευρωπαίους αλλά και για το Ισραήλ και θεωρώ ότι θα ήταν ενδιαφέρον να μας δοθούν οι απαντήσεις για να αποφύγουμε τη σύγκρουση τους επόμενους μήνες. <clears throat> Ο Γιούλιο Βίνκλερ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Διαβάζω τις σημειώσεις Ραμόνα Μανέσκο που είναι αρμόδια για το θέμα αυτό. Εγώ απλώ παρουσιάζω τη δική τη άποψη. Τα τελευταία χρόνια είχαμε πολλέ συνεδριάσει για το θέμα αυτό και έχει περάσει αρκετό χρόνο από τότε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το ερμηνευτικό σημείωμα για την ετικετοθεσία, τη σήμανση των προϊόντων των επικισμών. Θα μπορούσαμε να σταθούμε στα εξή σημεία τώρα. Καταρχήν, η υπάρχουσα νομοθεσία λειτουργεί στην πράξη ή όχι. Ε, μήπως α, απαιτεί δυσανάλογες ε, προσπάθειες ε, για να γίνει λειτουργική, οπότε θα πρέπει να επέμβουμε και να την τροποποιήσουμε για να γίνει πιο λειτουργική. Τι επίπτωση έχει στην ειρηνευτική διαδικασία και στην καθημερινότητα των πολιτών ε, στα εδάφια αυτά και απότερο σκοπός κάθε νομοθετικής προσπάθειας είναι να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών και εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά την πρώτη ερώτηση, διαπιστώνω ότι Ακόμη και οι νομοθέτες δεν αντιλαμβάνονται πλήρως ε, τις διατάξεις που ισχύουν για τη σήμανση των προϊόντων από τους επικισμούς. Ε, η σήμανση δεν σημαίνει απαγόρευση. Τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να εισάγουν προϊόντα από τους επικισμούς αρκεί να επισημαίνονται σωστά, ε, επισημαίνεται σωστά η προέλευση. Ως προς τη δεύτερη ερώτηση σε ό,τι αφορά τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα της νομοθεσίας, γιατί ε, πειράζει αρνητικά και τις θέσεις απασχόλησης και την κατάσταση του Παλαιστινιακού πληθυσμού. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή των Παλαιστινίων και θέλουμε να στηρίξουμε την Παλαιστινιακή Αρχή και την ειρηνευτική διαδικασία. Επίσης, ε, ε, η πολλές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα κατεχόμενα είναι παλαιστινιακές, οπότε το εμπάργο, ο εμπορικός αποκλεισμός των προϊόντων από τα κατεχόμενα δεν βοηθάει τους Παλαιστινίους, το αντίθετο. Επονομεύει την απασχόληση στις περιοχές αυτές. Επίσης, ε, θέλουμε και οι Παλαιστίνοι να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, τη βοήθεια και συνδρομή μας. Αυτό είναι με των δημοκρατικών μας προσπαθειών στην Μέση Ανατολή και από κοινού με το Ισραήλ θα πρέπει να συνεργαστούμε με την Παλαιστινιακή Αρχή για την ανάπτυξη της Παλαιστινιακής οικονομίας. Γιατί νομίζω ότι αυτή θα είναι η καλύτερη βάση για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Αυτά θα έλεγε η Ραμόνα Μονέσκου. Ο κύριος Μπάναμον από το ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ECR με αναγνωρίζει ότι η πολιτική τη σήμανση των ε, προϊόντων από τους επικισμούς δεν αντιστοιχεί με εμπορικό αποκλεισμό των Ισραηλινών προϊόντων, παρόλα αυτά στιγματίζει χωρίς λόγο τα Ισραηλινά προϊόντα. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι μόνο το 1% των Ισραηλινών προϊόντων προέρχονται από τα υψίπεδα του Γκολάν και τη Δυτική Όχθη. Ε, ήδη μάλλον έχουμε αποκλείσει τις εξαγωγές ε, εισαγωγές των προϊόντων από τις ε, προτιμησιακές ε, διατάξεις της συμφωνίας με το Ισραήλ. Πάντως, ε, αυτό το ερμηνευτικό σημείωμα υποτίθεται έχει στόχο την, τις για προστασία του καταναλωτού και λέει ότι όταν είναι, είναι υποχρεωτική η σήμανση της προέλευσης εφόσον η παράληψη της πληροφορίας αυτής παραπλανεί τον καταναλωτή για την πραγματική προέλευση του προϊόντος. Θεωρούμε ότι συνιστά διάκριση ει βάρο του Ισραήλ. Γιατί δεν εφαρμόζουμε κάτι τέτοιο και για τη Δυτική Σαχάρα, για παράδειγμα. Γιατί ουσιαστικά μια τέτοια διάταξη απομονώνει το Ισραήλ ή προσβάλλει τους μετριοπαθείς Ισραηλινούς που είναι υπέρα του συμβιβασμού και ουσιαστικά ενισχύει τις ε, ριζοσπαστικές, πιο ριζοσπαστικές ε, παλαιστινιακές θέσεις. Ε, και σίγουρα η ερευνητική διαδικασία θα υπονομευθεί από την απώλεια θέσεων απασχόλησης ε, στα εδάφια αυτά. Γιατί νομίζω ότι με τέτοια λύση δεν βλάπτει μόνο τους Ισραηλινούς, αλλά και τους Παλαιστινίους κυρίως, γιατί ε, κλείσιμο εργοστασίων στα κατεχόμενα οδήγησε σε απώλεια 500 θέσεων εργασίας Παλαιστινίων. Έτσι θα βοηθήσουμε την ενευτική διαδικασία. Αντίθετα, έτσι δηλητηριάζουμε ε, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Και είναι υπεραπλουστευτική ε, μια τέτοια πρόταση και είναι παράλογη αυτή η οριζόντια σήμαση. Ουσιαστικά υποδαβλίζει τη σύγκρουση αντί να την ε, αμβλύνει. Δεν νομίζω ότι είναι σωστή μια τέτοια πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρους της ΓΚΟΕ, η κυρία Σάντσες. Ευχαριστώ. Το Νοέμβριο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τι κατευθυντήριε γραμμές για τα εισαγόμενα προϊόντα από παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Οι κατευθυντήριε γραμμέ είναι σαφεί. Τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα προέρχονται από τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα, τα υψίπεδα του Γκολάν και τη Δυτική Όχθη, δηλαδή από τα κατεχόμενα, από τα δάφη που, στα οποία εισέβαλε το 67 το Ισραήλ, δεν πρέπει να, ε, θέτουν, να έχουν σήμα προϊόν Ισραήλ ε, και μάλιστα οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών στην Παλαιστίνη αλλά και οι διεθνείς οργανώσεις ε, διαβεβαιώνουν ότι τέτοιες διατάξει δεν εφαρμόζονται και παρόλο που τα εισαγόμενα αυτά προϊόντα αφορούν μόνο το 1% των εισαγωγών, δεν νομίζω ότι από τη στιγμή που παραβιάζεται το διεθνέ δίκαιο θα πρέπει να μένουμε σαν ποσοστά των παραβιάσεων. Θεωρείτε ότι οι Ισραηλινέ αρχέ τηρούν τι υποχρεώσει τικετοθεσία επισήμα και πραγματικά αναφέρουν την ε, γεωγραφική προέλευση των, προϊόντων που εξάγουν. Πώ εφαρμόζονται τα, πώς τα κράτη-μέλη τι κατευθυντήριε γραμμέ, και πώς εξασφαλίζεται την τήρηση αυτών των υποχρεώσεων από το Ισραήλ, γιατί η τήρηση των υποχρεώσεων αυτών δεν είναι μόνο εμπορικό θέμα, αλλά πολιτική υποχρέωση και από τη στιγμή που δεν γίνονται σεβαστές οι κατευθυντήριες γραμμές, ουσιαστικά ε, επιτρέπουμε στο Ισραήλ να παρακάμπτει όχι μόνο ε, την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Και γινόμαστε συνένοχοι σε αυτό. Επαναλαμβάνω, τα υψίπεδα του Γκολάν, η Δυτική Όχθη και η Ανατολική Ιερουσαλήμ είναι κατεχόμενα εδάφια από το Ισραήλ και θα πρέπει να απαιτούμε το σεβασμό του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το EFTD τώρα, ο κύριος Ντάρτμουθ φαντάζομαι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, ο αξιότιμος συνάδελφος Κέβιλ Καμελμπάνεμαν έδωσε ε, μια πολύ ξεκάθαρη παρουσίαση της υπόθεσης. Δεν θα προσπαθήσω να το μιμηθώ. Ένα θέμα θέλω να επισημάνω στους συναδέλφους, ότι το παράδειγμα της Δυτικής Σαχάρας είναι πολύ χαρακτηριστικό. Θέλω να επισημάνω ότι η πρόταση αυτή, και ελπίζω να είναι απλώς μια πρόταση, γιατί δεν μου ακούγεται απλώς ως πρόταση. Είναι αντιισραηλινή και θα στηριχθεί από αυτούς που είναι κατά του Ισραήλ. Αυτό δεν, είναι, δεν έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Δεν είναι αυτή μια κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε κάτι που ε, είναι ουσιαστικά νέο παρόλα όσα λέγονται. γιατί αυτό θα γίνει αντιληπτό ότι στρέφεται κατά του Ισραήλ. Και προτείνω στους συναδέλφους και στην Κομισιόν να το ξανασκεφτούν. Το προτείνω εμφατικά. Ευχαριστώ. Θέλω να επαναλάβω αυτά που είπε ο Γιούνις Μπίτλι. Βίνκλερ. Το να μποϊκοτάρουμε προϊόντα στη Γάζα, της Γάζας ή στη Δυτική Όχθη που εξάγονται μέσω του Ισραήλ δεν στηρίζει την ειρηνευτική διαδικασία. Απλώς καθιστά φτωχότερου τους κατοίκους των περιοχών. Όχι μόνο δηλαδή είναι υποκατοχή, αλλά γίνονται και φτωχότεροι. Και αυτό ε, δεν είναι καλή ιδέα. Αυτό που με προβληματίζει εδώ είναι ότι αυτή η συζήτηση έχει γίνει επανειλημμένος και ξέρω ότι υπάρχει μια αιμονή με τη συγκρουση σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων. Αλλά μας διαφεύγει η ουσία. Το γεγονός ότι το Ισραήλ είναι μια προηγμένη οικονομία, δημοκρατία, στενός φίλος της Ευρώπης και ενοχλεί περισσότερο από την παλιά ανεπαρκή συμφωνία σύνδεσης. Θα πρέπει να βάλουμε κάτι περισσότερο που να περιλαμβάνει τις υπηρεσίε, τη μεταφορά δεδομένων, την θεσμική συνεργασία που θα ωφελήσει και τις δύο πλευρές, και το Ισραήλ και την Ευρώπη. Σήμερα έχουμε ε, διαπραγματευτεί και συνάψει με την Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία πολύ πιο προχωρημένες συμφωνίες. Και ο κόσμος λέει άλλη υπόθεση του Ισραήλ διαπραγματευόμαστε με το Μαρόκο και την Τινησία, κάνουμε συμφωνίες επενδύσεων με την Κίνα και ξέρω ότι ο κόσμος έχει μια ειδική σύγκρουση με το Ισραήλ, αλλά για σκεφτείτε σε σύγκριση με την Κίνα τι γίνεται. Ως εκ τούτου, το λογικό που θα έπρεπε να κάνουμε θα ήταν να σταματήσουμε να κοιτάζουμε μόνο το εμπόριο με το Ισραήλ από μέσα από τη σκοπιά της συγκεκριμένης σύγκρουσης και να δούμε την ευρύτερη εικόνα το τι μπορούμε να κάνουμε για να ωφεληθεί και η Ευρώπη και το Ισραήλ μέσω μιας νέας πιο προχωρημένης συμφωνίας σύνδεσης. Η κυρία Μαργαρίτα Άουκ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής ε, της Αντιπροσωπής με την Παλαιστίνη. Ναι, λέτε να ξεκινήσουμε δεν μας νοιάζει ε, δεν μας νοιάζουν οι νόμοι. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για διεθνές δίκαιο. Είναι κάτι που υπάρχει, ε, δεν είναι κάτι το καινούριο, 50 χρόνια από τότε που η, έγινε η κατοχή. Και ακούω εδώ τον κόσμο να λέει ότι θα ήταν λίγο καλύτερα να ξέρω εγώ τι για το θέμα της κατοχής δεν συνάδει με την πολιτική της Ένωσης, με το Κοινοβούλιο, με αυτό που επανειλημμένως υπόθηκε. Για να είμαστε σαφείς, εξακολουθούμε να έχουμε τους κανόνες μας. Και θα πω, εκπλήσωμε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για την επισήμανση δεν παρακολουθούνται από την Κομισιόν. Ω θεματοφύλακα των, συνθήκων η Κομισιόν θα έπρεπε να φροντίσει και όχι να κατηγορεί τα κράτη-μέλη ότι δεν είναι σε θέση ότι μπορούν να τηρήσουν του κανόνε, Να εξασφαλίσει ότι υπάρχει σωστή επισήμανση από το Ισραήλ με του κωδικού και να μην προσφέρει προτιμησιακό καθεστώς. Αυτό το πολύ ωραίο μπουκάλι κρασί παράγεται στα υψώματα του Γκολάν, μπαίνει στι Βρυξέλλες και λέει κρασί Ισραήλ. Αυτό είναι παράνομο είναι παράνομο. Αυτό είναι ε, ψευδείς πληροφορίες προς τον καταναλωτή. Δεν είναι Ισραηλινό, είναι παράνομο και δεν θα πρέπει να απολαμβάνει προτιμησιακού καθεστώτος. Θα πρέπει η Κομισιόν άμεσα να αρχίσει να ανταποκρίνεται σε αυτό που εννοούμε όταν λέμε συμμόρφωση εδώ. Και αν τα κράτη-μέλη δεν τηρούν τους νόμους να επισημαίνεται αυτό. Μπορώ να πω πολλά από αυτού. Ελάχιστα μέσα έχουμε, αν δεν θέλουμε να κάνουμε πραγματικό μποϊκοτάζ. Έχουμε όμως μέσα νομικά. Αν θέλουμε να στερήσουμε τον εαυτό μας από τα μέσα αυτά και να πούμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε κατευθείαν σε γενικό μποϊκοτάζ, δεν συμφωνώ. Εγώ αντιμετωπίζω οτιδήποτε δεν είναι νόμιμο εδώ. Υπάρχει η γενική πρόταση ότι «Α, κοιτάξτε, δεν μας ενδιαφέρουν οι νόμοι». Ε, θα κάνουμε ό,τι θέλουν οι φίλοι μας, μας ε, πιέζουν, γίνεται lobbying κλπ. Και τελικά θέλω να πω, α, όχι, πρέπει και στατιστικά στοιχεία να συγκεντρώσουμε. Πόσα, έρχονται, πόσα προϊόντα έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τους πικρισμούς αυτούς, από, από αυτά τα εδάφη. Και τέλος, θέλω να αναφερθώ πώς κάνατε και εσείς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με το ε, ψήφισμα 2334 πριν από 1,5 περίπου χρόνο και τώρα το διεθνές δίκαιο προβλέπει ότι πρέπει να κάνουμε διαφοροποίηση που είναι πολύ πιο δύσκολο θέμα από ότι αυτό, αυτή η επισήμανση εδώ. στις τράπεζες, στην παιδεία, στις διάφορες αρχές, γιατί είναι θέμα νομιμότητας. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν υπέρ αυτού. Ακόμα και όμως αν, αν καταψήφισε κανείς κάτι το οποίο εγκρίθηκε εξακολουθεί να ε, είναι νόμος αυτό το να στείλουμε ένα σήμα στην μόνη δημοκρατία της περιοχής. Τι είναι αυτό. Το ότι δεν ε, τηρούνται οι νόμοι δεν είναι ότι καλύτερο μπορούμε να δείξουμε. Ο καλύτερος τρόπος είναι να βρεθούν ειρηνικοί τρόποι να επιτευχθεί ο κοινό μας στόχος, ελπίζω να συμφωνούν όλοι, ότι θα οδηγηθούμε σε μια ε, λύση δύο κρατών στα διεθνή σύνορα η μόνη ελπίδα μας είναι να είμαστε αξιόπιστοι και να ζητήσουμε αυτή τη στιγμή από την Κομισιόν τουλάχιστον να οδηγήσει σε τήρηση αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών και να εξασφαλίσει ότι δεν θα χορηγείται αυτή η προτιμησιακή μεταχείριση προς αυτά τα προϊόντα που θεωρείται ότι είναι από το Ισραήλ ενώ σαφώς δεν είναι. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που έγινε και η συζήτηση. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Εγώ θα εστιάσω στα ερωτήματα που ετέθησαν και αφορούν στην εφαρμογή των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και στη Συμφωνία Σύνδεσης. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι προφανώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να σέβεται πλήρως ε, την νομιμότητα την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να εφαρμόζονται οι συμφωνίες σύνδεσης με το Ισραήλ που αφορούν βέβαια μόνο στο ε, αναγνωρισμένο κομμάτι του Ισραήλ που σημαίνει ότι όλα τα άλλα προϊόντα τα οποία προέρχονται από περιοχές εκτός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων του Ισραήλ δεν μπορούν να εισέρχονται νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το καθεστώς προτιμήσεων, δηλαδή με μηδενικούς ε, δασμολογικούς συντελεστές. Εδώ θέλω όμως να κάνω μια διαφοροποίηση ανάμεσα στη σήμανση της προέλευσης και τη σήμανση για τα τελωνία, για τελωνιακούς σκοπούς. Αυτό είναι σημαντική διαφοροποίηση τα προϊόντα για να αποφελούνται από τις προτιμήσεις πρέπει να καλύπτουν τις ε, απαιτήσει ε, περί προέλευσης ε, που αναφέρονται στη συμφωνία με το Ισραήλ που σας λέω και πάλι μιλάμε για τα αναγνωρισμένα σύνορα του Ισραήλ και αποκλείονται, ξερούνται τα κατεχόμενα. Αυτό είναι απόλυτα σαφές τελείως διαφορετικό θέμα είναι κατά πόσον ένα προϊόν το οποίο εισάγεται ας πούμε από τα κατεχόμενα το οποίο μπορεί να εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει απαγόρευση το μόνο που ισχύει είναι ότι αυτά τα προϊόντα από τα κατεχόμενα δεν μπαίνουν με προτιμησιακό καθεστώς, μπορούν να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όπως διευκρινίστε στις κατευθυντήριες γραμμέ του 2015, δεν μπορούν να φέρουν την ετικέτα Made in Israel ή προέλευση Ισραήλ. Αυτό είναι παράνομο. Το πώς ελέγχονται όλα αυτά διαφέρει. Αφενός πρέπει να ξέρουμε τι κάνουν τα τελωνία στα σύνορα. Τα τελωνία ελέγχουν το κατά πόσον τα προϊόντα έχουν ετικέτα όπου να αναφέρεται ταχυδρομικός κωδικά που να αντιστοιχεί σε ε, κατεχόμενα εδάφη. Αυτό το έχει συμφωνήσει, το έχει δεχτεί και το Ισραήλ ότι στην ονομασία προέλευσης, στη δήλωση προέλευσης, θα πρέπει να αναφέρεται η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Άρα δηλαδή τα τελωνία βλέπουν κατά πόσον ε, υπάρχει κώδικας ε, που αν ο κώδικας αυτός είναι αποκατεχόμενα δεν ισχύουν οι ε, προτιμήσεις, οι προτιμησιακές σχέσεις. Άρα δηλαδή νομίζω ότι η κατάσταση είναι σαφής. Βέβαια, το να επαληθέψει κανείς ε, το τι περιέχει ένα προϊόν ως το, προ, περιεχόμενο, αν είναι μέσα κρασί ή όχι, ε, αυτό δεν το εξετάζουν τα τελωνία, γιατί διότι τα τελωνία βασίζονται στις ε, δηλώσεις. Ισχύει καλή πίστη που διέπει τις δηλώσεις και τις ετικέτες. Ως εκ τούτου, κανονικά, δεν ανοίγουν τώρα στα τελωνία τα μπουκάλια για να δουν τι έχει μέσα, αν είναι κάτι παράνομο ή όχι. Αυτό κατά κανόνα δεν συμβαίνει. Η επαλήθευση της δήλωσης, προέλευσης, αυτό κατά κανόνα γίνεται από την ε, εποπτική αρχή του κράτους μέλους και αυτό γίνεται για όλα τα πρόοδα, από όπου και αν έρχονται, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Αυτό δεν το κάνουν τα τελωνία. Τα τελωνία κατά κανόνα αντιδρούν μόνο αν έχουν αποχρώσεις ενδείξεις ότι υπάρχει συστηματική απάτη όσον αφορά στις ετικέτες. Αλλά σας λέω συστηματική όχι δειγματοληπτική, τυχαία, απάτη. Και μάλιστα τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που θα αξιολογήσουν το επίπεδο του κινδύνου και την, ε, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι ανάλογα δηλαδή με τον κίνδυνο. Γιατί ξέρετε τα τελωνία έχουν διάφορες, έχουν ιεράρχηση, ναρκωτικά, όπλα, βασανιστήρια, παράνομες ε, παράνομη διακίνηση, ε, παράνομα προϊόντα. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλέ προτεραιότητε που ισχύουν για τα τελωνία. Και αυτά πρέπει να τα ελέγχουν τα κράτη-μέλη. Εμείς από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είμαστε πάντα πολύ ευαίσθητοι σε θέματα ενδείξεων, αποδείξεων και αυτές τις πληροφορίες θέλουμε να τις διαβιβάζουμε και στα κράτη-μέλη έτσι ώστε και τα ίδια τα κρατη να αξιολογούν με βάση τις δικές τους ε, μεθόδους ε, αξιολόγηση κινδύνου ε, να αξιολογούν πόσο επικίνδυνο είναι να μπουν παράνομα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήθελα να το διευκρινίσω αυτό. Επανέρχομαι τώρα στο θέμα του πώς ελέγχονται όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, εμείς δεν γνωρίζουμε να υπάρχει συστηματική ε, είσοδος προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από κατεχόμενα, τα οποία προϊόντα να εισάγονται με προτιμησιακό καθεστώς. τουλάχιστον τα κράτη-μέλη δεν έχουν ε, λάβει γνώση περί τέτοιου είδους ε, συστηματική εισαγωγή προϊόντων. Τώρα, αν πράγματι υπάρχει συστηματική εισαγωγή, αυτό μπορεί να προκαλέσει πράγματι την αντίδραση ενός κράτους μέλους. Κατά δεύτερον, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε απαραίτητα ότι παραβιάζει τη συμφωνία. Ίσως να υπάρχουν ε, λάθος ε, παράνομες δηλώσεις από μεμονωμένες επιχειρήσεις, αλλά όχι απαραίτητα από το κράτος του Ισραήλ. Απαντώ εδώ στην τρίτη ερώτηση. της κυρίας ε, Αρένα. Οι αρχές του Ισραήλ, να σας πω κάτι, συνεργάζονται. Υπήρχε μια συμφωνία το 2004, εκτότε, εκτότε, με έκτοτε μας ανακοινώνουν τους ε, ταχυδρομικούς κώδικες ε, και τους κώδικες των περιοχών από όπου μπορούν να εισάγονται προϊόντα με προτιμησιακό καθεστώς. Και με το Ισραήλ είμαστε σε συνοχή επαφή, επικαιροποιούνται οι κώδικες, οι τελευταίοι κώδικες δημοσιεύτηκαν τον Ιούνιο του 2015, συνεργαζόμαστε με το Τελαβίβ με την αντιπροσωπεία μας στο Τελαβίβ για να υπάρχει τακτική επικαιροποίηση των κωδίκων. Και πρέπει να σας πω ότι από αυτού του θέματος επικρατεί αγαστή συνεργασία. Ε, εμείς βεβαίως και επιθυμούμε να υπάρχει πιο συστηματική ε, συνεργασία, αλλά ξέρετε δεν μπορούμε να πούμε ότι το Ισραήλ δεν συνεργάζεται. Δεν ισχύει αυτό. Εμείς ε, θα θέλαμε να υπάρχει ένα τέλειο σύστημα, εν πάση περιπτώσει τα πράγματα βαίνουν καλώς προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτά ήθελα να πω, εκτός βέβαια αν οι συνάδελφοί μου θέλουν να πούνε κάτι για το θέμα της ε, σήμανσης για τα στατιστικά δεδομένα τώρα. Πόσα προϊόντα προέρχονται από τα κατεχόμενα. Δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία. Μόνο τα τελωνία των κρατών μελών ενδεχομένως να έχουν κάποια στοιχεία. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης εμείς δεν συγκεντρώνουμε τέτοια στατιστικά στοιχεία. Γιατί μόνο τα κράτη-μέλη έχουν τέτοιου τους πληροφορίες, τα πληροφορικά τους συστήματα, ε, γιατί τα μαζεύουν τα στοιχεία από τις δηλώσεις και από την προέλευση των προϊόντων. Εμείς μάλιστα δεν ξέρουμε καν αν τα κράτη-μέλη έχουν όλες τις λεπτομέρειες για εισαγωγές από περιοχές ε, για τις οποίες ε, εμείς έχουμε ζητήσει τον ταχυδρομικό κώδικα, διότι από εκεί φαίνεται ότι πρόκειται κατεχόμενα αυτή είναι μια έτσι πολύ εντελεχή έρευνα που δεν έχει λάβει η χώρα. Ε, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι τα τελωνία εντάσσονται σε μια ευρύτερη πολιτική αλλά βέβαια η προστασία των πολιτών είναι η πρώτη προτεραιότητα και κατόπιν όλα αυτά ε, θα εξαρτηθούν και από τους πόρους που υπάρχουν, αλλά εμείς δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα τίποτα πιο συγκεκριμένο. Πρόεδρος. Αν δεν κάνω λάθος όμως, ε, τι αίσθηση έχετε από όλο το εγχείρημα που γίνεται. Παρακολούθηση δεν υπάρχει, στατιστικές ε, πληροφορίες δεν υπάρχει, δεν υπάρχει προτεραιότητα στα τελωνία, δεν υπάρχει έλεγχος από τα κράτη-μέλη. Έχει κανένα νόημα τελικά αυτό το εγχείρημα. Εξαρτάται, εξαρτάται. Οι τελωνιακές αρχές εφαρμόζουν σωστά και δεν έχουμε ε, λόγους να πιστεύουμε το αντίθετο γιατί ε, κάποιες ε, έκτακτες περιπτώσεις δεν αποδεικνύουν το κανόνα. Πάντως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση με το σύστημα αξιολόγηση του κινδύνου που έχουμε μπορούμε να σας κοινοποιήσουμε τα πορίσματα, αλλά χρειαζόμαστε ε, πραγματικές αποδείξεις, τεκμήρια και όχι ε, κάποιες ε, τυχές, υπερ, ε, έκτακτες παραβιάσεις. Όταν έχουμε θέματα παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας λόγω των εισαγωγών, τότε γίνεται αναφορά από τα τελωνία. Οπότε, μπορεί να υπάρχουν κάποιες ε, παρεμπίπτουσες ε, αποδείξεις, αλλά γενικώ ε, και κατά κανόνα τα ευρωπαϊκά τελωνία επιτελούν στο έπακρο το έργο τους. Και αν έχουμε ε, τσάντες Λουί που κατασκευάστηκαν κατά παράβαση της πνευματικής ιδιοκτησίας και περνάνε από τα τελωνία μερικέ παρτίδε, αυτό δεν σημαίνει ότι τα τελωνία δεν κάνουν καλά τη δουλειά του, αλλά άμα είναι ε, ε, άπειρες οι περιστάσει, δεν μπορούν να εντοπίζονται κάθε φορά από τα τελωνία. Πάντως δεν μπορούμε να ε, θεωρήσουμε ότι υπάρχει συστηματικό λαθρεμπόριο ή συστηματική παράνομη εισαγωγή τέτοιων προϊόντων. Και δεν έχουμε κανεί, μία υπόνοια, μία αποχρώσα αιτία που να αφιβάλλουμε για την νομιμότητα του Ισραήλ. Κυρία Ρενά, ε, συμφωνώ με τις ερωτήσεις του Πρόεδρου, γιατί και πάλι δεν είναι σαφή τα πράγματα. Εγώ θα προτιμούσα... Βέβαια, είναι δύσκολο να έχουμε στατιστικά στοιχεία για τα προϊόντα που παράγονται στους επικισμούς και που εισέρχονται στο ευρωπαϊκό έδαφος με προτιμησιακούς δασμούς. Είναι δύσκολο, όπως είπατε, γιατί τα τελωνία δεν ελέγχουν κάθε φορά τα προϊόντα, γιατί δεν θεωρούν ότι γίνεται συστηματικά τέτοια παραβίαση, οπότε το ποσοστό κινδύνου δεν είναι σημαντικό. Αυτό θα μπορούσα να το καταλάβω ίσως, αλλά έχετε στατιστικά στοιχεία για προϊόντα που παράγονται στους επικισμούς, εισέρχονται στην Ευρώπη και δεν τυχάνουν της προτιμησιακής διάταξης του προτιμησιακού δασμού. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε ως στοιχεία, γιατί ε, αυτά τα προϊόντα εισάγονται ως με σήμανση προϊόν επικισμού και χωρίς προτιμησιακό δασμό. Αν λέμε ε, προϊόντα αξίας 230 εκατομμυρίων από ε, επικισμούς που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, φαντάζομαι ότι θα είναι χωρίς προτιμησιακούς δασμούς και φαντάζομαι ότι τα στοιχεία σας θα πρέπει να συμπίπτουν με αυτό το ποσό. Έχουμε τουλάχιστον τέτοια στοιχεία. Ε, αυτό θα ήταν ενδιαφέρον. Επίσης, είχαμε διαρροή κάποιων εγγράφων ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λένε ότι και που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανίκανη να επιτελέσει το έργο της. Οπότε υπάρχει μια ασυνέπεια ε, ε, σε σχέση με αυτά που είπατε εσείς που λέτε ότι συνεργάζονται οι αρχές ε, και εργαζόμαστε σωστά, ενώ η έκθεση που διέρευσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ομολογεί την ανικανότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορώ να σας στείλω τα έγγραφα που έχουν διαρρεύσει και που διαπιστώνουν ανικανότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ελέγξει την κατάσταση και υπάρχει αντίφαση μεταξύ αυτών που μας είπατε εσείς ότι όλα πάνε καλά θέλουμε τέτοιε πληροφορίε για να καταλήξουμε σε συμπέρασμα, γιατί σε αντίθεση με αυτά που είπε ο κύριο Φιέλνερ, η συμφωνία σύνδεση, εμπορική σύνδεση με το Ισραήλ δεν είναι μια τυχαία συμφωνία σαν τι είπα Η συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ, όπω και αντίστοιχη με την Παλαιστίνη, έχουν στόχο την ε, ε δημιουργία πρόσφορου εδάφου για την ειρηνευτική διαδικασία ενώ σήμερα θέλουμε αποδείξεις ότι όντως η Συμφωνία Σύνδεσης διευκολύνει την ειρηνευτική διαδικασία και θέλουμε επιχειρήματα που να συνηγορούν υπέρ αυτής της κατεύθυνσης. Οι δεν θα έχουμε τα αντίθετα επιχειρήματα γιατί αν θέλουμε όντως μια ειρηνευτική διαδικασία θα πρέπει να είμαστε να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας ε, για αυτά που υιοθετούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να μην περιμένουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να κρίνει ότι υπάρχει παρανομία. Δεν μπορούμε ε, να περιμένουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να εντοπίσει αυτή την παρανομία. Δεν θέλω να μας φέρετε σε τέτοια θέση να περιμένουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να χαρακτηρίσει μια τέτοια κατάσταση και χρειαζόμαστε στοιχεία για το έργο μας. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Ευχαριστώ πολύ. Όταν λέτε ότι όλα είναι καλά, ο προηγούμενος πρέσβης στο Τελαβίβ είπε αυτή η επισήμανση δεν λειτουργεί. Είπε δεν. Δεν. That's a small comment. Μια σύντομη παρατήρηση. Ευχαριστώ. Στο θέμα των στατιστικών στοιχείων. Θα το ψάξουμε για να δούμε τι μπορούμε να συγκεντρώσουμε. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ, αλλά θα το δούμε. Δεύτερον, τα έγγραφα που διέρευσαν, όπως λέτε. Μιλάμε, νομίζω, για έγγραφα και διορθώστε με γιατί θα το ξέρετε καλύτερα, που είχαν ε, ημερομηνία πριν από 6 μήνες, το Σεπτέμβριο ίσως, ή και πιο πολύ. Εν τω μεταξύ, ε, ε, συνεργαστήκαμε με τις Ισραηλινές αρχές για την ενημέρωση των κωδίκων. Δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλαμε, αλλά προχωρούμε και ελπίζουμε σε καλό αποτέλεσμα και το γεγονός πιστεύω ότι ε, δημιουργούνται ε, αυτές οι ευαισθησίες εντός του Κοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικό γιατί ανεβάζει το επίπεδο προσοχής ε, ώστε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή ανταπόκριση από πλευράς Ισραηλινών αρχών. Τώρα, το θέμα της πιθανής κατάστασης η απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τα κατεχόμενα εδάφη έχουν ε, ομοιότητα με τη Δυτική Σαχάρα για ένα λόγο. Από άποψη Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άποψη διεθνή, πριν από το Δεκέμβριο του 2016 υπήρξε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που έλεγε ότι όλα τα προϊόντα της Δυτικής Σαχάρας έμπαιναν χωρίς δασμούς. Η κατάσταση με το, το Ισραήλ είναι διαφορετική γιατί σε σχέση με τα κατεχόμενα. Γιατί αυτά τα προϊόντα νομικά δεν μπορούν να μπουν με προτιμησιακό καθεστώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δικαστήριο λοιπόν θα μα πει, θα πει σε οποιονδήποτε ισχυριστεί ότι αυτά τα προϊόντα δεν μπορούν να μπουν με προτιμησιακό, θα λέει βεβαίω δεν μπορούν να μπουν με προτιμησιακό καθεστώ δεν μπορούν. Δεν μπορούν να μπουν νόμιμα με προτιμησιακό καθεστώς. Παράνομα όπως και πολλά άλλα έχουμε και τα τσιγάρα, μπαίνουν λαθρέα κλπ. Ναι, ακούστε. Δεν είναι ιδεολογία αυτό λέει ο πρόεδρος. Δεν, τηρεί, δεν τηρούν όλοι τον νόμο βεβαίως, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Δεν μας ικανοποιεί αυτό. Λοιπόν, στο σημείο αυτό κλείσαμε το ζήτημα αυτό. Θα παραμείνει και για τις επόμενες συνεδριάσεις. Τώρα φτάνουμε στο θέμα 24, επίσης ένα θέμα που δεν με διασκεδάζει καθόλου. Το σκέλος ε, το εμπορικό σκέλος της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου. Είχαμε απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 21 Δεκεμβρίου του 2016 σύμφωνα με την οποία η παρούσα κατάσταση και χωρίς την ε, ε, τροποποίηση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου δεν καλύπτει τα προϊόντα που προέρχονται από τη Δυτική Σαχάρα και με βάση αυτή την απόφαση έλαβε εντολή η Κομισιό να διαπραγματευτεί μια τροποποίηση με το Μαρόκο. Πριν από λίγες ημέρες έλαβα μια επιστολή από την Γενική Διεύθυνση Ταξούντ ότι έχει, μόνο ε, έχει φτάσει στην τελική φάση ένα σχέδιο συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκο στις 31 Ιανουαρίου και επιτρέπει την, την κάλυψη αυτών των προϊόντων. Τώρα, η διαδικασία αυτή, στη διαδικασία αυτή δεν συμμετείχε το Κοινοβούλιο, πρέπει να έγινε εν Και διάβασα στην επιστολή ότι το σχέδιο αυτό συμφωνίας θα συνοδεύεται από δύο ε, εκθέσεις αξιολόγησης για τα ωφέλη της συμφωνίας και δεύτερον ε, για την εμπλοκή για τη συμμετοχή του λαού της Δυτικής Σαχάρας. Κατάλαβα ότι οι εκθέσεις αυτές θα βελτιώσουν, δεν έχουν οριστικοποιηθεί, και άρα η απόφαση θα αποφασίσει αν και κατά πόσον θα υποβάλει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο το σχέδιο συμφωνίας. Θέλω λοιπόν φυσικά να μάθω λίγο περισσότερα πράγματα για αυτό το σχέδιο συμφωνίας και τις εκθέσεις. Και ο κύριε Περόντε Πινίκ. Μπορείτε να πείτε σε μένα και στους συναδέλφους λίγο περισσότερα από αυτού. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας ε, ενημερώσω για το πώς έχουν τα πράγματα στη συμφωνία με το Μαρόκο. Από ε, την συνεδρίαση της ομάδας παρακολούθησης της ΣΥΝΤΑ για το Μαρόκο και τη Δυτική Σαχάρα που έγινε στις 24 Ιανουαρίου ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει μια πλήρη επικαιροποίηση της κατάστασης, ιδιαίτερα στα τρία σκέλη που ενδιαφέρουν. Καταρχήν, ε, μια, ένα σχέδιο συμφωνίας που τροποποιεί τη συμφωνία σύνδεσης και προβλέπει ρητά ότι προϊόντα, ε, το σχέδιο λοιπόν ε, συμφωνία σύνδεσης με το Μαρόκο προβλέπει στην τροποποίηση ότι προϊόντα από τη Δυτική Σαχάρα ε, ευνοούνται από, τις από τους προτιμησιακούς δασμούς όπως και τα υπόλοιπα προϊόντα της ε, Συμφωνίας Σύνδεσης. Αυτό είναι το πρώτο σκύλος. Δεύτερον, ε, όπως είπε ο Πρόεδρος, μια έκθεση αξιολόγησης για τα ωφέλη που έχει παρά η επέκταση των προτιμησιακών δασμών και στη Δυτική Σαχάρα, στον πληθυσμό. Και τρίτο θέμα, η διαβούλευση με τον τοπικό πληθυσμό της Δυτικής Σαχάρας ώστε να εξασφαλίσουμε υποστήριξη και του τοπικού πληθυσμού για την επέκταση των προτιμησιακών δασμών και στη Δυτική Σαχάρα. Ε, η ανταλλαγή επιστολών ε, μονογράφη και ολοκληρώθηκε στις 21 Ιανουαρίου και το κείμενο που μονογράφηκε είναι σχεδόν κατά λέξη αυτό που παρουσίασε στην ε, ομάδα παρακολούθησης ε, ο κύριος Ε Το γεγονός ότι μονογράφηκε ένα κείμενο σημαίνει απλώς ότι οριστικοποιήθηκε. Δεν ε, υπάρχει καμία πολιτική δέσμευση μέχρι ότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει πρόταση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για Συνένεση γιατί οι αρμόδιες για την νομοθεσία αρχέ, οι συνομοθέτε δηλαδή αποφασίζουν για το κείμενο. Απλώ το κείμενο οριστικοποιήθηκε, αυτό το νόημα έχει μονογραφή Μπορεί να έχουμε νέε εξελίξεις, γιατί εκρεμεί μια νέα υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αναμένεται η απόφαση 27 Φεβρουαρίου. Μπορεί αυτό να αλλάξει κάπως τα πράγματα, δεν νομίζω, αλλά δεν αποκλείεται κιόλας. Δεύτερο στοιχείο η έκθεση για τα ωφέλη. Ε, εκπονούμε αυτή την έκθεση και ελπίζουμε πολύ σύντομα να είναι έτοιμη. Αυτή η έκθεση αξιολόγησης επισημαίνει σημαντικά ωφέλη για τις εξαγωγές από τη Δυτική Σαχάρα, κυρίως ε, στα γεωργικά προϊόντα καθώς και στα αλληλευτικά προϊόντα. Δεύτερο, η μη επέκταση των προτιμησιακών δασμών και στη Δυτική Σαχάρα θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ε, τωρινές αλλά και στις μελλοντικές εξαγωγές και τις επενδύσεις στη Δυτική Σαχάρα. Και όλα αυτά τεκμηριώνονται και όλα στην έκθεση αξιολόγησης. Ακόμη βέβαια δεν έχει ολοκληρωθεί η επαλήθευση των στοιχείων γιατί τα συγκεντρώνουμε από διάφορες πηγές και ελέγχουμε την εγκυρότητά τους ώστε να είμαστε σίγουροι για το πόρισμα της αξιολόγησης. Και τρίτο στοιχείο, διαβούλευση με τον τοπικό πληθυσμό. Έγινε τέτοια διαβούλευση. Ε, πραγματοποιήθηκε αποστολή με επικεφαλής ε, τον κύριο Βενσάν Πικέ από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που θα σας ενημερώσει για το τι διαμεύθει εκεί. Ε, και είναι σχεδόν, έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν αυτές οι διαβουλεύσεις. Τώρα, τι γίνεται με το χρονοδιάγραμμα και τα επόμενα βήματα. Αναμένουμε την ολοκλήρωση του προπαρασκευαστικού έργου σε επίπεδο υπηρεσιών τις επόμενες 10-15 ε, μέρες και στόχος μας είναι να υποβάλουμε την πρόταση στο Συμβούλιο για ένα σχέδιο απόφαση του Συμβουλίου επί της υπογραφής της ε, συμφωνίας και ε, σχέδιο απόφαση του Συμβουλίου για την ολοκλήρωση της συμφωνίας μετά τη χορήγηση της συνένεσης και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να συντάξουμε αυτές τις προτάσεις κατά τη διάρκεια του Μαρτίου. Και θα σας ενημερώσω ο κύριος Βεσάν Πικί για το τι διεμήθη στο Ραμπάτ την περασμένη εβδομάδα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Γραμματεία του Συμβουλίου έστειλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ε, εντολή της διαπραγμάτευσης και εκεί θα διαβάσατε τι περιμένουν τα κράτη-μέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΕΔ στις διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο. για το θέμα της ανάμειξης του τοπικού πληθυσμού που θα επηρεαστεί από την επέκταση των προτιμησιακών δασμών. Η διαδικασία διαβούλευσης ή ε, ανάμειξης ε, εμπλοκής ε, του, των ενδιαφερομένων ήδη έχει ξεκινήσει και μάλιστα καταρτήσαμε ένα πρόγραμμα συνεδριάσεων που προβλέπει συναντήσεις και στο Ραμπάτ και στις Βρυξέλλες και μάλιστα για το σκοπό αυτό έχουμε επιλέξει ένα κατάλογο, ευρύ κατάλογο και πλούσιο κατάλογο συνομιλητών. Έχουμε μέλη του Κοινοβουλίου, μέλη των Περιφερειακών Δημοτικών Συμβουλίων από τη Δυτική Σαχάρα. Έχουμε οικονομικούς φορείς και παράγοντες, ε, εμπορικά επιμελητήρια, ε, γεωργικούς συνεταιρισμούς και επιμελητήρια, λευτικό επιμελητήριο, κυρίως ε, από το Ντάκλα και το Λαγιούν, από τη Δυτική Σαχάρα, έχουμε ερευνητικά ιδρύματα, οικονομικούς φορείς, αναπτυξιακούς οργανισμούς από τη Δυτική Σαχάρα και μια τρίτη κατηγορία συνομιλητών είναι οργανώσει της κοινωνίας των πολιτών με τη στενή έννοια που επικεντρώνονται κυρίως στα ανθρώπινα δικαιώματα και δει τα ανθρώπινα δικαιώματα των Σαχαραουιτών. Ε, είναι πολύ εκπρόσωποι και αυτών των ΜΚΟ και μάλιστα πρόκειται για ΜΚΟ που είναι καταχωρημένο στο Μαρόκο αυτή ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για μας, δηλαδή να είναι αναγνωρισμένες και εγγεγραμμένες στο Μαρόκο η ΜΚΟ, αλλά και ε, εκεί το φάσμα είναι ευρύ. Έχουμε και πολιτικά ουδέτερες ΜΚΟ, αλλά και πιο στρατευμένες ΜΚΟ που στηρίζουν το μέτωπο Πολυσάριο. Και το μέτωπο Πολυσάριο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των συνομιλητών μας άλλωστε και μάλιστα είχαμε μια συνάντηση ήδη στις αρχές Φεβρουαρίου. Φυσικά δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Βρισκόμαστε περίπου στα μισά του δρόμου. Έχουμε διεκπαιρεώσει το μισό πρόγραμμα μέχρι στιγμής των συναντήσεων και ευελπιστούμε ότι μέχρι τα τέλη του Φεβρουαρίου θα ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας και χάρη στις συναντήσεις αυτές πιστεύω ότι δημιουργούμε μια ε, αξιόπιστη εντύπωση για το πώς βλέπει ο τοπικός πληθυσμός τις τροπολογίες της Συμφωνίας Σύνδεσης και το κατά πόσο θεωρεί ότι θα ευνοηθεί από την Συμφωνία Σύνδεσης είτε από οικονομική είτε από κοινωνική άποψη ή αν έχει οτιδήποτε άλλες αντιρρήσεις ε, για τη σύνδεση ή την υποστηρίζει. Τα πορίσματα των συναντήσεών μας ε, θα συμπεριληφθούν στην έκθεση αξιολόγηση που θα στείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με την επίσημη πρόταση για τροποποίηση της Συμφωνίας Σύνδεσης με το Μαρόκο. Δεν θα επισέλθω ακόμη στο περιεχόμενο, γιατί παραλαμβάνω δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι οι Μαροκινές αρχές θα πραγματοποιήσουν και αυτές διαβουλεύσεις. Η κυβέρνηση μάλιστα θα θέσει και σε ψηφοφορία την τροποποίηση της Συμφωνίας Σύνδεσης και σε δύο επίπεδα. Πρώτα στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων σε εθνικό επίπεδο και εν συνεχεία θα ζητήσουν και από τα περιφερειακά συμβούλια της Δυτικής Σαχάρας να ψηφίσουν. Πρόκειται για περιφερειακά συμβούλια που εθετούν ε, μια πιο περιφερειακή τοπική σκοπιά και εξυπηρετούν περίπου τα τοπικά και περισσότερο τα τοπικά και περιφερειακά συμφέροντα. Μετά την έκβαση και των ε, ψηφοφοριών αυτών, ε, η μαροκινή κυβέρνηση θα καταλήξει στην στη στάση των Σαχαροϊωτών και σε επίπεδο Εθνικού Κοινοβουλίου και σε επίπεδο Περιφερειακών Συμβουλίων. Έτσι θα αποκομίσει μια εντύπωση για τη γνώμη των Σαχαροϊτών και θα διαπιστώσει κατά πόσο υπάρχει υποστήριξη εκ μέρους Σαχαροϊτών ε, υπέρ της τροποποίησης της Συμφωνίας Σύνδεσης. Ευχαριστώ. Και εμείς, λέει ο Πρόεδρος, ε, για να είμαι ειλικρινής δεν ικανοποιήθηκα γιατί έχω την εντύπωση ότι η Γενική Διεύθυνση Τάξου έχει διαφορετική άποψη από το Κοινοβούλιο. Η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, Trade, είναι πολύ συνεργάσιμη. Ε, τα πάμε καλά. αλλά εσείς ε, είναι άλλη στάση σας. Ε, τα επεξεργάζετε το γραφείο σας, μετά έρχεστε εδώ και λέτε αυτό είναι, πάρτε το. Η τροπολογία έγινε, η τροποποίηση μάλλον έγινε τον Μάιο και τη φέρετε εδώ στο Κοινοβούλιο λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Δεν είναι σωστό αυτό, απαράδεικτο. Παρόλα αυτά, ε, δεν είναι δική μου δουλειά να σχολιάζω αυτή τη στιγμή. Τώρα ένα πρόβλημα. Εννέα μέλη θέλουν να λάβουν το λόγο και έχουμε 20 λεπτά μόνο στη διάθεσή μας που σημαίνει 1,5 λεπτό καθένας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την εισηγητριά μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έστειλαν εκπροσώπους για να μας ενημερώσουν λεπτομερέστερα για τις ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις με τον Ερετέρο, το Μαρόκο, παρά τη Συμφωνία Σύνδεσης που μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου που βρίσκεται σε φάση οριστικοποίησης. Ως μόνιμη ε, εισηγήτρια για τις σχέσεις με τις χώρες Μαγκρέμπ για την Κοινοβουλευτική Επιτροπή θέλω να επισημάνω τα σημαντικά σημεία στο πλαίσιο της διαπραγματεύση, επί των οποίων πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι προσεκτικό. Όπω γνωρίζετε και επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν ήδη. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου στις 21 Δεκεμβρίου του 2016, το Συμβούλιο ανέθεσε στην Κομισιό να διαπραγματευτεί συμφωνία με το Μαρόκο που τροποποιεί το, ε, ε, το εδαφικό πλαίσιο των προτιμήσεων έτσι ώστε τα προϊόντα της Δυτικής Σαχάρας να έχουν τις ίδιες συνθήκες όπως και τα προϊόντα του Μαρόκου. Ε, εκεί αναφέρεται ρητά εξ όσων γνωρίζουμε η Δυτική Σαχάρα έτσι ώστε τα προϊόντα που εξάγονται από αυτή την περιοχή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξακολουθούν να χαίρουν των ίδιων προτιμησιακών συνθήκων υπό ορισμένε προϋποθέσεις που έχει θέσει το δικαστήριο. Δύο σημαντικά ε, στοιχεία ε, ε, εμπλέκονται εδώ. Πρώτον, και αυτό είναι σημαντικό, να μην παρεμβεί με τη διαδικασία που είναι εν εξελίξει στα Ηνωμένα Έθνη για την ειρήνευση. Αυτό ε, είναι προπόθεση και για τι δύο πλευρές. Δεύτερον, να μην τεθεί υπό αμφισβήτηση η θέση της Ένωση όσον αφορά την κυριαρχία της ε, περιοχής δυτική Σαχάρας. Διότι αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο τη διαπραγματεύση. Τα στοιχεία αυτά είναι αυτά και κατόπιν θέλω να αναφερθώ σε τρία θέματα επί των οποίων πρέπει να είναι σε τη φυλακή το κοινοβούλιο μας και να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες στη συμφωνία. Πρώτον, η, αναφορά της Δυτικής Σαχάρας στο, εδαφικό πλαίσιο της συμφωνίας. Δεύτερον, η τροποποίηση της συμφωνίας πρέπει να γίνει προς όφελος των τοπικών πληθυσμών, τα, προς οικονομικό όφελος και τρίτον, ο λαός και λέω ο λαός που ε, τον αφορά να συνενέσει. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης εμπλέκεται λόγω της πολιτικής και διπλωματικής διάστασης ε, της ε, διαδικασίας των διαβουλεύσεων. Βεβαίως είναι ευθύνη μας να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα των οργανισμών με τους οποίους γίνεται η διαπραγμάτευση και ότι θα είναι ξεκάθαρη η συνένεση του λαού που τον αφορά. Φυσικά αυτό είναι η λέξη κλειδί. Ολοκλήρωσα σχεδόν. Θα ήθελα να ανοίξω μια παρένθεση σημαντική για να πω ότι ο πρώην Γερμανός πρόεδρος, ο κύριος Ασκόλερ, ε, έστειλε ειδικό ε, διαπραγματευτή των ε, Ηνωμένων Εθνών στη Δυτική Σαχάρα και ότι η διαδικασία η ίνευση Σαχάρας Δυτικού Μαρόκου έχει επανέλθει και αυτό είναι πολύ καλό. Πρέπει να κλείσω, αλλά είχα να πω κι άλλα, αλλά τι να κάνουμε. Αυτά. Ευχαριστώ. Ήμουν λίγο γενναιόδωρος γιατί εσείς είστε η εισηγήτρια, αλλά πραγματικά θα είμαι αυστηρός τώρα, 1,5 λεπτό ο καθένας. Ευχαριστώ πολύ για τη γενναιοδορία σας, λέει η ομιλήτρια. Είχα κι άλλα να πω, θα τα πω μετά. Ο κύριος Μπούχνε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τι ακριβώς αποφάσισε, είπε ότι η ε, κάτοικοι της Δυτικής Σαχάρας πρέπει να δεχθούν όλες τις συμβάσεις. Και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή μιλάει με την κυβέρνηση, ε, καταλήγει σε μια τεχνική συμφωνία και εκ των υστέρων ε, απευθύνεται στους ε, κατοίκους που ζουν στη Δυτική Σαχάρα, αλλά αυτοί είναι κυρίως οι κατακτητές. Οι ε, πραγματικοί Σαχαροίτες ε, είναι πολύ λίγοι. Οι άλλοι που ζουν εκτός της Δυτικής Σαχάρας δεν μπορούν καν να ε, απαντήσουν. Άρα δηλαδή τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλεί τους περισσότερους ντόπιου κατοίκους και αυτό σημαίνει για μένα ότι η απόφαση του δικαστηρίου ποδοπατείται πολλοί λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας θεσμός ε, ο οποίος ε, υπηρετεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά τι συμβαίνει τώρα. Εδώ βλέπουμε ότι πρόκειται για όνειδος γιατί προστατεύουμε μόνο τους ε, κατακτητές οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να εκμεταλλεύονται και να κερδίζουν χρήματα από αυτήν την κατάσταση. Ευχαριστώ. Μία υπενθύμηση γιατί βρισκόμαστε εδώ σήμερα, γιατί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, έβγαλε απόφαση που λέει ότι η συμφωνία για τα γεωργικά προϊόντα δεν ε, τηρείται, δεν γίνεται σεβαστή, γιατί υπάρχουν προϊόντα της Δυτικής Σαχάρας που μπαίνουν στο ευρωπαϊκό έδαφος, ενώ η συμφωνία δεν το προβλέπει. Οπότε πρέπει να την αναθεωρήσουμε. Και το δικαστήριο λέει, έχετε δύο δυνατότητες. Είτε θα συνεχίσετε να θεωρείτε ότι ε, η Δυτική Σαχάρα είναι εκτός συμφωνίας αλλά δεν επιτρέπεται εισαγωγή προϊόντων, είτε θα τη συμπεριλάβετε αλλά χρειάζεται η συνένεση του τοπικού πληθυσμού. Δεν θα λύσουμε εμείς στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου το πρόβλημα της Δυτικής Σαχάρας, αλλά θα ήταν σκόπιμο και καλό η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα διαπραγματευτεί με την μαροκινή κυβέρνηση να συνάδει με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό που θα πρότεινα λοιπόν είναι Εμεί στην Επιτροπή ΙΝΤΑ να θέσουμε ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το κατά πόσο είναι ε, νομότυπη η διαδικασία διαπραγμάτευσης με την νομολογία. Αν το δικαστήριο την κρίνει νομότυπη, τότε μπορούμε να ψηφίσουμε την συμφωνία που διαπραγματευτήκατε. Αν όμως το δικαστήριο μας πει ότι το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης δεν ανταποκρίνεται ή δεν τηρεί την νομολογία του, τότε θα ήταν κάπως περίεργο να ζητάτε από ευρωβουλευτές να υπερψηφίζουν κάτι που είναι παράτυπο. Ε, θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, ζητήσει, να θέσει την ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αφού δεν το κάνει, θα πρέπει να το κάνουμε εμείς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα σας πω την αλήθεια. Ε, μένω άναυδος με τις προτάσεις που μας κάνατε. Έχω πάθει σοκ. Ε, μας είπατε για πολλά πράγματα, αλλά δεν μιλάμε εμείς για διαβούλευση. Εδώ ε, αναμένεται η συνένεση του λαού της Σαχάρας. Και αυτά που μας είπατε δεν α, μας επιτρέπουν να διαβλέψουμε καμία συνένεση. Ουσιαστικά ε, κάνει κάποια διαβήματα η μαροκινή κυβέρνηση για να, και φροντίζει για τη συνένεση του Σαχαρο, των Σαχαροϊτών. Δηλαδή τι θα κάνουμε, ε, στους επίκους του Ισραήλ θα ζητήσουμε να, να εκμεύσουν την συνένεση από τους Παλαιστινίους. Όχι. Η Δυτική Σαχάρα είναι ξεχωριστό έδαφος, δεν εμπίπτει στην επικράτεια του Μαρόκου. Δεν θα πρέπει λοιπόν το Μαρόκο να ζητήσει τη συνένεση από τους Σαχαραουίτες. Επίσης το έχουμε πει ε, ότι, και το έχουν πει και οι οργανώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολλές ΜΚΟ της Δυτικής Σαχάρα δεν επιτρέπεται να ταξιδέψουν στο Ραμπάτ, γιατί ε, το Μαρόκο δεν τι αναγνωρίζει. Πώς είναι λοιπόν... Ε, πώς είναι δυνατόν να αγνοείτε αυτά τα στοιχεία. Επίσης, πώς θα μεριμνήσετε, πώς θα συνάψετε μια τέτοια συμφωνία χωρίς στοιχεία. Από ό,τι ξέρουμε έχουμε 7.000 ε, ευρώ εισαγωγές από τη Δυτική Σαχάρα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι θα σας πιστέψει κανείς 7.000 ε, ευρώ ε, ύψος των εμπορικών συναλλαγών με τη Δυτική Σαχάρα. Είναι δυνατόν να περιμένετε από εμάς το πιστέψουμε. Συμφωνώ με τη Μαρία Ρενά να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κύριε Πρόεδρε, ακριβώς όπως και άλλοι και εγώ πραγματικά ε, τα έχω χάσει με την κατάσταση που έχει προκαλέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και νομίζω ότι η απόφαση είναι απόλυτα σαφής. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να υπάρξει καμία σύμβαση με το Μαρόκο και τη Δυτική Σαχάρα αν δεν υπάρχει κατηγορηματική ε, συνένεση των κατοίκων της Δυτικής ε, Σαχάρας. Η Κομισιόν τα κάνει όλα περίπλοκα. Η Δυτική Σαχάρα είναι μια χώρα υπό υποκατοχή. Εδώ, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ισχύει το διεθνέ δίκαιο και το Μαρόκο ε, δεν μπορεί να υποφελείται από προϊόντα από τα κατεχόμενα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά ε, φέρνει την Επιτροπή σε πολύ δύσκολη θέση. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να εφαρμόσετε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου και να ζητήσετε την ε, αδιαπραγμάτευτη συγκατάθεση των κατοίκων της Δυτικής Σαχάρα. Σαχάρας. Κύριε Πρόεδρε, ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι υπάρχει αυτή η απόφαση του δικαστηρίου του 16 που αναφέρει με απόλυτη σαφήνεια ότι η Δυτική Σαχάρα δεν είναι τμήμα του Μαρόκου και τα εδάφη της Δυτικής Σαχάρας δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε καμία συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαρόκου χωρίς την ε, αδιαμφισβήτητη συγκατάθεση και συνένεση ε, των κατοίκων. Η Επιτροπή πρέπει να μας πει Πώς θα αποκτήσει αυτή την ε, συγκατάθεση. Η άποψη των Πολυσάριων και της κοινωνίας είναι πολύ σημαντική. Ε, Επίση, εξ όσων κατάλαβα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δεν έκανε μελέτη αντικτύπου πριν από τις διαπραγματεύσεις, γιατί ε, το, τα εδάφη εκεί είναι υπό το φακό των παρατηρητών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Είμαι και εγώ κατάπληκτη όπως και όλοι οι άλλοι. Πώς ε, διαχειρίζεστε αυτό το θέμα. Περίμενα τουλάχιστον να προσπαθήσετε να μας κάνετε να πιστέψουμε ότι ε, ευθυγραμμίζεστε με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά μας λέτε το ακριβώς αντίθετο, ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είπε το δικαστήριο. Και αυτό αφορά κατεχόμενα εδάφη. Δεν είναι το ίδιο με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, λέτε. Μα περί αυτού ακριβώς πρόκειται για κατεχόμενα εδάφη. Και θέλετε να συμφωνήσουμε ότι το Μαρόκο θα πουλάει προϊόντα από αυτά τα κατεχόμενα. Ισχυρίζεστε ότι έχετε συμπεριλάβει τον πληθυσμό. Λέτε ότι θα αποφεληθεί ο κόσμος, ο λαός, αλλά δεν λέει το, αυτό το πράγμα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει ότι πρέπει να ρωτήσετε το ε, ε, νόμιμο εκπρόσωπο του λαού της Δυτικής ε, ε, και συμφωνώ με αυτούς. Μπορούμε να διαπραγματευόμαστε όπως θέλουμε με το Μαρόκο ή με τη Δυτική Σαχάρα, αλλά μιλάμε για δύο διαφορετικές κυβερνήσεις, δύο διαφορετικές περιοχές. Και το θέμα είναι από πού προέρχονται τα προϊόντα. Για την Παλαιστίνη είπατε ότι θα γράψετε θα δηλώνετε ότι τα προϊόντα προέρχονται από κατεχόμενα εδάφη. Θα το κάνετε και εδώ αυτό. Θα εξασφαλίσετε ότι στα προϊόντα αναφέρετε ότι προέρχονται από κατεχόμενα εδάφη. Αυτό σημαίνει ότι αποδέχεστε ότι πρόκειται για, ε, για κατεχόμενα. Κυρία Σάντσουτς. Ευχαριστώ. Η νομολογία του ΔΕΚ ε, προβλέπει ρητά ότι οι συμφωνίες με το Μαρόκο δεν εφαρμόζονται στη Δυτική Σαχάρα χωρίς τη συνένεση του τοπικού πληθυσμού. Και μάλιστα η απόφαση πιστεύει ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού του λαού είναι το μέτωπο Πολυσάριο. Και το Πολυσάριο δεν είναι ένας ακόμη από τους ε, συνομιλητές σας. Μακρύς κατάλογος και ένας από αυτούς καλεσμένους στις ε, διαβουλεύσεις είναι και το μέτωπο Πολυσάριο. Όχι, έτσι προσπαθείτε απλώ να σώσετε τα προσχήματα και με τη διαπραγμάτευση νέων συμφωνιών. Και το νέο σχέδιο διαβούλευση έχει πολλέ ελλείψει, πολύ σοβαρέ. Για παράδειγμα, δεν έγιναν ε, στο, στα εδάφια, αλλά στη, στα γραφεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σχολείο και συνάδελφοι. Ξεχάσαμε και τα τα σχόλια του Γενικού Εισαγγελέα για την Ελευτική Συμφωνία. Και εκεί αναφέρεται ότι η Δυτική Σαχάρα θεωρείται κατεχόμενο έδαφο και θα πρέπει να τηρηθεί το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο. Όπως είπαμε προηγουμένως και για το Ισραήλ, η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Δυτική Σαχάρα επουδενή δεν θα πρέπει να ωφελεί το κράτος που έχει εισβάλλει στα κατεχόμενα, που είναι το Μαρόκο. Θα πρέπει λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρήσει την νομολογία του ΕΛΚ πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Συμφωνώ με τη Μαρία Ρενά ότι δεν μπορείτε να ζητάτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ψηφίσει κάτι το παράνομο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Είναι Σαγιάλα Σέντερ. Ε, είστε πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες Μαγκρέπ. Θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν, ζήτησε, δεν είχα ζητήσει το λόγο γιατί δεν είμαι μέλος της Επιτροπής, αλλά σας ευχαριστώ παρόλα αυτά που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Και να πω πως πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διορθώσει την πορεία της. Δεν, θα είναι το 10 αυτό που θα αποφασίζει ε, στη θέση των Ηνωμένων Εθνών και με ενοχλεί η τροπή που πήραν οι διαβουλεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να έχει ένα ευρύ φάσμα συνομιλητών δεδομένων των περιστάσεων, αλλά διαρωτώ με αν θα πρέπει να γίνει αυτή η διαβούλευση. Γιατί το πρόβλημα της διαβούλευσης είναι κάτι που πρέπει να δεξαχθεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υπεύθυνη για να οργανώσει τη διαβούλευση και να πάρει την απόφαση για τους Σαχαροίτες ή να κρίνουμε εμείς ποιοι είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι των Σαχαροϊτών. Αυτή είναι η βασική μου ανησυχία, γιατί από την άλλη πλευρά έχουμε τη μαροκινή κυβέρνηση και το μαροκινό λαό που επίσης έχουν πολλά προβλήματα, ήδη έχουν αρκετά και αυτοί στο κεφάλι τους. Και εγώ ως ε, πρόεδρος αντιπροσωπείας για τις σχέσεις ε, με τις χώρες Μαγκρέπ δεν μπορώ να εκφράσω την ανησυχία μου για τη μεγάλη αστάθεια που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Μαρόκο. Ήταν δηλητηριασμένο το δώρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ΔΕΚ προσπάθησε με την απόφασή του να ε, ρυθμίσει μια κατάσταση που κανονικά τα Ηνωμένα Έθνη είναι αρμόδια να επιλύσουν. Και εκεί θα πρέπει να αφήσουμε σε αυτό το φόρουμ, όχι στα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στα Ηνωμένα Έθνη την ευθύνη να λάβει την απόφαση. Εντάξει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πέντε λεπτά για να σχολιάσει. Πέντε λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την γενεδορία σας. Το εκτιμάμε πολύ. Τώρα, το θέμα ε, πλήρως αντιλαμβανόμαστε την απογοήτευσή σας ε, Πρόεδρε ότι τα έγγραφα δεν σας έχουν σταλεί για το φάκελο αυτό, όπως έχει συμβεί ε, σε άλλες περιπτώσεις ε, εμπορικών διαπραγματεύσεων. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα όσον αφορά την επικεφαλής γενική διεύθυνση. Είμαστε κομισιόν, αλλά λόγω της ευαισθησίας του φακέλου και των πολιτικών επιπτώσεων. Αυτός είναι ο μόνος λόγος εντός της κομισιόν εμείς ε, συντονίζουμε όλες τις θέσεις. Δεύτερον, σεβόμαστε το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Προβλέπεται στις οδηγίες διαπραγμάτευσης που έχει λάβει η Κομισιόν από το Συμβούλιο. Αναφέρεται ότι πρέπει να αξιολογηθεί η επίπτωση, τα ωφέλη για το, για το λαό και ότι να εξασφαλιστεί ότι όσους αφορά η συμφωνία έχουν γνωμοδοτήσει αυτό. Και βεβαίως θα τηρήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις, όπως επίσης και όσα προβλέπει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Υπάρχει όμως ένα μικρό πρόβλημα. Πώς θα μετρήσουμε ή θα αποκτήσουμε τη συνένεση χωρίς πρόσβαση σε κάθε και ποιος θα καθορίσουμε ποιος είναι από τη Δυτική Σαχάρα. Γι' αυτό χρειάζεται μία διαβούλευση με, τον τρόπο, με τρόπο που να φτάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον πληθυσμό της Δυτικής Σαχάρας. Αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική. Όσον αφορά το ερώτημα το αν μπορούμε να ελέγξουμε και αν πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προϊόντα από τη Δυτική Σαχάρα όπως και αυτά από τα, κατεχόμενα δεν είναι το ίδιο. Γιατί στην περίπτωση τα προϊόντα της Δυτικής Σαχάρας δεν θα είχαν προτιμησιακό καθεστώς και θα έπρεπε να εισαχθούν με πλήρης δασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ τα προϊόντα από τα κατεχόμενα δεν μπορούν. Και επίσης θα ήθελα να πω και θα το πει ο συνάδελφος ε, μάλλον αν, έχετε, αν δεν έχετε αντίρρηση. Θα είμαι πολύ σύντομος. Απλώς να πω ότι σημειώνουμε πολύ προσεκτικά τις ε, παρατηρήσεις σας και θα τις αντιμετωπίσουμε με μεγάλη σοβαρότητα. Ειλικρινά θα σας πω ότι δεχόμαστε ότι το θέμα της συνένεσης είναι ο καθοριστικός παράγων για, την, για το επίπεδο πεποίθησης που μπορούμε ε, να μεταφέρουμε στο Κοινοβούλιο πόσο πιστικοί θα είμαστε για την πρότασή μας. Αντιμετωπίζουμε απολύτως ε, σοβαρά το θέμα αυτό. Δεν είναι πράγματα αυτά που γίνονται γρήγορα, που διεκπεραιώνονται απλώς. Βεβαίως δεν πάμε στο πεδίο να συναντηθούμε με τους απευθείας με αυτούς που άμεσα ή έμεσα επηρεάζονται από τη συμφωνία. Μιλάμε στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Μιλάμε σε επίπεδο πολιτικό, μιλάμε στο Πολυσάριο και έχω επαναλάβει το σχόλιο αυτό και στο παρελθόν και εδώ και αλλού, ναι, ότι ναι, το Πολυσάριο παίζει ρόλο ε, εδώ, αλλά το Πολυσάριο δεν είναι ο μοναδικός συνομιλητής μας. Δεν είναι δυνατόν αυτό γιατί δεν έχει γνωρίσει το Πολυσάριο ως τέτοιο κανένα κράτος μέλος. Κανένα κράτος μέλος δεν έχει αναγνωρίσει το SARD την, λαϊκή δημοκρατία της Σαχάρας, άρα ούτε εμείς μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε, συνομιλούμε μαζί τους γιατί έχουν φωνή φυσικά. Όμως μπορώ επίσης να σας πω ότι οι Σαχαράουοι οι οποίοι ζουν στη Δυτική Σαχάρα δεν αναγνωρίζουν ούτε αυτή το πολυσάριο. Οπότε ε, αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρήσαμε στις συζητήσεις μας η, η αντιπροσωπευτικότητα του πολισαριο και αυτή καθεαυτή δεν είναι πλήρης. Θα είμαι σύντομος, δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά είναι κάτι που προσπαθούμε να το προχωρήσουμε με μεγάλη προσοχή και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να συμμορφωθούμε όχι μόνο με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά και με την διαδικασία του ΟΗΕ, την διεθνή νομοθεσία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κλπ. Και γνωρίζω ότι είναι μια δοκιμασία, πιστεύω όμως ότι θα την περάσουμε, ότι θα τα καταφέρουμε να συνδυάσουμε όλα τα στοιχεία και να σας πείσουμε για αυτό το οποίο λέμε. Πρόεδρος, ε, έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι πρέπει να παραμείνουμε σε επαφή για αυτό το θέμα. Και τώρα, τελευταίο θέμα για σήμερα είναι η παρουσία της μελέτης με θέμα η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόσβαση στην αγορά επιτυγχάνει τους κύριους στόχους της. Έχουμε 25 λεπτά και θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Χέκμαν να μας παρουσιάσει τη μελέτη αυτή για να μπορούμε μετά να υποβάλουμε και κάποιες ερωτήσεις. Όποιος θέλει να φύγει, παρακαλώ να αποχωρήσει ησύχως. Quietly. Okay, Mr. <clears throat> Λοιπόν, ο στόχος αυτής της έκθεσης είναι να αξιολογήσουμε την στατική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόσβαση στην αγορά για να δούμε ε, πώς ακριβώς ε, βρίσκεται σε επαφή με τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Η μελέτη αποτελείται από τέσσερα τμήματα. Το ένα μας παρουσιάζει την στρατηγική μετά τις συνεργασίες. Υπάρχει ένα τμήμα για την ε, στρατηγική και τις αντιλήψεις που υπάρχουν. Αυτά απορρέουν από τις απόψεις των άμεσα ενδιαφερόμενων. Από συνδεύξεις που έχουμε κάνει, το τρίτο τμήμα της μελέτης εστιάζει στις προκλήσεις που αφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Επιτροπή, στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε εξαγωγικές αγορές για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να εντοπίσουμε ποιες είναι οι διαδικασίες που οδηγούν σε αυτό το συγκεκριμένο μηχανισμό και στο τέλος της μελέτης καταλήγουμε σε πορίσματα και συστάσεις και σε ε, κάποιες προτάσεις για το τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να είναι πιο επιτυχημένη αυτή η στρατηγική. Είμαι σίγουρος ότι όλοι σας γνωρίζετε αυτό το συγκεκριμένο εργαλείο το οποίο έχει εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να διευκολύνονται οι εξαγωγές των ε, ευρωπαϊκών κρατών σε αγορές τρίτων χωρών να έχει κανείς πάντα κατά νου τις εξαγωγές. Ε, αυτό που χρειαζόμαστε είναι να συγκεντρώσουμε πληροφορίες, ε, να γίνεται αξιολόγηση, να δούμε λιγάκι τι μπορούμε να κάνουμε, το πόσο σημαντικό είναι να υπάρξει ιεράρχηση της δουλειάς μας και κατόπιν ε, συγκεκριμένα μέτρα για να εντοπίσουμε τους φραγμούς. Οι μηχανισμοί που έχουν σχέση με αυτή τη στρατηγική είναι ε, ουσιαστική και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον ιδιωτικό φορέα, από εταιρείε, από ε, ε, ενώσεις εταιριών. Κυρίως αυτό που ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσον αυτοί όλοι οι φραγμοί έχουν κάποια οικονομική σημασία, ε, κατά πόσον σέβονται τους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ε, πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ε, σχετικά με αυτούς τους φραγμούς, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι ε, να υπάρχει συνεργασία με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και των κρατών μελών. Υπάρχει εδώ μια σημαντική, ένα σημαντικό στοιχείο λογοδοσίας. Η λογοδοσία αφορά κυρίως ε, την Τράπεζα εντομένων για την πρόσβαση στις αγορές. Αυτά τα μέτρα τα οποία έχει συμφωνηθεί ότι κατ' ουσίαν αποτελούν φραγμούς ε, στο εμπόριο και ότι έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά όλα αναφέρονται στην Τράπεζα και πρόκειται να συνταχθεί μια έκθεση για το τι ακριβώς ε, έχει επιτευχθεί, πώς μπορούν να αρθούν συγκεκριμένοι φραγμοί και όλα αυτά έχουν συμπληρωθεί από μια διαδικασία έτσι ώστε ε, να ε, επεξεργαστούμε τις ιστορίες, τις επιτυχημένες περιπτώσεις, να δούμε πώς έχουν αποφεληθεί συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Ξέρετε ότι υπάρχει μια διαδικασία να υπάρχει καλύτερη στρατηγική πρόσβαση στην αγορά, ε, να εφαρμόζεται, να συνδέεται αυτή περισσότερο με τις εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα ερώτημα που ετέθη είναι το τι ακριβώς μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να έχετε έτσι μια ιδέα για το τι ακριβώς μιλάμε, για το ποια είναι τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτή την τράπεζα δεδομένων και στην ε, ε, ιεράρχηση. Ε, πάρα πολλά μέτρα προφανώς ε, και έχουν ε, να κάνουν κατά κάποιον τρόπο με τον περιορισμό των εισαγωγών που πολλά από αυτά τα, πολλοί από αυτούς τους φραγμούς δεν είναι δασμοί, πολλοί έχουν με την τυποποίηση προϊόντων, τεχνική φραγμή, οι φραγμοί που τίθενται από τον ΠΟ είναι πολλά μέτρα ε, φραγμοί που υπάρχουν στην τράπεζα δεδομένων. Η στρατηγική είναι μια στρατηγική που ξεκινάει εκ των άνω προς τα κάτω. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν είναι απαραίτητα η άποψη Επιτροπής για το τι είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια συγκεκριμένη αγορά. Κατ' ουσίαν υπάρχει αντίδραση σε συγκεκριμένες διαμαρτυρίες από εταιρείε, από ενώσεις επιχειρήσεων ε, όταν για την παρέμβαση επιτροπής είναι η επιτροπή παρεμβαίνει για να δει πώς μπορεί να ιεραρχήσει ένα συγκεκριμένο μέτρο και υπάρχει μια ολόκληρη σειρά ε, μέτρων και παρεμβάσεων που μπορούν να λάβουν χώρα έτσι ε, ας πούμε μπορεί κανείς ε, να απευθυνθεί στον ΠΟΕ αν θεωρείται ότι ένα συγκεκριμένο μέτρο παραβιάζει μια υποχρέωση του ΠΟΕ. Από το 2008 ε, έχουν αρθεί περίπου 280 εμπόδια λόγω αυτής της διαδικασίας και ε, οι περισσότερες διαδικασίες εμφανίζονται στις ε, αναπτυσσόμενες οικονομίες αλλά και στις γειτονικές χώρες. Κατά μέσο όρο ένα τρίτο των μέσων που έχει ε, αρθεί, έχει σχέση με τη στρατηγική και τα υπόλοιπα με τα προϊόντα. Κάτι που πρέπει να έχουμε κατανοηθεί, αν, έχουμε, ε, αν δούμε τα μέτρα και την τράπεζα δεδομένων, το 20% κάποια στιγμή καταργήθηκαν, αφαιρέθηκαν. πολύ βέβαια φραγμοί εξακολουθούν να υπάρχουν. Είναι δύσκολο να τους απομακρύνει κανείς όλους. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ε, θα πρέπει να αρθούν περισσότεροι φραγμοί και αυτό είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε. Κάναμε μια έρευνα στους ενδιαφερόμενους με επίκεντρο της Ενώσης της Βιομηχανίας που ενδιαφέρονται κυρίω για, για το μηχανισμό αυτό αλλά και συνομιλήσαμε με επιχειρήσεις μικρομεσαίες, μεγάλες στέλνοντας ένα ερωτηματολόγιο Καταρχήν, η πρώτη ερώτηση ήταν ε, γνωρίζετε αυτό το μηχανισμό και από τις ε, απαντήσεις που λάβαμε, όσους, και ακόμη και από όσους γνώριζαν το μηχανισμό, δεν γνώριζαν, δεν ήταν σίγουροι πόσο, πώς και πόσο ε, αποτελεσματικός μπορεί να είναι. 181 απαντήσεις λάβαμε, κυρίως από το ιδιωτικό τομέα, στην έρευνά μας, από ε, βιομηχανικές ενώσεις και ούτω καθεξής. Το αποτέλεσμα της έρευνας ε, δείχνει ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις έμειναν ικανοποιημένες από τη διαδικασία αυτή και από το πώς ε, λειτουργεί, αλλά κατέστησα σαφές από την έρευνα ότι πολλές επιχειρήσεις δεν είχαν ιδέα για το μηχανισμό αυτό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να ξεπεράσουν τους φραγμούς ε, των άλλων δαπών αγορών. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας. Όσοι συμμετέχουν ενεργά πάντως και γνωρίζουν το μηχανισμό και τον ε, εφαρμόζουν, είναι υπέρμαχοί του. Στο έγγραφο έχω περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα επειδή πιέζει ο χρόνος ε, δεν πρόκειται να σταθώ σε όλα τα θέματα διεξοδικά. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι δεν γνωρίζουν όλες οι επιχειρήσεις το μηχανισμό. Πολλές τον αγνοούν. Αυτό όμως δεν είναι επίκριση για το μηχανισμό. Ο μηχανισμός ε, στοχεύει κυρίως προς τις ε, ενώσεις τις βιομηχανικές ε, που προωθούν αυτά τα θέματα και που συζητούν τα ζητήματα των φραγμών, αλλά ας λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν την ύπαρξη αυτού του μηχανισμού. Ε, Μα ρώτησαν και πώ λειτουργεί ο μηχανισμό. Ήταν και τμήμα τη εντολή. Ποια ήταν καταρχήν τα βασικά επιτεύγματα, ήταν και ερώτηση τη έρευνα τη στρατηγικής για την πρόσβαση στις αγορές. Όλοι συμφωνούν ότι η στρατηγική πρόσβαση στις αγορές ήταν αποτελεσματικό μέσο που ενίσχυε την διαφάνεια. Γιατί ε, αυτό είδαμε και από τις συνεντεύξεις, γιατί εκτός από την έρευνα κάναμε και συνεντεύξεις με κυβερνητικούς εκπροσώπους, με εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα και η έρευνα και τα αποτελέσματα της έρευνας ευθυγραμμίζεται με το feedback και τις πληροφορίες που λάβαμε από τις ε, ε, συνεντεύξεις που διοργανώσαμε. Όλοι συμφωνούν λοιπόν ότι η στρατηγική πρόσβαση στην αγορά κέρδισε σε αποτελεσματικότητα ε, από όσο εφαρμόζεται και μείωσε τους φραγμούς ε, στην πρόσβαση άλλων αγορών. Επίσης, ποιο είναι το ποσοστό επιστροφής για τη μέση επιχείρηση την ένωση που χρησιμοποιεί αυτό το μηχανισμό, γιατί είναι πολύ χρονοβόρη διαδικασία, απαιτεί πολλές προσπάθειες, ε, πολλούς πόρους και η επιστροφή δεν είναι αρκετά ικανοποιητική, τότε δεν θα χρησιμοποιήσουν το μηχανισμό οι ενδιαφερόμενοι και δεν θα καταθέσουν ε, αιτιάσεις. Και εδώ είναι πολλές οι μεταβλητές που λαμβάνονται υπόψη. Δεν θα σταθώ λεπτομεριακά σε αυτές γιατί ο χρόνος πιέζει. Πάντως, σε τελική ανάλυση ο μηχανισμός ουσιαστικά εξαρτάται από ε, τις καταγγελίες των επιχειρήσεων. Όταν η διαδικασία της καταγγελίας είναι δαπανηρή χρονοβόρα, φυσικά δεν θα μπουν στον κόπο επιχειρήσει να κάνουν τις καταγγελίες. Οπότε ε, το κατά πόσο είναι σκόπιμο να μπει κανείς στη διαδικασία ε, θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα ανταποκρίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις καταγγελίες. Καταρχήν έχει αποτελεσματικά μέσα στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και υπάρχει εμπορική συμφωνία με τη συγκεκριμένη χώρα, γιατί όταν έχουμε εμπορική συμφωνία έχουμε και πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα επιρροή για να αρθεί ο συγκεκριμένος φραγμός. Γιατί αν ο φραγμός παραβιάζει το γράμμα είτε το πνεύμα της εμπορικής συμφωνία. υπάρχουν πολλά μέσα πολιτικής που μας επιτρέπουν να ασκήσουμε πίεση για να αρθεί ο φραγμός. Πάντως πολλές εταιρείε μας είπαν ότι σε τελική ανάλυση αυτά τα θέματα είναι θέματα εξωτερικής πολιτικής. Έχει, είναι έντονη η πολιτική διάσταση, ίσως αξίζει να μπούμε στον κόπο να κάνουμε την καταγγελία ή την αιτίαση. Οπότε αυτό, αυτό που θα επηρεάσει το κατά πόσο αξίζει να μπει στον κόπο ε, της καταγγελίας η επιχείρηση είναι αν υπάρχει κάτι παράνομο, αν παραβιάζεται είτε η εμπορική συμφωνία είτε οι κανόνες του ΠΟΕ. Αν υπάρχει παρανομία τότε έχει νόημα κανείς να κάνει την καταγγελία γιατί έχει την ευκαιρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσει πιο αποτελεσματικά. Τώρα, ο τελικός παράγοντα είναι ο, πραγματικό το πραγματικό ποσοστό επιστροφής, ε, η απόδοση. Τι συντονισμός υπάρχει με τις Βρυξέλλες μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών ή τι συντονισμός υπάρχει ε, μεταξύ των γραφείων και του ιδιωτικού κλάδου. Αυτό θα κρίνει κατά πόσο θα μπει μια επιχείρηση στη διαδικασία της καταγγελίας. Οπότε προσπαθήσαμε με την έρευνα αυτή να δούμε ποιε είναι οι προκλήσει τη εφαρμογή στρατηγικής πρόσβαση στην αγορά. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλοί υπέρμαχοι τη διαδικασία που επαναλαμβάνουν από τη βάση προ την κορυφή. Λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίε των επιχειρήσεων. Υπάρχει μια αίσθηση ότι θα μπορούσαν να ενημερώνονται καλύτερα οι εταιρείε ε, για το τι, για τι θέματα μπορούν να να γύρουν αγωγές, γιατί δεν έχουν όλες νομικούς συμβούλους και δεν ξέρουν όλες αν ο συγκεκριμένος φραγμός στοιχειοθετεί έγερση αγωγής και θα έχει πιθανότητα να τελεσφορήσει μια τέτοια αγωγή. Πάντως από την έρευνα και τις συντεύξεις ε, μας προέκυψε ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την ενημέρωση προς τις επιχειρήσεις γιατί όπως είπα πολλές επιχειρήσεις δεν γνώριζαν καν την ύπαρξη αυτού του μηχανισμού. Και πολλές επιχειρήσεις είπαν ότι μπορείτε κάπως να βελτιώσετε την ε, επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων και την ενημέρωση για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτοί οι φραγμοί στην πρόσβαση. Πάντως ε, χρειάζεται σίγουρα αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων της διαδικασίας. Αν και μερικοί είπαν ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη μόχλευση και άλλων μέσων, όπως είναι η αναπτυξιακή αρρωγή. Ε, τώρα, στις συστάσεις. Αυτό δεν είναι κάτι δικό μας, αλλά ε, συστάσεις που λάβαμε για το πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτή η στρατηγική για την πρόσβαση φαίνεται ότι υπάρχει μία διαφορά μεταξύ των εκθέσεων του ΠΟΕ, μεταξύ των εκθέσεων παρακολούθησης του τι συμβαίνει στην εμπορική πολιτική σήμερα και το τι βλέπουμε στη βάση δεδομένων για την πρόσβαση στην αγορά. Και μερικά πράγματα που δεν υπάρχουν στη βάση δεδομένων πολύ πιθανό να μην αντιμετωπίζονται. Είναι μια εμπειρική αυτή η ερώτηση και δεν ξέρουμε τι διαστάσεις έχει κάτι τέτοιο, αλλά ας το λάβουμε και αυτό υπόψη. Μερικοί πιστεύουν ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ποσοτικοποιημένους δείκτες για να δούμε τι πρόοδος έχει συντελεστεί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη χρήση εμπορικών συμφωνιών. Μερικοί ζητούν πιο διεξοδική ενημέρωση είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι γίνεται προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένοι φραγμοί στη βάση δεδομένων και γιατί μετά από μία πενταετία και ε, μετά από ακόμη περισσότερα χρόνια εξακολουθούν να παραμένουν ενισχύ οι φραγμοί. Αλλά αυτή είναι περισσότερο μια διάσταση διαφάνειας. Και τέλος, ε, κάτι που ρωτήσαμε ρητά τους συνομιλητές μας ε, είναι το τι θα μπορούσε να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια μιας διαβριμένης εταιρική σχέση, ώστε να γίνει μια τέτοια εταιρική σχέση πιο αποτελεσματική σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά. Ε, πολλά σχόλια ε, είπαν ότι θα μπορούσαν να γίνουν πολλά για να υπάρξει μόχλευση σε περιφερειακό, εθνικό επίπεδο μέσω των εθνικών βουλών στις αλληλεπιδράσεις με τις εκλογικές περιφέρειες, ώστε να γνωστοποιηθεί αυτή η διαδικασία, αυτός ο μηχανισμός. Ε, αυτόν, αυτή τη μέθοδο επισήμαναν πολύ για να ε, υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και γνωστοποίηση αυτής της διαδικασίας. Επίσης, θα μπορούσαμε το θέμα της πρόσβασης ε, της αγοράς να το έχουμε συστηματικά στις συζητήσεις με τις τρίτες χώρες όταν πραγματοποιούμε αποστολές στις τρίτες χώρες, ιδιαίτερα όταν η πρόσβαση στην αγορά είναι τμήμα του διαλόγου. Αυτό ήταν ένα συχνό σχόλιο των επιχειρήσεων, γιατί θέλουν να αυξηθεί η πίεση προς τους εμπορικούς εταίρους ε, για τα θέματα πρόσβαση στην αγορά. Και τέλος, ένα θέμα που αφορά τους πόρους αν δείτε τι πόροι αφιερώνονται για την εφαρμογή της συγκεκριμένη στρατηγικής από πλευράς ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένα μικρό τμήμα του συνόλου. Και παρόλο που υπάρχουν πολλές προτάσεις για βελτίωση, σίγουρα θα απαιτηθούν πολύ περισσότεροι πόροι, δηλαδή το θέμα εσωτερικής ανακατανομής ε, των πόρων και το προσωπικό. Αυτό θα το κανονίσει βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως, αν θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση των φραγμών πρόσβαση στην αγορά που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων, τότε θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και άρα θα χρειαστούν και περισσότεροι πόροι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. <clears throat> Ερωτήσει. Σχόλια. Χέλμουτ, εν συντομία. Μία ερώτηση που αφορά τη Συμφωνία Διευκόλυνση του Εμπορίου του ΠΟΕ, γιατί είπε ότι στον ΠΟΕ υπάρχουν δύσκολα θέματα. Αυτό το εργαλείο βοηθάει κάποιους συμμετέχοντες στο διεθνές εμπόριο ή και τις ε, επιχειρήσεις ή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να το χρησιμοποιήσουν. Έχει δηλαδή κάτι προσφέρει αυτό το παραπάνω ας πούμε στην αρχιτεκτονική Ευχαριστώ, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πολύ εύθετος ο χρόνος για αυτή τη συζήτηση και επειδή είναι εύθετος ο χρόνος γιατί τα θέματα πρόσβαση στην αγορά έχουν άμεση σχέση με την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όλο και πιο σημαντικά θα γίνονται στο θεματολόγιο της Ένωσης και τώρα και στο μέλλον. Για δύο λόγους. Όπως είπε και ο καθηγητής κ. Χούκμαν υπάρχει σαφής αύξηση του προστατευτισμού από τους εταίρους μας και δεύτερον πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο κόσμος άλλαξε. Δεν ζούμε πλέον σε ένα κόσμο όπου όλοι οι εμπορικοί εταίροι τηρούν τους κανόνες. Ε, γίνονται πολύ περισσότερες συναλλαγές. Δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα σε εταίρους που ε, δρούν με αυτόν τον τρόπο. Τους γνωρίζετε όλοι πολύ καλά, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Αλλά αυτό είναι σαφές ότι θα απαιτηθεί πλέον προσπάθειες από πλευράς μας για να αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια αυτά. Αυτό το οποίο κάνουμε για την πρόσβαση στην αγορά και η εταιρική σχέση πρόσβαση στην αγορά, το MAP βάζει στα, ε, στις τσέπες των ευρωπαϊκών ε, επιχειρήσεων πάνω περίπου 2,5%. 5 ε, δισεκατομμύρια ε, κάθε χρόνο, δηλαδή δεκάδες χιλιάδες θέσεων εργασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύπτει ένα τεράστιο φάσμα διαφορετικών κλάδων από τον αγροτικό τομέα, ICT, ηλεκτρονική, φαρμακευτικά προϊόντα, καλλιντικά και πολύ σημαντικό βοηθά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε αγορές. Αυτές είναι επιχειρήσεις που, έχουν που βοηθάμε περισσότερο γιατί αυτές έχουν και ανάγκη βοήθεια θα μας βρείτε σύμφωνος με πολλά από τα ζητήματα που έθεσε ο καθηγητής Χούκμαν, αλλά ε, βρίσκουμε τις ε, προτάσεις του επίσης πολύ χρήσιμες. Το γεγονός ότι προσθέσουμε τόσο πολλές νέες εξαγωγές επιχειρήσεις μας σημαίνει το σύστημα λειτουργεί. Όμως με τον αυξημένο προστατευτισμό πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω και πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω συνολικά και από κοινού συμπεριλαμβανομένων των οργάνων και είναι πρόσδεκτα κυρίως τα σχόλια που ακούστηκαν. Πώς θα λύσουμε το θέμα. Συμφωνούμε με τον κύριο Χούκμαν ότι περισσότερα πρέπει να γίνουν όσον αφορά την ευαισθητοποίηση. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε. Η Κομισιόν και οι αρχές των κρατών μελών πρέπει να εμπλακούν πολύ περισσότερο εκτός του χώρου των Βρυξελών. Και ακριβώς αυτό κάνουμε. Φέτος ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα, θα πάμε σε όλα τα κράτη-μέλη. Αρχίσαμε στην Κοπενχάγη πριν από περίπου μια εβδομάδα, μια μισή εβδομάδα, για να δημιουργήσουμε ημέρες εθνικής πρόσβασης στην αγορά. Θα πάμε σε όλες τις ενώσεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώσεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όλες τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρουν να του πούμε ότι αυτό, αυτή η πρόσβαση στην αγορά, το εργαλείο ή την πρόσβαση στην αγορά είναι στη διάθεσή τους. Και αυτό ε, είναι κάτι που θα κάνει η Κομισιόν. Τώρα, τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την άποψή μας. Θα το εκτιμούσαμε όλος ιδιαίτερος αν εσείς που είστε σε επαφή σε καθημερινή βάση με τις ε, εκλογικές περιφέρειες και τις μικρομεσαίες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας, που έχουν προβλήματα εξαγωγών, να τους βοηθήσετε να γνωρίσουν το εργαλείο. Θα, θα σας βοηθήσουμε το μήνυμα να γίνει σαφές σε όλους. Η ενισχυμένη επικοινωνία και η ευαισθητοποίηση είναι πολύ σημαντικό θέμα προφανώς, αλλά υπάρχει και άλλο σημαντικό θέμα που είναι οι καλύτερες προτεραιότητες και δεν ξέρω αν θα πρέπει να διαφωνήσω ή όχι με το συμπέρασμα του κυρίου Χούκμαν. Θεωρεί ότι θα πρέπει ίσως να διευρύνουμε ε, το, το, το πεδίο της πρόσβασης στην αγορά. Εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η διαδικασία θα παραμείνει δημοκρατική. Μπορεί να έχει πολλές και διάφορες ιδέες για το ποια είναι τα εμπόδια που πρέπει να παλεύουμε ως Κομισιόν, αλλά ας αφήσουμε τις ίδιες επιχειρήσεις να μιλήσουν, να μας πούν τι θέλουν. Τέλος, καλύτερος συντονισμός Προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας σε αυτό το χώρο. Έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια που λέγεται Ευρωπαϊκή Οικονομική Διπλωματία, δηλαδή προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε όλα τα τμήματα της, και τους επικεφαλής των τμήματων της Κομισιόν και τους επικεφαλής αντιπροσωπιών για να ενισχύσουμε ένα τον άλλον στο μέγιστο βαθμό. Και αυτό είναι σημαντικό. Ένα πράγμα όμως θα σας πω από την εμπειρία μου. Στην προηγούμενη θέση μου ήμουν επικεφαλής του τμήματος ε, της αντιπροσω... αντιπροσωπείας στην Κίνα. Ήταν πραγματικά θέμα πρόσβαση στην αγορά. Είχα τη χαρά να οργανώσω επισκέψεις φύσεως επιτρόπους από, και πολλών άλλων συναδέλφων από κλάδους του, της βιομηχανίας και του Πρόεδρου Σούλτς, παραδείγματος χάρη. Δεν θα πιστέψετε πόσο ισχυρό είναι ε, να μιλάει και να λέει τα ίδια πράγματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν μετακινείται και πηγαίνει. Υπάρχει χέρι τεράστιου σεβασμού και αξιοπιστία και ο κόσμο ακούει. Συμπεριλαμβανομένου και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά πόσο ο πρόεδρο Τσιμπίνγκ άκουσε προσεκτικά αυτά που του είπε ο πρόεδρο Σούλτ για θέματα πρόσβαση στην αγορά. Ε, και έχουν εν μέρη λυθεί κάποια εμπόδια στην Κίνα. Η πρότασή μου από την εμπειρία μου είναι πολύ απλή. Κάθε φορά που οποιοδήποτε, οποιαδήποτε την προσωπία του Κοινοβουλίου μεταβαίνει οπουδήποτε στον κόσμο να αναφέρεστε σε πρόσβαση στην αγορά. Και είμαστε στη διάθεσή μα να σα ενημερώσουμε. Δεν υπάρχουν καλύτεροι πρέσβεις από ότι εσεί, κύριε και κύριοι στην αγώνα αυτό όπου όλοι πρέπει να συντονίζουμε τι προσπάθειές μα. Αυτά είχα να πω και είμαστε στην πλήρη, πλήρως στη διάθεσή σας ε, ε, στην κοινή αυτή προσπάθεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου πηγαίνουμε στην Κίνα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Κύριε Χόκμαν, σύντομη απάντηση στην ερώτηση του συναδέλφου. Ναι, Νομίζω ότι σαφές είναι μέρος αυτού που είπατε. Δεν έχουμε δει μεγάλο, ε, σοβαρά αποτελέσματα, αλλά η συμφωνία έτσι λειτουργεί. Ο τρόπος που βλέπουμε να λειτουργεί η Συμβουλευτική Επιτροπή Πρόσβαση στην Αγορά έχει σχέση με σύνδεση με τα θέματα του ΠΟΕ, τις εμπορικές συμφωνίες, συμφωνίες για ε, θέματα υγιεινής. Δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει τη Συμφωνία διευκόλυνση του Εμπορίου να ενταχθεί σε αυτή τη διαδικασία και θεωρώ ότι θα γίνει ότι θα ενταχθεί. Και υπάρχουν, δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένα ότι το θέμα αυτό το έχει προωθήσει αυτή η συμφωνία, αλλά είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίζετε το θέμα, σαφώς. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε το θέμα 25, το θέμα 26 είναι τα διάφορα. Ε, δεν υπάρχει κανένα νομίζω. Και το 27 είναι οι επόμενες συνεδριάσεις, 21 και 22 Μαρτίου. Και τελειώσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.